Καλημέρα σας αγαπητοί συνάδελφοι. Είδαμε και χθε ότι δεν υπήρχε προσέλευση, όχι μόνο στην δική μα έμαθα επιτροπή. Υπάρχει πρόβλημα γενικώ λόγω των ε, κυρικών συνθήκων. Δεν μπορούμε όμω να καθυστερήσουμε άλλο, γιατί έχουμε αρκετά γεμάτη περίσσια διάταξη. Σας καλωσορίζω όλου λοιπόν να σας πω ότι δεν υπήρξε έτοιμα για τροποποίηση της μερικής διάταξης. Επίσης, όσοι ε, ήθιστε μεταδίδεται στο διαδίκτυο η συνεδρίασή μας και είναι ενδεικτικές οι ώρες ε, που αφιερώνουμε στο κάθε της διάταξης, οπότε παρακαλώ τους βοηθούς ιδίως να προσέχουν μήπως υπάρξουν απρόβλεπτες αλλαγές στην ομερήσια διάταξη και να μετατεθούν κάποια σημεία, οπότε να ειδοποιηθούν ε, οι βουλευτές. Θέλω να περάσω τώρα στο σημείο της μερισιάς διάταξης, που είναι η έγκριση των πρακτικών της συνεδρίασης της 26 και 27 Νοεμβρίου. Έχουν διανέμηθει τα πρακτικά. Είναι διαθέσιμο για όλους και θα θα εγκρίνουμε στο τέλος της συνεδρίασης εκτός αν υπάρξουν ενστάσεις. Σημείο 3. Ανακοινώσεις της Προέδρου. Δεν έχω κάποια ανακοίνωση μέχρι στιγμής τουλάχιστον. Και οι σημερινές αποφάσεις των συντονιστών θα σας ανακοινωθούν αύριο προς έγκριση. Σημείο 4 είναι το πρώτο ουσιαστικό σημείο της διάταξης και αφορά μια παρουσίαση, παρουσίαση μελέτη μελετη σχετικά με τι ολοκληρωμένε αστικέ μεταφορές και την πολιτική της συνοχή. Οι εμπειρογνώμονε είναι ήδη μαζί μας και προτείνουμε να γίνει σε εξή παρουσίαση. Να ακούσουμε καταρχά τον κύριο Βόλφκαν Ξάντε, τον κύριο επίσης Στέφαν Κλουκ από το Fraunhofer Institute for Systems and Innovation Research και εν συνεχεία την Μπετίνα Κάμπμαν από μια εταιρεία παροχή συμβουλών από την Ολλανδία, την Easy Delft και θα ακολουθήσει ανταλλαγή απόψεων και ερωταπαντήσεις. Σε ό,τι αφορά το χρόνο, δεν θα σας περιορίσω, ελπίζω όμως να είστε να κάνετε μια λογική χρήση του χρόνου, ίσως 10 λεπτά, για να μείνει και κάποιος χρόνος για συζήτηση μετά. Δεν ξέρω ποιος θα λέει πρώτος το λόγο. Σάντε, Κλουγκ, παρακαλώ. Σας ευχαριστούμε κυρία Χούμπνερ για την εισαγωγή σας. Να καλημερίσω και τους βουλευτές. Χαιρόμαστε πολύ που μπορούμε εδώ να σας παρουσιάσουμε τη μελέτη μας. Βέβαια περιμένουμε τις διαφάνειες. Θα μπορούσα να ξεκινήσω και χωρίς, ε, αλλά θα τις δείτε, φαντάζομαι, σιγά σιγά στο επιδιασκόπιο. Έχουμε και σε έντυπη μορφή τα σχετικά slides βέβαια. Λοιπόν, σας ξανακαλημερίζω. Θα μιλήσουμε λοιπόν για μια μελέτη σχετικά με τις ολοκληρωμένες αστικές μεταφορές και την πολιτική της συνοχής. Είναι ένα σημαντικό, όπως καταλαβαίνετε, θέμα, διότι γίνεται συζήτηση για την επόμενη περίοδο χρηματοδότησης και για την πολιτική συνοχή. Επίσης υπάρχει λευκή βίβλος ε, για την ε, πολιτική μεταφορών που δημοσιεύτηκε το 2011, νέος όρος μεταφορών συγκεκριμένα λέγεται και εκεί εισάγονται νέες προτεραιότητες για την πολιτική μεταφορών. Άρα είναι δύο τομείς ε, σχετικοί που θα πραγματευτούμε και στη δική μας παρουσίαση στη μελέτη. Και στην ε, μελέτη αυτή είχαμε εκτός από την EC Delft και μια άλλη βρετανική εταιρεία DGR. Still waiting for the slides. Δεν βλέπω να προβάλλει διαφάνειες, τέλος πάντων. Α, έχετε την έντυπη μορφή. Ωραία. Presenting you the agenda, which Θα σας παρουσιάσω τώρα το δεύτερο slide που είναι ουσιαστικά μια διάταξη. Το, μάλλον τα περιεχόμενα. Πρώτα είναι μια εισαγωγή, το ιστορικό, κάποια στήματα πολιτικής κτλ. Το δεύτερο κομμάτι είναι κάποιες μελέτες περιπτώσεων, τις οποίες αναλάβαμε στο πλαίσιο της μελέτης μας. Και το τρίτο τμήμα είναι τα συμπεράσματα και οι συστάσεις μας. Τρία τμήματα λοιπόν. Θα ξεκινήσω εγώ με την εισαγωγή και θα πάρω τη σκητάλη συνάδελφή μου και θα ολοκληρώσω ο Κλουκ με τις συστάσεις και τα συμπεράσματα. Λοιπόν, Όλο κάτι δεν λειτουργεί. Τώρα βλέπουμε μέσα στην οθόνη, αλλά το pointer δεν λειτουργεί. Λοιπόν, εισαγωγή της μελέτης. Δύο ήταν σημαντικοί στόχοι της μελέτης. Πρώτος, να δοθεί μια ξεκάθαρη εικόνα των μέσων σχεδιασμού αστικών μεταφορών και κυρίως τα SAMP, Sustainable Urban Mobility Plans και τα SUTP, Sustainable Urban Transport Plans. Δεν ορίζονται ακόμη ξεκάθαρα αυτοί οι δύο όροι. Ουσιαστικά το ίδιο σημαίνουν βιώσιμα σχέδια αστικής κινητικότητας ή αστικών μεταφορών. SUTP πάντως θα τα παρουσία, θα τα αναφέρω από εδώ και πέρα. Λοιπόν, για να καταλάβουμε μερικά πράγματα. Θα σας πω ποιος ήταν ε, ο βασικός μας στόχος. Ήταν τα ΣΑΜΠΙ και την πολιτική συνοχή να τα συνδέσουμε. Δηλαδή να συνδέσουμε το σχεδιασμό και τη χρηματοδότηση και τα σχετικά εργαλεία. Στην επόμενη διαφάνεια βλέπετε το ιστορικό, το υπόβαθρο της χρηματοδότησης των μεταφορών στο πλαίσιο της τρέχουσας πολιτικής συνοχής, δηλαδή στη δέκα περίοδου 2007-2013. Ε, αντιλαμβάνεστε ότι ο προπολογισμό ε, είναι 347 δις, το βλέπετε στη διαφάνεια, και το 1 τέταρτο περίπου, λίγο παραπάνω του 1 τετάρτου, του προπολογισμού αυτού είχε ε, διατεθεί για τη χρηματοδότηση έργων στον τομέα των μεταφορών. Εδώ εξετάζουμε ένα κομμάτι μόνο της πολιτικής μεταφορών και των έργων στον τομέα των μεταφορών, το αστικό σκέλος δηλαδή, το σχέλος των αστικών μεταφορών, όπου εδώ βλέπουμε να έχει τεθεί μόνο το 2,3% του συνολικού υπερπολισμού των 347 δις. Άρα μιλάμε για ένα ποσό της τάξης των 8,1 δις ευρώ. Μέχρι το 2011 μιλάμε. Δηλαδή μπορεί να έχουν προσθεθεί τα δύο τελευταία χρόνια και κάποια ακόμη δις. Το 70% του πληθυσμού της Ένωσης ζει σε αστικές περιοχές. Οι αστικές μεταφορές, επομένως, είναι ένας πολύ σημαντικός παράγοντας που διαμορφώνει και τη βιώσιμη ανάπτυξη των πόλεων. Εξού και πιστεύουμε ότι οι πόροι που διατίθενται είναι περιορισμένοι. Δηλαδή γύρω στο 2% σε αστικά ε, σχέδια μεταφορών. Στην επόμενη διαφάνεια πάντα σε σχέση με το υπόβαθρο το ιστορικό της χρηματοδότησης της πολιτικής μεταφορών. Βλέπουμε εδώ κάπως ε, αναλυτικά τα χρηματοδοτικά μέσα. Τα αστικά σχέδια βέβαια μπορούν να, να χρηματοδοτηθούν είτε από το Ταμείο Συνοχής είτε από το ΕΤΠΑ ή και από τα δύο μαζί. και για την ανάπτυξη βιώσιμων πολιτικών αστικών μεταφορών Δημιουργήθηκαν πρόσφατα επιχειρησιακά προγράμματα, τα οποία χρηματοδοτούνται από το ΕΠΑ για δίκτυα μάθηση ή ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών αστικών πολιτικών. Το Airbact 2, Interreg, EVG, ESPON είναι τρία από αυτά. Επίση, έχουμε και δύο μέσα μια στήριξη, το Jaspers και το Γέσικα, για την ανάπτυξη και το σχεδιασμό των έργων. Το Τζάσπερς και το Τζέσικα για την παροχή χρηματοδότησης για επενδύσεις ε, με απόδοση κατά κάποιο τρόπο. Λοιπόν, ωραία τώρα λύθηκαν τα τεχνικά προβλήματα με τις διαφάνειες. Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο, πάντως σε σχέση με το υπόβαθρο, είναι η πολιτική μεταφορών. που θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη και από την πολιτική συνοχή. Υπάρχουν δύο έγγραφα, το 2007 και το 2009, η πράσινη βίβλος ε, και το σχέδιο δράσης για την αστική κινητικότητα αντίστοιχα, τα οποία αναγνωρίζουν ότι οι πόλεις χρειάζονται υποστήριξη για να ε, προωθήσουν την βιώσιμη κινητικότητα στα αστικά κέντρα. Και όπως σας είπα και πριν, το 2011 δημοσιεύθηκε το, η Λευκή Βίβλος για μια ενιαία ευρωπαϊκή περιοχή μεταφορών που ζητά 60% μείωση των ε, εκπομπών άνθρακα από τον τομέα των μεταφορών μέχρι το 2050. το 40% του διοξιδίου του άνθρακα εκπέμπεται στις πόλεις από τις μεταφορές. Άρα και αστικές μεταφορές μπορούν να συνεισφέρουν σημαντικά στη μείωση του διοξιδίου του άνθρακα, που συνολικά θέλουμε, επαναλαμβάνω, η μείωση αυτή να είναι της τάξης του 60% μέχρι το 2050. Και τα τρία έγγραφα τα οποία σας προανέφερα προτείνουν ε, την ανάπτυξη ΣΑΜΠ, δηλαδή βιώσιμων ε, σχεδίων αστική κινητικότητα και επίσης αναφέρουν την σύνδεση μεταξύ πολιτική συνοχής και ΣΑΜΠ. Και θα μπορούσε ενδεχομένω να υπάρξει και ένα σχέδιο στήριξη τη Ευρωπαϊκή Ένωση για την προοδευτική εφαρμογή ε, σχεδίων αστική κινητικότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επόμενο σημείο ορισμός των ΣΑΜΠ, όπως σας είπα, δεν υπάρχει ένας κοινός ορισμός ακόμη για το TST ΣΑΜΠ. Υπάρχουν βέβαια έγγραφα, υπάρχει τεκμηρίωση, βιβλιογραφία, που εκεί γίνεται μια απόπειρα ορισμού του όρου και ήταν και το σημείο κίνησης και για τη δική μας μελέτη είναι μια ε, μελέτη Ρούπρεχτ που λέει ότι ένα στρατηγικό σχέδιο που στόχο έχει να ικανοποιήσει τις ανάγκες κινητικότητας ατόμων και επιχειρήσεων στις πόλεις και στα περίχωρα αυτών για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Αυτός είναι ένας ορισμός. Υπάρχουν και κάποια όμως πιο αναλυτικά κριτήρια που ορίζουν ένα ΣΑΜΠ και εμείς τα χρησιμοποιούμε αργότερα στις μελέτες περιπτώσεων για να αναλύσουμε κατά πόσο ένα συγκεκριμένο σχέδιο αστική κινητικότητας πληρεί τα κριτήρια ενός ΣΑΜΠ ή δεν πληρούνται ενδεχομένω ένα ή δύο κριτήρια. Πρώτο κριτήριο. Το σχέδιο θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη το κόστος και το όφελος των μεταφορών. Θα πρέπει επίσης να εντάσσεται σε ένα μακροχρόνιο όραμα και θα πρέπει να υπάρχουν συγκεκριμένοι μετρήσιμοι στόχοι βάσει των οποίων να αξιολογείται. Φυσικά οικονομική ανάπτυξη ε, και εξισορρόπησή της με την κοινωνική δικαιοσύνη και τα θέματα περιβαλλοντικής ποιότητας. Πρέπει να υπάρχει μια εξισορρόπηση όλων αυτών θα πρέπει επίσης το σχέδιο να εφαρμόζει μια ισορροπημένη, μια ολοκληρωμένη προσέγγιση, λαμβάνοντας υπόψη όλους τους τομείς πολιτική, όχι μόνο τον τομέα των μεταφορών, αλλά και τον αστικό σχεδιασμό, για παράδειγμα. Και κάποια ζητήματα που αφορούν ε, την ενέργεια, ηλεκτροκινητικότητα, για παράδειγμα, σημαντικό τομέα πολιτική που και αυτό πρέπει να λαμβάνεται υπόψη. Επίσης εμπλέκονται διαφορετικά επίπεδα ε, αρχών, αστικές αρχές, αλλά μπορεί να υπάρχουν και αρχές περιφερειακού σχεδιασμού, που και αυτοί οι φορείς εμπλέκονται. Τέλος, σημαντικό είναι να υπάρξει μια συμμετοχική προσέγγιση, με τη συμμετοχή δηλαδή όλων των ενδιαφερομένων. Έρχομαι στην διάρθρωση των διαφόρων επιπέδων πολιτικής και το πώς αλληλεπιδρούν μεταξύ τους για τη χρηματοδότηση μιλοπάντα, αλλά και για την υλοποίηση ενός ΣΑΜΠ. Υπάρχουν τα τρία επίπεδα, Ευρωπαϊκή Ένωση, κράτη-μέλη, περιφέρειες και αστικές περιοχές, πόλεις. Αυτά είναι τα τρία επίπεδα. Και υπάρχουν και διαφορετικά χρηματοδοτικά μέσα, αλλά και έργα, σχέδια, τα οποία πρέπει να διασυνδέονται από πάνω προς τα κάτω. Πρώτον έχουμε τα χρηματοδοτικά μέσα, που θα πρέπει να τηρούν κανόνες για την εφαρμογή. Τους ορίζει τις κανόνες αυτούς στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και σε πιο στρατηγικό επίπεδο έχουμε τα επιχειρησιακά προγράμματα που ορίζουν τα κράτη-μέλη με συγκεκριμένους στόχους για κάθε επιχειρησιακό πρόγραμμα. Και έπειτα από κάτω προς τα πάνω βέβαια έχουμε τα έργα μεταφορών, και τα στρατηγικά σχέδια αστικής κινητικότητας ή ΣΑΜΠ. Βλέπετε στη διαφάνεια αυτή λοιπόν και από κάτω προς τα πάνω και από πάνω προς τα κάτω έχουμε αντίκτυπο, έχουμε επιπτώσεις και αλληλεπιδράσεις. Και βέβαια θα πρέπει και οι δύο πλευρές και τα δύο ε, σκέλη να λαμβάνονται υπόψη. Τι κριτήρια λοιπόν ε, χρησιμοποιήσαμε για να επιλέξουμε τις μελέτες που περιπτώσεων. Πήραμε κάποια στοιχεία από τη βάση δεδομένων της ΔΓ ΡΕΓΚΙΟ για να δούμε ποια επιχειρησιακά προγράμματα περιλάμβαναν σημαντική χρηματοδότηση για αστικά προγράμματα και είχαμε δύο κωδικούς που τους βλέπετε 25 και 52, δηλαδή αστικές μεταφορές και καθαρές αστικές μεταφορές. Εκεί βλέπουμε να δίδεται σημαντικός προϋπολογισμός, να, να προβλέπονται σημαντικά κονδύλια. Κάτι άλλο σημαντικό είναι η πόλη που είναι στο πρόγραμμα το επιχειρησιακό και επίσης άλλο κριτήριο ήταν να υπάρχει ισορροπία μεταξύ των τριών στόχων της πολιτικής συνοχής. Και να υπάρχει επίσης και μια γεωγραφική ισορροπία. Αυτά είναι τρία σημαντικά κριτήρια που επιλέξαμε. Και ένα άλλο κριτήριο ήταν να παρέχεται και στήριξη μέσω του Τζέσικα. Λοιπόν, μπαίνουμε τώρα στις μελέτες περιπτώσεων και οι στάντις. Οι μελέτες περιπτώσεων έγιναν ε, και με βιβλιογραφική έρευνα, μελετήσαμε δηλαδή έγγραφα πολιτικής, έγγραφα σχεδιασμού, τα οποία διατίθενται στο διαδίκτυο αλλά ήρθαμε και σε επαφή με τους φορείς, δηλαδή τις διαχειριστικές αρχές, τους διαχειριστές επιχειρησιακών προγραμμάτων, τους δικαιούχους, αλλά και τις δημοτικές αρχές. Εφαρμόσαμε την προσέγγιση σε οκτώ μελέτες. Τις βλέπετε Βαρκελόνη, Κλούνα Πόκα, Κρακοβία, Λίβερπουλ, Ρέν, Στρασβούργο, Κέλ, Ταλίν και Χάλε. Δύο έχουν να κάνουν με τους στόχους που αφορούν την συνεργασία, την ανταγωνιστικότητα, δύο για τους επιχειρησιακούς στόχους κτλ. Και τώρα θα δώσω το λόγο στην άλλη κυρία Κάμπμαν, η οποία θα σας παρουσιάσει τις πρώτες μελέτες περιπτώσεων. Παρακαλώ. Thank you very much. Σας ευχαριστώ πολύ. Ας δούμε τώρα τις διαφάνειες. Τρεις διαφάνειες ανά περίπτωση, και θα δούμε εδώ πέρα τα προγράμματα τα οποία εφαρμόστηκαν, καθώς επίσης και τα βιώσιμα σχέδια αστικής κινητικότητας, τα οποία εφαρμόστηκαν σε κάθε πόλη. Ξεκινήσουμε με την περίπτωση της Βαρκελόνης. Βλέπετε εδώ πέρα μία επισκόπηση, μία σφαιρική μελέτη των βασικών παραμέτρων. Εξετάσαμε γενικότερα την περιφέρεια της ε, Καταλωνίας. Εδώ πέρα ο αρμόδιος φορέας είναι το Υπουργείο Οικονομικών της ε, περιοχής. Βλέπετε εδώ πέρα τον προπολογισμό 679 εκατομμύρια ευρώ. Είναι ο προπολογισμό ο οποίος προβλέπεται, καθώς επίσης και τον καταμερισμό που υπάρχει εδώ πέρα για τις αστικές μεταφορές προβλέπεται ένα ποσό 46,2 εκατομμύρια ευρώ. Όσον αφορά το ΣΑΜΠ της Βαρκελόνης, το σχέδιο ονομάζεται εδώ πέρα PMU, Master Plan, βασικό σχέδιο για την αστική κινητικότητα και βασικός φορέας είναι ο Δήμος της Βαρκελόνης. Ασχοληθήκαμε εδώ πέρα με ένα συγκεκριμένο μια συγκεκριμένη περίπτωση, την χρησιμοποίηση λεωφορείων σε ένα συγκεκριμένο αυτοκινητόδρομο της περιοχής, τον C58, η περίπτωση της ε, Βαρκελόνης είναι ιδιαίτερα χαρακτηριστική γιατί τα όσα εφαρμόζονται στην περιοχή αυτή επηρεάζουν γενικότερα και την αστική περιοχή της Βαρκελόνης αλλά και τη γύρω περιοχή. Βλέπετε εδώ πέρα τον αυτοκινητόδρομο εδώ. Υπάρχουν δύο ζώνες στο στερικό τμήμα του αυτοκινητοδρόμου δύο λωρίδες οι οποίες προβλέπονται μόνο για τα λεωφορεία. Κατά αυτόν τον τρόπο μειώνεται η κυκλοφοριακή συμφόρηση και αυξάνεται τελικά η κινητικότητα καθώς επίσης και η προσβασιμότητα στην πόλη της Βαρκελόνης. Ποια είναι τα βασικά συμπεράσματα από την περίπτωση της Βαρκελόνης. Καταρχάς, τα βιώσιμα σχέδια αστική κινητικότητα για τη Βαρκελόνη ανταποκρίνονται σε όλα τα κριτήρια του ΣΑΜΠ, επομένω τα πράγματα εδώ εξελίσσονται πολύ καλά. Είδαμε ότι το λειτουργικό πρόγραμμα καθώ επίση και το PMU έχουν συγκρίσιμου στόχου. Η μεταξύ του όμω διασύνδεση ήταν αρκετά περιορισμένη. Ουσιαστικά όμω ε, αντιστοιχούν και τα δύο σχέδια στου βασικού στόχου. Άρχισε να Εφαρμόστε το σχέδιο αστικής κινητικότητας αφού έχει αρχίσει να εφαρμόζεται το OP. Και βλέπουμε επίσης ότι συμμετέχει ο Δήμος της Βαρκελόνης στο βασικό πρόγραμμα PMU. Είδαμε επίσης ότι υπήρχαν ε, κάποιες διαφορές ανάμεσα στον OP Manager και την, το Δήμο της Βαρκελόνης. Ο διαχειριστής του λειτουργικού προγράμματος ασχολείται με τη γενικότερη περιφέρεια, ενώ ο Δήμος της ε, Βαρκελόνης έχει ασχοληθεί περισσότερο με την ίδια την αστική περιοχή. Και οι δύο φορείς ασχολούνται με την ε, λειτουργία του προγράμματος αυτού, καθώς επίσης και τις ε, επιπτώσεις που έχει το πρόγραμμα στην αστική περιοχή και τη γύρω περιοχή. Η επόμενη μελέτη έχει να κάνει με την Ρουμανία, με το Κλουίν Ναπόκα. Εδώ πέρα το επιχειρησιακό πρόγραμμα ονομάζεται Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξη. Είναι πολύ σημαντικό πρόγραμμα με ένα συνολικό προπολογισμό πάνω από τα 3,5 εκατομμύρια ευρώ. Και το τμήμα το χρηματοδοτικό το οποίο αντιστοιχεί στι αστικέ μεταφορέ είναι 111,8 εκατομμύρια ευρώ. Η πόλη του Κλουναπόκα έχει ένα σχέδιο στρατηγικής ανάπτυξης. Επεξεργάζεται ένα ΣΑΜΠ, αλλά αυτή τη στιγμή πρόκειται μόνο για ένα πρόγραμμα στρατηγικής ανάπτυξης, που έχει όμως και μια συνιστόσα που έχει να κάνει με τις μεταφορές. Ασχοληθήκαμε με δύο διαφορετικά σχέδια αστικής μεταφοράς. Ένα πρώτο δίκτυο για, την, για τα ποδήλατα και κυρίως για την, τη δυνατότητα των ποδηλάτων να σταθμεύσουν συγκεκριμένα σημεία της πόλης με ένα προπολογισμό 3,1 εκατομμύρια ευρώ και είδαμε επίσης και ένα δεύτερο πρόγραμμα που έχει να κάνει με τον εξυγχρονισμό του δικτύου τραμ στην πόλη. Το πρώτο σχέδιο που έχει να κάνει με τους ποδηλατόδρομους και τα ποδήλατα έχει να κάνει με την ανάπτυξη ενός δικτύου ποδηλατοδρόμων όπου να μπορούν να κυκλοφορούν έως το δυνατόν περισσότερα ποδήλατα, να προωθεί τη χρήση των ποδηλάτων και να υπάρχει και μία εκστρατεία προώθησης της χρήσης τους. Και γίνεται επίσης παράλληλα και το δεύτερο σχέδιο που σας είπα, το οποίο έχει να κάνει με τον εξυγχρονισμό του δικτύου τραμ. Και εδώ πέρα γίνονται πολλές επενδύσεις. Και τα δύο αυτά σχέδια πάντως συμβάλλουν τόσο στο στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης και ουσιαστικά συμβάλλουν και στο ΣΑΜΠ, το βιώσιμο σχέδιο στική κινητικότητας, το οποίο βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη. Ας δούμε εδώ πέρα τα βασικά συμπεράσματα. Πρέπει να ολοκληρωθεί το ΣΑΜΠΑ τον Ιούλιο του 2013. Υπάρχει χρηματοδοτική υποστήριξη από το Τζάσπερς. Μέχρι να αρχίσει να ισχύει όμως το ΣΑΜΠΑ θα λειτουργεί το σχέδιο στρατηγικής ανάπτυξης. Το σχέδιο στρατηγικής ανάπτυξης λαμβάνει υπόψη του την ανάλυση του επιχειρησιακού προγράμματος SWOT για τη βόρειο-δυτική περιοχή και έχει προσαρμοστεί ουσιαστικά το πρόγραμμα αυτό στις αστικές συνθήκες που ισχύουν στην Κλούγινα Πόκα. Το προσωπικό του Δήμου, καθώς επίσης και οι συντονιστές από τη βόρεια-δυτική περιοχή, συνεργάζονται προκειμένου να λειτουργήσει σωστά το επιχειρησιακό πρόγραμμα. Υπάρχει λοιπόν μια καλή συνεργασία. Η διευθύνουσα όμω αρχή μα είπε ότι θα ήθελε να συνεργαστεί πιο στενά με τι τοπικέ αρχέ, με την τοπική αυτοδιοίκηση, ιδίω όσον αφορά το τμήμα των δημοσίων συμβάσεων. Α περάσουμε τώρα στην Πολωνία. Κρακοβία. Εδώ πέρα εξετάσαμε κάποια αστικά προγράμματα για τις υποδομές και το περιβάλλον. Έχουμε εδώ πέρα και ένα περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα με συγχρηματοδότηση από την Πολωνία και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αρμόδιος φορέας για αυτό το OP είναι το Εθνικό Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και βλέπετε εδώ πέρα τα κονδύλια τα οποία έχουν εγκριθεί η συμβολή από τις αστικές μεταφορές είναι αρκετά περιορισμένη σε σχέση με το συνολικό προπολογισμό. Ωστόσο, γίνεται μια πολύ σημαντική εργασία προς τις υποδομές προκειμένου να αυξηθεί η διασύνδεση ανάμεσα στις διάφορες περιοχές, στις διάφορες περιοχές της Πολωνίας. Μολονότι ε, το μερίδιο των αστικών μεταφορών είναι μικρό, ο συνολικό προπολογισμό είναι πάρα πολύ σημαντικό, με αποτέλεσμα να χρηματοδοτούνται πολλά προγράμματα στα πλαίσια του ΟΠΗ. Η πόλη τη Καρκοβία βρίσκεται στην Νότιο Πολωνία. Έχει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανάπτυξη των δημοσίων ε, μέσων μεταφορά. Και εμεί εξετάσαμε δύο διαφορετικά προγράμματα αστική ανάπτυξη. Το πρώτο έχει να κάνει με την ανάπτυξη ενό ε, αστικού συστήματος διαχείρισης των μεταφορών με ένα συνολικό προπολογισμό 11 εκατομμυρίων ευρώ και εξετάσαμε και ένα ακόμα πρόγραμμα που έχει να κάνει με την κατασκευή μιας νέας γραμμής τραμ και τη δημιουργία ενός κόμβου για τα τραμ με ένα προπολογισμό 4,7 εκατομμύρια ευρώ. Όσον αφορά το σύστημα ανάπτυξης αστικών μεταφορών και διαχείρισης των αστικών μεταφορών, έχει διαμορφωθεί κατά τέτοιον τρόπο ώστε να επιφέρει πολλές βελτιώσεις αστικές μεταφορές, ιδίως στις δημόσιες μεταφορές, όπου πρέπει να βελτιωθεί τόσο το λογισμικό το οποίο χρησιμοποιείται όσο και το hardware. Και πρέπει να βελτιωθούν ε, βέβαια και κάποιες υποδομές όπως οι φωτεινοί σηματοδότες. Και να υπάρχει ένας καλύτερος έλεγχος της πρόσβασης στους, ε, ε, στις ζώνες εκείνες της πόλης με, τις, ε, με περιορισμένα μέσα μεταφοράς ή όπου επιτρέπεται να μπουν μόνο συγκεκριμένα αυτοκίνητα μέσα μεταφοράς. Επίσης, ένα άλλο σχέδιο έχει να κάνει με την γενικότερη ανάπτυξη των μεταφορών και της υποδομής, με τη δημιουργία ποδηλατοδρόμων, με την επέκταση των πεζοδρομίων και το καθεξής. Ποια είναι τα βασικά συμπεράσματα από τη μελέτη αυτή. Βλέπουμε στην περίπτωση Κρακοβίας ότι το ΣΑΜΠΑ εξελίσσεται, βελτιώνεται, αλλά δεν έχει ακόμα εφαρμοστεί πλήρως. Ανταποκρίνεται σε πολλά από τα αρχικά κριτήρια του ΣΑΜΠΑ, αλλά όχι σε όλα. Για παράδειγμα, είναι περιορισμένη η συμμετοχή των ενδιαφερομένων μερών και δεν έχει ολοκληρωθεί η μελέτη Επίσης θα πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη διασύνδεση ανάμεσα στο λειτουργικό σχέδιο της Πολωνίας και το σχέδιο αυτό το οποίο ισχύει για την περίπτωση της Κρακοβίας. Υπάρχει μια επικοινωνία και ένα τονισμός ανάμεσα στους αρμοδίους για το ΣΑΜΠ και τους αρμοδίους για το ΟΟΠ. Φαντάζομαι ότι η συνεργασία στην περίπτωση της Κρακοβίας είναι πιο εύκολη από ό,τι στην περίπτωση της Βαρκελόνης, για παράδειγμα ακριβώς επειδή όλη η κλίμακα εφαρμογής των σχεδίων γίνεται σε αστικό επίπεδο, σε επίπεδο πόλης, ενώ σε άλλες περιπτώσεις, όπως στη Βαρκελόνη, είδαμε ότι το σχέδιο αστικών μεταφορών είχε να κάνει και με ένα πιο περιφερειακό σχέδιο επενδύσεων. Το ΣΑΜΠ επίση αναθεωρείται σε τακτικά χρονικά διαστήματα προκειμένου να ληφθούν υπόψη και νέα σχέδια, νέα έργα στα πλαίσια του επιχειρησιακού προγράμματος του ΟΠΗ. Υπάρχουν βέβαια και κάποιες ε, εξαιρέσεις, αλλά εν γέννη μπορούμε να πούμε ότι οι προσπάθειες που καταβάλλονται είναι πολύ θετικέ. Ας περάσουμε τώρα στο Λίβερπουλ, στη βορειοδυτική Αγγλία. Το επιχειρησιακό πρόγραμμα για το Λίβερπουλ ονομάζεται North West England, βορειοδυτική Αγγλία. Αρμόδιος φορέας ε, είναι το Υπουργείο της ε, τοπικής η χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι περίπου 750 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η συνιστότητα που έχει να κάνει με τις αστικές μεταφορές είναι 36 εκατομμύρια ευρώ. Το Λίβερπουλ έχει ένα ΣΑΜ που ονομάζεται Local Transport Plan, τοπικό σχέδιο, τοπικό σχέδιο μεταφορών και η τοπική αρχή μεταφορών είναι η αρμόδια αρχή. Εξετάσαμε εδώ πέρα δύο σχέδια. Ένα σχέδιο που ονομάζεται Knowledge Quarter Public Real Mount Pleasant, αρμόδιο αρμόδιος είναι Δήμος του Λίβερπουλ για το σχέδιο αυτό, καθώς επίσης και ένα άλλο σχέδιο που είχε να κάνει με τις πράσινε πράσινες μεταφορές, οικολογικές μεταφορές. Και στις δύο περιπτώσεις η πόλη του Λίβερπουλ είναι η αρμόδια αρχή. Το πρώτο σχέδιο, Knowledge Quarter Public Real Mount Pleasant, ουσιαστικά αναφέρεται σε πάρα πολλές επενδύσεις που γίνονται προκειμένου να βελτιωθούν οι υποδομές όπως τα, πεζοδρόμια, οι ποδηλατόδρομοι, οι χώροι στάθμευσης των ποδηλάτων, ενώ τα σχέδια για τις οικολογικές μεταφορές είναι κάπως διαφορετικά, ουσιαστικά έχουν να κάνουν με επενδύσεις σε υποδομές μεν, αλλά στα σχέδια αυτά υποστηρίζονται περισσότερο κάποιες τουριστικές περιοχές ή κάποιοι χώροι αναψυχής. 15 διαφορετικοί οργανισμοί συμμετέχουν στο σχέδιο αυτό και μέσω του σχεδίου αυτού υποστηρίχθηκαν προκειμένου να καταφέρουν να δημιουργήσουν μεταξύ τους ένα δίκτυο επικοινωνίας. Για παράδειγμα βλέπετε εδώ πέρα μία πινακίδα που εξηγεί πώς μπορεί να πάει κανείς στο Εθνικό Κέντρο άγριας χλωρίδας. Και τα δύο αυτά σχέδια συνέβαλαν πολύ σημαντικά στο ΣΑΜΠ και έλαβαν χρηματοδότηση από την αρμόδια αρχή. Ποια είναι τα βασικά συμπεράσματα από τη μελέτη αυτή για την πόλη του Λίβερμπουλ. Βλέπουμε ότι το τοπικό σχέδιο μεταφορών ικανοποιεί όλα τα κριτήρια του ΣΑΜΠ. Ουσιαστικά απαιτείται να υπάρχει ένα ΣΑΜΠ από τον Βρετανικό νόμο. Επομένω έχουν συσσωρεύσει μια πολύ θετική εμπειρία. Το επεξεργακό σχέδιο καθώς επίσης και το σχέδιο τοπικών μεταφορών έχουν ευθυγραμμισμένους στόχους. Ουσιαστικά το προσωπικό το οποίο συμμετέχει στο ένα σχέδιο συμμετέχει και στο δεύτερο, επομένως υπάρχει μια πολύ καλή συνεργασία μεταξύ τους. Το προσωπικό γνωρίζετε πολύ καλά και συνεργάζονται πολύ θετικά, πολύ επικοδομητικά. Εκφράστηκαν βέβαια κάποιες ε, ανησυχίες για την ε, γραφειοκρατία που εμπεριέχεται στα σχέδια αυτά, καθώς επίσης και τις απαιτήσει τις διοικητικές τις οποίες πρέπει να ικανοποιήσουν. Περνάμε τώρα στη Γαλλία, ένα πρόγραμμα στην ΡΕΝ. Η ΡΕΝ είναι μια πόλη της ε, Βρετάνης, έτσι ονομάζεται και το επιχειρησιακό σχέδιο, το OP, Brittany αρμόδιος φορέας για αυτό το επιχειρησιακό πρόγραμμα είναι η επαρχία της ε, Βρετάνης με έναν προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης 301,7 εκατομμύρια ευρώ και μια αστική συνιστόσα 30 περίπου εκατομμύρια ευρώ, το 10% δηλαδή, του συνολικού προπολογισμού. Η ΡΕΝ έχει ήδη ένα ΣΑΜΠ, το PDU, το αστικό σχέδιο κινητικότητας. Αρμόδιος φορέας είναι η ΡΕΝ Μέτροπολ και εξετάσαμε εδώ πέρα δύο ξεχωριστά σχέδια αστικών μεταφορών. Το πρώτο είναι η διασύνδεση με τρένο υψηλής ταχύτητας για την Βρετάνη. Ο παρμόδιος φορέας εδώ πέρα είναι η περιφέρεια της Βρετάνης και ο προπολογισμό εδώ πέρα είναι πολύ σημαντικό, όπω βλέπετε 100 εκατομμύρια ευρώ από την Ευρωπαϊκή Ένωση για ένα σύνολο 260 εκατομμύριων ευρώ. Και εξετάσαμε επίση και ένα άλλο σχέδιο πιο περιορισμένο αυτή τη φορά, που έχει να κάνει με τη δημιουργία μια δεύτερη γραμμή για το μετρό. Αρμόδιε φορέ εδώ πέρα είναι η ΡΕΝ Μετροπόλ. Όσον αφορά το πρώτο σχέδιο, διασύνδεση με τρένο υψηλή ταχύτητα για την Βρετάνη, Βλέπετε εδώ πέρα ότι το σχέδιο είναι ιδιαίτερα φιλόδοξο. Έχει να κάνει με την δημιουργία 7 διαφορετικών τμήματων σιδηροδρομικής γραμμής, συνολικά 336 χιλιόμετρα. Και στόχος εδώ πέρα είναι να βελτιωθεί η διασύνδεση της ΡΕΝ και γενικότερα της Βρετάνης με το Παρίσι, με ένα τρένο υψηλής ταχύτητας διασχίζει ουσιαστικά την REN η γραμμή αυτή, και διασυνδέεται με άλλα συστήματα αστικών μεταφορών στην πόλη. Το δεύτερο σχέδιο που είχε να κάνει με τη δεύτερη γραμμή του μετρό, εδώ πέρα προβλέπεται μια επέκταση του φυστάμενου συστήματος μετρό και προβλέπεται επίσης η δημιουργία μιας δεύτερης γραμμής για το μετρό. Ποια είναι τα βασικά συμπεράσματα από την περίπτωση της REN. Το Urban Mobility Plan, το PDU αντιστοιχεί σε όλα τα κριτήρια του ΣΑΜΠ. Το PDU και το OP αναπτύχθηκαν παράλληλα την ίδια χρονική στιγμή. Η πρόταση OP λήφθηκε υπόψη στην κατάρτιση του σχεδίου ΣΑΜΠ. Είδαμε όμως ότι η ανάπτυξη αυτή ήταν μονομερής γιατί η αρμόδια αρχή για το OP δεν γνώριζε ε, ποια ήταν τα στοιχεία του προγράμματος ε, ΣΑΜΠ. Είδαμε ότι οι στόχοι ήταν ευθυγραμμισμένοι, αλλά δεν υπήρχαν αρκετές διασυνδέσεις, ότι ουσιαστικά η ανάπτυξη του προγράμματος γινόταν μονομερός, τουλάχιστον τη χρονική στιγμή που το εξετάσαμε εμείς. Και αρμόδιοι μας είπαν ότι η επικοινωνία μεταξύ των δύο φορέων περιορίζεται μόνο στα όσα να κάνουμε τη χρηματοδότηση των σχεδίων, αλλά δεν επεκτείνεται σε άλλους τομείς και θα παραδώσω τώρα να παρέμβετε εσείς. Θα παρουσιάσω τις, ε, τα τελευταία στοιχεία της μελέτης. Θα είμαστε στη, παραμείνουμε στη Γαλλία, θα πάμε στο Στρασβούργο και το λειτουργικό πρόγραμμα που εξετάστηκε ήταν ένα διαπεριφερειακό πρόγραμμα που συγχρηματοδοτήθηκε από το EIDC και την, ε, το στόχο της Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας σε σχέση με το Στρασβούργο είχαμε ένα πρόγραμμα και ένα σχέδιο κινητικότητας ε, και το αρμόδιο σώμα ήταν η ευρύτερη περιοχή του Στρασβούργου, η αστική περιφέρεια, κοινότητα περιφέρεια του Στρασβούργου. Και σε σχέση με τα προγράμματα, σχέδια μεταφορών, είδαμε και την επέκταση που θα ένωνε το ΚΕΛ στη Γερμανία με το Στρασβούργο στη Γαλλία, όσον αφορά τη γραμμή του Τραμ. Και βλέπουμε κάτω δεξιά ότι είχαμε σχετικά χαμηλό τμήμα, μόνο 2 εκατομμύρια συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο λόγος ποιος είναι, είναι ότι μόνο το πρόσθετο κόστος του διαμεθοριακού χαρακτήρα ενός προγράμματος προκαταβάλλεται κατά το ίμιση δηλαδή του κόστους για τη δημιουργία μιας νέας γέφυρας που θα περνά ε, πάνω από το Ρήνο και το σύνολο είναι 2,5 χιλιόμετρα με την έναρξη φέτος που θα φτάσουμε ως το 2015 και που θα ε, είναι ε, θα το εκμεταλλεύεται στη λειτουργία του η κοινότητα του Στρασβούργου. Αυτό που βρήκαμε από τη μελέτη είναι ότι το πρόγραμμα αστικής κινητικότητας που είχε ανανεωθεί υλοποιεί το, τα κριτήρια του ε, αστικού αυτού προγράμματος ε, αηφόρου κινητικότητας και βλέπουμε εδώ ότι οι εθνικοί κανονισμοί προσδιορίζουν ότι σε ένα περιφερειακό πρόγραμμα πρέπει να εντάσσεται ώστε να εντάσσεται στο σχεδιασμό για να μπορεί να τύχει η χρηματοδότηση Ωστόσο δεν λαμβάνεται ρητά ε, υπόψη να το λειτουργικό σχέδιο υπόψη. Υπάρχει όμως ευαισθησία, ευαισθητοποίηση λόγω των ε, ε, ανταλλαγών απόψεων και ανακοινώσεων υπάρχει ευρύτερη πείρα σε σχέση με αυτό και υπάρχουν κοινά όργανα όπως το κοινό όργανο γραμματείας όσον αφορά την Διευθύνουσα Επιτροπή που έχει αναλάβει την επαφή μεταξύ του οργάνου της, ε, του αστικού κέντρου του Στρασβούργου και των ε, ε, αρμόδιων για την εκτέλεση αυτού του σχεδίου. Διευκολύνεται δηλαδή η διεξαγωγή αυτού του προγράμματος. Η επόμενη περίπτωση που μελετήσαμε είναι στην, στο Ταλίν της Εσθονίας ανάπτυξη οικονομικού περιβάλλοντος, το ένα ανάπτυξη προ, περιβάλλοντος διαβίωσης living environment το άλλο καλύπτουν ένα ευρύτερο πλαίσιο κονδυλίων πάνω από ένα εκατομμύριο ευρώ το καθένα από αυτά και επίσης η πόλη Ταλίν έχει ολοκληρωμένα σχέδια μεταφορών που έχει συντάξει. Το ένα είναι το πρόγραμμα στρατηγικής ανάπτυξης του 2007, το άλλο είναι το πρόγραμμα μεταφορών του 2010. Έχουν αναπτυχθεί, έχουν εκπονηθεί από διαφορετικές υπηρεσίες της πόλης του Ταλίν. Το πρώτο από το τμήμα μελέτης μεταφορών της πόλης ε, του, της Ταλίν, το δεύτερο όσον αφορά ένα άλλο τμήμα Βλέπουμε εδώ σε σχέση με μια συγκεκριμένη γραμμή τραμ την υπαριθμό 4 που για να λειτουργήσει θα απαιτήσει αναβαθμισμένες υποδομές. Και τα νέα οχήματα αυτού του σειρμού τραμ και σε σχέση με την αναδιάρθρωση αυτής της γραμμής τράμου που απαιτείται να προηγηθεί χρηματοδοτούνται αυτά και σε σχέση με το πρόγραμμα για την μείωση των εκπομπών ρήπων η χρηματοδότηση αυτή για την πώληση των μη χρησιμοποιούμενων εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα και έτσι Μέσω του προγράμματος ανάπτυξης που εκπονήθηκε το 2007 δεν υπήρξε όμως αμοιβαία ε, επιρροή. Τα περισσότερα προγράμματα, σχέδια του Ταλίν χρηματοδοτήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ένα από ένα πιλωτικό πρόγραμμα σε σχέση με τις ε, ολοκληρωμένες ε, αστικές μεταφορές δεν έχουν όλα υλοποιηθεί. Εκείνο το οποίο απουσιάζει ακόμα είναι δεν εμπεριέχονται βραχυπρόθεσμοι στόχοι. Και ένα άλλο ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι ο προγραμματισμός που υπάρχει τώρα για να δημιουργηθεί ένα νέο ΣΑΜΠ δεν είναι ιδιαίτερα ικανοποιημένοι πολύ με τα υφιστάμενα δύο σχέδια που ε, υφίστανται και δεν έχουν επίσημα υιοθετηθεί από το Συμβούλιο της πόλης, ε, το Δημοτικό Συμβούλιο, διότι δεν ανταποκρίνονται με τις ε, απαιτούμενες προδιαγραφές. Η τελευταία μελέτη περίπτωση είναι η περίπτωση της πόλης Χάλε, που ισχύει αυτό που διαπιστώνεται για το σύνολο του κρατηδίου Σαξονίας Ανχάλτ. Το αρμόδιο σώμα είναι το Υπουργείο Οικονομικών του κρατηδίου Σαξονίας Ανχάλτ. Έχει αρκετά μεγάλο, έχει πολύ μεγάλο προϋπολογισμό πρικοδότησης και μόνο ένα μικρό τμήμα είναι για τις αστικές μεταφορές από πλευρά σχεδίου. Και το ΣΑΜΠ το οποίο λειτουργεί είναι <clears throat> το Transport Policy Vision που όμως θα αντικατασταθεί από ένα νέο πρόγραμμα ανάπτυξης μεταφορών το πρόγραμμα που εξετάσαμε είναι μια μεγάλη κατασκευή, οδική κατασκευή και ένα νέο τμήμα γραμμής τραμ από πλευράς του δικτύου του τραμ, συνολικού δικτύου χρηματοδοτούμενο με 7,6 εκατομμύρια ευρώ. Αυτή η μεγάλη ανοικοδόμηση, ας την πούμε έτσι, προβλέπει σύνδεση συνολικά εγκάρσια ανατολικά δυτικά προς την κατεύθυνση στην πόλη της Χάλε με ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα μέσα στο ίδιο πλαίσιο το νέο ποσό που βρίσκεται, το νέο ΣΑΜΠ που βρίσκεται υπό εξέλιξη εν μέρη υλοποιεί τις διατάξεις και προδιαγραφές και επίσης από τα όσα γνωρίζουμε αυτή τη στιγμή προσωρινά διότι δεν έχουν ολοκληρωθεί όλα. Δεν υπάρχουν όμως στο σχέδιο οι βραχυπρόθεσμοι στόχοι και δεν εμπεριέχονται αναθεωρήσεις των στοιχείων κόστους κόστους-οφέλους. Και πάλι εδώ βλέπουμε ότι με το λειτουργικό πρόγραμμα έχουμε κυρίως τον, στην στόχευση αναδημιουργίας, ανακατασκευής κάποιων δρόμων, κάποιων οδικών τμήματων και δεν εστιάζονται τόσο στο ίδιο το αστικό κέντρο. Θεωρείται αηφόρο αυτό το πρόγραμμα επειδή θα μπορέσει να ανακουφιστεί το βάρος της οδικής συχνότητας μεταφορών στο οδικό δίκτυο και σε σχέση με την ε, διαδικασία για την ε, χρηματοδότηση υπάρχουν και παράπονα για γραφειοκρατική επιβάρυνση. Δεν υπάρχουν τακτές ε, συνεδριάσεις όπως αναφέρεται σε σχέση με τη Βαρκελόνη. Αυτές είναι οι μελέτες περιπτώσεων και θα ήθελα να δώσω κάποια στοιχεία τώρα όσον αφορά τα συμπεράσματά μας επιλέξαμε αυτές τις 8 μελέτες περιπτώσεων και είδαμε πολύ διαφορετικό επίπεδο συνεργασίας μεταξύ των εμπλεκομένων και είδαμε ότι υπάρχουν τρία μαθήματα που πρέπει να συναγάγουμε εδώ ως συμπεράσματα. Το πρώτο από αυτά τα μαθήματα είναι ότι πρώτα και κύρια μια συνδυασμένη εκ των άνω προς τα κάτω αλλά ταυτόχρονα και εκ των κάτω, ε, από κάτω προς τα πάνω προσέγγιση πρέπει να συνδέεται και να συνδυάζεται και να υπάρχει ένα μέσο το οποίο θα καλύπτει ε, στρατηγικούς στόχους ε, και ευρύτερες ε, ανάγκες επιτόπου στο τοπικό επίπεδο προγράμμα σχέδια αστικής κινητικότητας για τις πόλεις πρέπει εκ των κάτω προς τα άνω να αναπτύσσονται. Με αυτόν τον τρόπο έχουμε ολοκληρωμένη προσέγγιση για τη διασφάλιση της ευρύτερης δυνατής συμμετοχής. Επιπλέον όσον αφορά την επικοινωνία μεταξύ των ε, αρχών σχεδιασμού και των ε, αρχών διαχείρισης, ο συντονισμός έχει κέρια σημασία. Ο συνδυασμός σε σχέση με τα μέσα για την ε, Ευρωπαϊκή Συνοχή, ιδιαίτερα όσον αφορά τα ταμεία, τα ευρωπαϊκά ταμεία, είναι κατεπίγουσα ανάγκη. Ωστόσο, ο στόχος των, της κινητικότητας για την αηφορία της κινητικότητας δεν έχει ακόμα επιτευχθεί οι ε, διαχειριστικές εκθέσεις ε, και οι εκθέσεις ελέγχου μπορούν να δώσουν ε, κάποια στοιχεία ως βάση. Όμως καμιά φορά θεωρούνται υπερβολικά γραφειοκρατικά. Πρέπει να δούμε τις εναλλακτικές δυνατότητες που μπορούν να προσφεθούν από τα το Διαθωτικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής. Συστάσεις λοιπόν πρώτα απ' όλα στον τομέα των κανονισμών και διατάξεων και των προσανατολισμών για να ξεπεράσουμε την απουσία, την έλλειψη πληροφόρησης πρέπει να έχουμε μια βάση δεδομένων στο διαδίκτυο που θα μπορούμε να χρησιμοποιούμε για να μπορέσουμε να τύχουμε πλήρους υποστήριξης. Η διαχειριστική αρχή θα μπορούσε να κάνει περισσότερα πράγματα ώστε να μεταφραστούν οι περίπλοκες αυτές διατάξεις σε εύληπτες διατάξεις για τους χρήστες. Συνολική επισκόπηση της πληροφόρησης πρέπει να είναι διαθέσιμη και πρέπει να θεσμοθετηθεί η διαδικασία πληροφόρησης ενημέρωσης με τη μορφή στρογγυλών τραπεζών για παράδειγμα όπως γίνεται και στο Στρασβούργο σε τακτική βάση, τακτική βάση. Θα πρέπει να υπάρξουν κατευθυντήριες γραμμές από πλευράς της Επιτροπής για παράδειγμα και για την διαχείριση ο συντονισμός μεταξύ των διαχειριστικών αρχών των OPs και των αρμοδίων αρχών για τα SAMPS πρέπει ε, να απαιτείται όπου αυτά τα τμήματα είναι, αυτά τα σχέδια είναι μέρη, θα είναι τμήματα του OP και θα πρέπει να υπάρχει ένα θεσμικό πλαίσιο συγκρίσιμο με μια, για παράδειγμα, με την γραμματεία, κοινή τεχνική γραμματεία των Ευρωπαϊκών Εδαφικών Προγραμμάτων, όπως το του Στρασβούργου, για παράδειγμα. Τελευταία μας σύσταση αφορά την χρηματοδότηση και λέμε ότι όταν λαμβάνονται αποφάσεις ε, για τη χρηματοδότηση ενός τέτοιου προγράμματος ε, για τις αστικές μεταφορές όσον αφορά ένα λειτουργικό πρόγραμμα θα πρέπει να διασφαλίζεται ότι το ΣΑΜΠ για μια τέτοια πόλη θα πρέπει να έχει ήδη θεσπιστεί. Αν δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο ε, από πλευράς ποι τα κονδύλια θα πρέπει να μπορούν να χρησιμοποιηθούν προς την ανάπτυξη ενός τέτοιου κατάλληλου ΣΑΜΠ ως όρο και προϋπόθεση, προαπαιτούμενο δηλαδή, για να μπορεί να εγκρίνεται η χρηματοδότηση αυτών των OP από αυτά τα OP. Αυτά είναι η σύνοψη ε, περιληπτικά των ε, συμπερασμάτων των μελετών μας. Ευχαριστούμε για την προσοχή σας. Ε, προσβλέπουμε σε ερωτήσεις και τα σχόλιά σας. Σας ευχαριστώ πολύ. Ήταν πάρα πολύ χρήσιμη αυτή η παρουσίαση γιατί θα μας βοηθήσει και σε αυτό που διαπραγματευόμαστε τώρα και το CSF, δηλαδή το Μέσο για το Σύνδεση της Ευρώπης και γενικότερα σε εργασίες μας. Σας ευχαριστώ πολύ λοιπόν για τα πολύ επίκαιρα τα αποτελέσματα. Ο Γιάνν Όλμπριχτ είναι ο πρώτος, θέλει το λόγο. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι η μελέτη αυτή ξεκάθαρα δείχνει τα καλά και τα κακά της πολιτικής. Βέβαια δεν ε, πρόκειται πιο πολύ για ερώτηση, μάλλον για παρατήρηση. Όταν ε, συζητούσαμε τον Επιτρόπο Μπαρό το θέμα της Πράσινης Βίβλου και του Σχεδίου Δράσης, είχαμε τότε ε, ρωτήσει τον Επιτρόπο ποια είναι η συνέχεια που δίδεται σε αυτά τα δύο έγγραφα. Τι δυνατότητα υπάρχει ε, να χρησιμοποιείται αυτό ως όρος, ως conditionality, γιατί φοβόμασταν τότε ότι θα, θα μείνουν στα λόγια όλα αυτά, θα μείνουμε στις υποδείξεις και στις συστάσεις. Και ποιε είναι αυτές οι συστάσεις. Είναι κάτι σαν κατευθύνσεις, κατευθύνσεις γραμμές. Δεν σημαίνουν δηλαδή τίποτα. Είναι ιδέες, καλές ιδέες, αλλά το θέμα είναι κάποιο να τις εφαρμόσει. Υπάρχουν πόλεις που ε, είναι επιτυχημένες ως προς τη διαχείρισή τους και πρέπει να στηρίξουμε τη δραστηριότητά του με ευρωπαϊκούς πόρου και αυτό είναι η επιτυχία. Έχουμε όμως και πόλεις με κακή διαχείριση που εν μέρη μόνο εφαρμόζουν κάποια πράγματα και το θέμα είναι τώρα Ποιο φταίει. Τα συμπεράσματα της εκθεσής σας, της μελέτης σας είναι σημαντικά για εμάς γιατί στην πράξη αυτό που παρατηρούμε είναι ότι υπάρχουν διαφορετικοί τομείς, επίπεδα, διαχειριστές Λέτε υπάρχουν διαφορετικοί διχειριστέ για τα ΣΑΜΠ και διαφορετικοί για τα επιχειρησιακά προγράμματα και διαφορετικοί για τα σχέδια τα αστικά. Ε, πρόκειται για χάος όπως καταλαβαίνετε. Η Ευρωπαϊκή Πόλη, Πόρη, είναι ένα πολύ καλό εργαλείο. Επομένω, είναι πολύ σωστό το συμπέρασμά σα. Αν έχουμε κάποια βασικά στοιχεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα πρέπει να τα χρησιμοποιήσουμε ω όρο, ω conditionality. Αν κάποιο θέλει για αστικά σχέδια πόρους θα πρέπει να υπάρχουν ε, εκ των προτέρων κάποιοι όροι. Ένα είδος SAMP δηλαδή, ένα είδος ε, βιώσιμου σχεδίου αστικής κινητικότητας. Και αν πληρεί τα κριτήρια θα μπορεί να χρησιμοποιεί τους ευρωπαϊκούς πόρους το σχέδιο αυτό. Επίσης, η διασύνδεση μεταξύ της διαχείρισης που λέγεται εκεί για τα επιχειρησιακά πρόγραμματα και τα COP. Αυτό είναι καταστροφή αν δεν υπάρχει διασύνδεση. Δηλαδή υπάρχει συνεργασία των τοπικών αρχών, μπορεί και να υπάρχει, μπορεί και να μην υπάρχει. Είναι σημαντικά τα συμπεράσματα λοιπόν και η Επιτροπή μας πρέπει να τα λάβει υπόψη. Και να πούμε ότι έχουμε αυτή την πολιτική, άρα και κριτήρια για τα ΣΑΜΠ, Ουσιαστικά δεν υποχρεώνεται η πόλη να κάνει κάτι συγκεκριμένο. Υποχρεώνεται όμως να πληρεί κάποια κριτήρια και αν δεν τα πληρεί δεν μπορεί να πάρει χρηματοδότηση ευρωπαϊκή. Μπορεί να κάνει ό,τι θέλει αλλά χωρίς ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Πρέπει να υπάρχει ευθύνη λοιπόν. Άρα αυτά τα συμπεράσματα είναι χρήσιμα και νομίζω ότι θα πρέπει να αξιοποιήσουμε τη μελέτη αυτή ως ένα από τα στοιχεία της αρεσιμότητας για την επόμενη περίοδο. Θέλω να ευχαριστήσω τους συντάκτες της μελέτης γιατί αποδεικνύουν ότι οι αμφιβολίες μας ε, ήταν ορθές πριν από μερικά χρόνια. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, πριν δώσω το λόγο στον Γιάννη Νίλσεν, θέλω να σας πω ότι από τη ΓΑΜΑ Δελταρέγγιο έχουμε τη Ζακλίνη Σουγέ Ολιβέηρα. Θέλουμε να της δώσουμε αργότερα το λόγο στη συζήτηση, αλλά ο Γιάννη Νίλσεν πρώτα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε τον λόγο. Θα είμαι θα, συντομότατα θα παρέμβω. Μπορώ να συμφωνήσω με αυτά τα οποία είπε ο κύριος Όλμπριχτ. Στα συμπεράσματα τι βλέπουμε. Λέμε ότι η τα αηφόρα σχέδια ανάπτυξης δεν έχουν επιτευχθεί όσον αφορά τους στόχους τους ε, σε όλα τα σχέδια. Διαρωτώ στο μέλλον αυτά μπορούμε να τα υποστηρίξουμε. Ποτέ δεν μπορούμε να υποστηρίξουμε ότι οι στόχοι δεν επιτυγχάνονται. Οι δεδομένοι στόχοι όσον αφορά την αηφορία. Δεν μπορούμε να δεχτούμε κάτι τέτοιο. Μπορούμε να πούμε δεν δεχόμαστε ότι αυτό μπορεί να είναι μια δικαιολογία, ότι δεν επετεύχθηκαν οι στόχοι. Πρέπει λοιπόν να είμαστε ξεκάθαροι σε αυτό και με αυτό συμφωνώ. Είναι μια καλή έκθεση που ανοίγει, προσφέρει δυνατότητες, αλλά όμως θα πρέπει να δούμε τα συμπεράσματά μας. Uh, uh, Υπάρχει κάποιο άλλο συνάδελφο που θα ήθελε να θέσει ένα ερώτημα, να κάνει ένα σχόλιο. Αλλιώ ε, θα ήθελα και εγώ να θέσω δύο σύντομα ερωτήματα. Το πρώτο. Βλέπετε κάποια διαφορά σε οποιαδήποτε θα έλεγα πτυχή μεταξύ των σχεδίων τα οποία εφαρμόστηκαν με μεγάλη συμμετοχή χρηματοδότηση από την πολιτική συνοχή. Υπήρχε η περίπτωση της Κρακοβίας, του Ταλίνα, αλλά και το Λιβερπούλ και Βαρκελόνη. Εκεί είχατε σχετικά μικρή ε, συμβολή. Είδατε κάποια διαφορά σε σχέση με το μείζονο στόχο της μελέτης σας. Και το δεύτερο, είδαμε κάποιες διαφορές μεταξύ των μελετών περιπτώσεων σε ό,τι αφορά τη σχέση μεταξύ επιχειρησιακού προγράμματος και διαχειριστών του επιχειρησιακού αυτού προγράμματος στο επίπεδο της περιφέρειας συνήθως και των ε, φορέων εφαρμογή του σχεδίου. Είπατε ότι κάποιε φορέ η αλληλεπίδραση η διασύνδεση ήταν μικρή, ήταν περιορισμένη, ενώ κάποτε είπατε ότι υπήρχε καλή συνεργασία. Γιατί λοιπόν υπάρχει αυτή η αποκλήση και πού οφείλεται. Θα ήθελα κάποια σχόλια πάνω σε αυτό. Τώρα, η Κομισιόν θέλει να μιλήσει τώρα ή αργότερα. Τώρα. Καλό θα ήταν, σωστό να πάρετε το λόγο. Καλημέρα σας και σας ευχαριστώ που μας δίνετε τη δυνατότητα να μιλήσουμε σήμερα. Πρώτα απ' όλα να πω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλωσορίζει την πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την παρουσίαση της μελέτης για τη διασύνδεση μεταξύ ολοκληρωμένων σχεδίων αστικών μεταφορών και της πολιτικής συνοχής. Θα μελετήσουμε τα συμπεράσματα της μελέτης πάρα πολύ προσεκτικά και προσβλέπουμε και σε μια ανταλλαγή απόψεων για το πολύ σημαντικό αυτό θέμα. Τα βιώσιμα σχέδια αστικής κινητικότητας, τα ΣΑΜΠ, είναι πρόσφατο, σχετικά πρόσφατος όρος. Πάντως η ίδια η έννοια δεν είναι εντελώς καινούρια. Πριν από 10 χρόνια ήδη η Κομισιόν είχε συγκροτήσει μια ομάδα εμπειρογνωμόνων για να εκπονήσει μια μελέτη για τα βιώσιμα σχέδια αστικών μεταφορών που όπως είπαν και οι συντάκτες μελέτης είναι λίγο πολύ το ίδιο με αυτό που συζητούμε σήμερα, δηλαδή τα σχέδια αστικής κινητικότητας. Η τότε μελέτη ολοκληρώθηκε το 2004, δηλαδή πολύ πριν το 2007. Μία ημερομηνία που αναφέρεται στην μελέτη που σας παρουσίασαν σήμερα. Σε ό,τι αφορά τώρα τα σχέδια αυταστικών μεταφορών, εμεί λάβαμε υπόψη μα τι προτάσει, την πρότασή μα, στρατηγική μα για το αστικό περιβάλλον το 2004. Όμω ε, τα βιώσιμα σχέδια αστικών μεταφορών δεν μπορούσαν να επιβληθούν από την Επιτροπή όταν διαπραγματευόμασταν με τα κράτη-μέλη τα τρέχοντα προγράμματα, τα τρέχοντα επιχειρησιακά προγράμματα. Όταν λέω τρέχοντα, μιλώ για το περίοδο 2007-2013. Γιατί? Διότι δεν υπήρχε ρυθμιστική βάση, νομική ρυθμιστική βάση για να το πράξουμε. Δεν μπορούμε λοιπόν να, έχουμε, να επιβάλλουμε αναδρομικές απαιτήσει για την τρέχουσα χρηματοδότηση. Αλλά αυτό μας δίδαξε κάποια πράγματα. Εξού και στηρίζουμε την ιδέα οι δαπάνες για τις αστικές μεταφορές να είναι πιο στρατηγικού χαρακτήρα το μέλλον. Δηλαδή, όταν δαπανώνται ευρωπαϊκά κονδύλια σε σχέδια αστικών μεταφορών, θα πρέπει να υπάρχει εγγύηση ότι τα σχέδια πληρούν πράγματι τι τοπικέ απαιτήσει και ευθυγραμμίζονται με τους στόχους πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κάτι που βέβαια μάλλον συμβαίνει περισσότερο στις πόλεις που έχουν αναπτύξει τοπικές στρατηγικές και έχουν και σχέδια για την βελτίωση της ε, επίτευξης των στόχων αυτών για καλύτερη βελτιωμένη αστική κινητικότητα. Με βάση λοιπόν αυτά, πρότεινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στη Λευκή Βίβλο για τις Μεταφορές που υιοθετήσαμε το Μάρτιο του 2011, Πρότεινε λοιπόν η Κομισιόν τη διασύνδεση της πρόσβασης σε χρηματοδότηση σε σχεδίων αστικών μεταφορών με την ύπαρξη ενός ΣΑΜΠ. Είναι η πρωτοβουλία παριθμών 31 της Λευκής Βίβλου. Επίσης, η Επιτροπή ανακοίνωσε ένα πακέτο αστικής κινητικότητας για το τρέχον έτος, το 2013, που μεταξύ άλλων θα αποσκοπεί στην υλοποίηση της πρωτοβουλίας που σας προανέφερα, της παριθμών 31. Γάμα Δελτα Μουβ είναι εδώ συνάδελφή μου από αυτή τη Γενική Διεύθυνση. Επεξεργάζεται το θέμα αυτό και η Γάμα στηρίζει την πιο στρατηγική, αν θέλετε, χρηματοδότηση στο μέλλον. Επίσης θα ήθελα να ολοκληρώσω λέγοντας ότι έχουμε και πολύ συγκεκριμένα σχόλια για συγκεκριμένα ε, κομμάτια της μελέτης. Θα σα τα διαβιβάσουμε ε, στη γραμματεία συγκεκριμένα της Επιτροπής σας. Αλλά θα σα δώσω ένα παράδειγμα. Υπάρχει ένα πολύ σημαντικό αριθμητικό στοιχείο για τι αστικέ μεταφορές που αναφέρθηκε. 8,1 δι ευρώ Λίγο πολύ, βέβαια πρέπει να το ελέγξουμε, να το παληθεύσουμε, αλλά συμφωνούμε. Συμφωνούμε λίγο πολύ. Δεν είναι όμως ένα ποσό παντιστική στο 2,3 του προϋπολογισμού, του συνολικού προϋπολογισμού ε, για τις μεταφορές στην τρέχουσα περίοδο προγραμματισμού, αλλά πρόκειται για 10% περίπου αυτού του ποσού, γιατί τα συνολικά ε, ποσά που έχουμε για τις μεταφορές ε, στα τρέχοντα επιχειρησιακά προγράμματα είναι 81,7 Αλλάζει βέβαια το χρόνο αυτό το ποσό γιατί τα κράτη-μέλη μπορούν να τροποποιούν τα ποσά που ε, κατανέμουν στους διάφορους τόμεις. Δεν είναι σταθερό ποσό, είναι μεταξύ των 81-82 δις. Άρα το 8,1 που αναφέρεται στη μελέτη είναι γύρω στο 10% του ποσού. Ένα παράδειγμα μόνο είναι αυτό, αλλά θα σας δώσουμε τα συγκεκριμένα αυτά σχόλια σε γραπτή μορφή και επαναλαμβάνω θα τα δώσουμε στην γραμματεία σας. Αυτά έχω να πω μέχρι στιγμή. Σας ευχαριστώ. Thank you very much. I would like also... Σας ευχαριστούμε πολύ. Γιάννα, θα ήθελα να δώσω πρώτα το λόγο στην DG Move. Δεν ξέρω αν θέλουν και αυτοί να πάρουν το λόγο ή ακούτε απλώς. Όχι, συμφωνούμε με τα όσα είπε η συνάδελφος από την DG Regio. Τα βιώσιμα σχέδια αστικής κινητικότητας και όλη η ιδέα πίσω από αυτά είναι ένα ζήτημα το οποίο μας απασχολεί εδώ και κάποιο καιρό. Η μελέτη που παρουσιάστηκε σήμερα είναι μια μελέτη την οποία πρέπει να εξετάσουμε περισσότερο, πολύ προσεκτικά. Θεωρώ πάντως ότι συμβάλλει πάρα πολύ στην όλη συζήτηση, η οποία πρέπει να λάβει χώρα και πρέπει να συνεχιστεί και στο εγγύς μέλλον καθώς θα προετοιμάζουμε την όλη δέσμη μέτρων για την κινητικότητα και πρέπει να δημιουργηθεί ένας ισχυρός σύνδεσμος ανάμεσα στα σχέδια αυτά και την απαραίτητη ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Πρέπει όμως για να γίνει κάτι τέτοιο να γνωρίζουμε ακριβώς ποιες είναι οι προϋποθέσεις που θα πρέπει να εφίστανται. Ξέρετε ότι υπάρχει μια κάποια ευελιξία αυτή τη στιγμή, πράγμα το οποίο σημαίνει Μάλλον οι άνθρωποι που κάναν τις μελέτες αυτές είχαν μια κάποια ευελιξία η οποία ενδεχομένω να μην υπάρχει στο μέλλον. Ξέρετε ότι σε ορισμένε περιπτώσει είδαμε ότι κάποια σχέδια ήταν SAMP, ανταποκρίνονται δηλαδή στα κριτήρια των βιώσιμων σχεδίων αστική κινητικότητα. Σε άλλε περιπτώσει τα σχέδια δεν ανταποκρίνονται στα κριτήρια αυτά. Αν όμω θέλουμε πραγματικά να υπάρχει μια ισχυρή διασύνδεση ανάμεσα στα σχέδια αυτά και την ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, πρέπει να υπάρχουν πολύ συγκεκριμένα κριτήρια τα οποία θα πρέπει βέβαια να τηρούνται και θα πρέπει να εκφραστούν με απόλυτη σαφήνεια. Πρόεδρος. Ναι, όντω και εμεί σα υποστηρίζουμε στη δημιουργία αυτή τη νομική ασφάλεια. Ξέρουμε και εμεί ότι μπορεί να είναι πάρα πολύ επιζήμιο το να μην υπάρχει νομική ασφάλεια και ότι μπορεί να οδηγήσει και σε πολύ μεγάλε καθυστερήσει. Γιάννη. Σα ευχαριστώ. Πιστεύω ότι πριν από το 2007 στη συζήτηση το επιχείρημα ότι αυτό είναι θέμα επικουρικότητας, τίποτα δεν μπορεί να επιβληθεί στις πόλεις. Το αποτέλεσμα είναι αυτό που βλέπουμε. Τελεία και παύλα. Με άλλα λόγια, αυτή είναι η απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ή θα παραμείνουμε πιστεί σε αυτές τις ε, προτάσεις ή θα έχουμε όρους και προϋποθέσεις και τότε θα πρέπει να υποστηρίξουμε αυτή την προσπάθεια. Δεν πρέπει να έχουν ε, ε όρους και προϋποθέσεις. Ε, κανένα, πρέπει να υπάρχουν όμως σαφείς αρχές. Κανείς δεν υποχρεώνεται να παίρνει ευρωπαϊκό ευρωπαϊκό κονδύλια. Αν όμω ε, κάποιο θέλει να έχει τέτοια κονδύλια στη διάθεσή του, τότε πρέπει να γίνεται αυτό με τι ορθές διαδικασίε. Θα σα υποστηρίξουμε σε σχέση με το θέμα αυτό για να δούμε πώ μπορεί να λειτουργήσει το θέμα αυτό. Και σε σχέση με τι προτάσει αυτέ θα χρειαστούν πολλά περισσότερα κονδύλια για την αστική κινητικότητα. Δεν μπορούμε να μεταθέσουμε χρήματα για προτεραιότητε, χωρί να υπάρχει ένα σαφέ νομικό πλαίσιο πιο πριν. Αυτή είναι νομίζω η πολύ διπλωματική απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που λέει ότι τίποτα δεν μπορεί να γίνει. Κάτι μπορεί να γίνει. Μπορεί να γίνει και πρέπει να αλλάξουν τα πράγματα τώρα. Γιατί αν δεν αλλάξουν τα πράγματα τώρα θα βλέπουμε τα πράγματα να συνεχίζονται όπως διαπιστώνονται σε αυτή τη μελέτη. Θα έχουμε διαχείριση από διαφορετικές αρχές που μπορεί να συνδέονται ή να μην συνδέονται μεταξύ τους. Αυτό είναι απόλυτα παράδεκτο. Σας ευχαριστώ, λέει η Πρόεδρος αν δεν θέλει να λάβει κανείς ε, τον λόγο από την Γενική Διεύθυνση Ρέτζη, θα ζητούσα από τους συντάκτες ε, της μελέτης να σχολιάσουν. Ή αν θέλετε σε σχέση με την πληροφόρηση να υπάρξει κάποια περαιτέρω παρέμβαση, ευπρόσδεκτη είστε. Ευχαριστώ για τις ερωτήσεις. Θα ήθελα πρώτα να απαντήσω στο σχόλιο από την Γενική Διεύθυνση Ρέγγιο για τη χρηματοδότηση. Έχουμε το 2,3% που ε, σε σχέση με τα ε, ε, σχέδια αυτά είναι περίπου το 1,4% ή και το 2,3% αναφέρεται στο συνολικό προϋπολογισμό που είχαμε. Αυτό είναι ο συσχετισμός αναλογίας για αυτό το 2,3% που είχαμε. Και κατανοώ ότι αυτό το μερίδιο είναι, ας το πω έτσι, κάπως περιορισμένο αυτό το ποσοστό. Το δεύτερο σημείο που θα ήθελα να αναφέρω είναι το εξής όχι σε ερώτημα που έγινε, αλλά να τονίσω για άλλη μια φορά την τελευταία σύσταση που διατυπώσαμε, ότι είναι σημαντικό τα ΣΑΜΠΣ να είναι επιλέξιμα για χρηματοδότηση από πλευράς ΟΠΗ. Αυτό ρητά το διατυπώνουμε. Είναι η τελευταία παύλα από πλευρά συστάσεων. Είναι σημαντικό να, να εντάσσεται αυτό μέσα στο ΟΠΗ και να μην έχουμε την, τον κίνδυνο να μην μπορούν κάποια τέτοια ε, σχέδια να χρηματοδοτηθούν επειδή δεν θα εντάσσονται στη διαδικασία επιλεξιμότητας. Ολοκλήρωσα μπορώ να δώσω τον λόγο στον συνάδελφο. Ευχαριστώ. Εγώ να απαντήσω τα ερωτήματά σας κυρία Χρύμνερ. Ρωτήσατε αν υπάρχει γενική διαφορά μεταξύ περιφερειών που έχουν ευρύτερη χρηματοδότηση και άλλων περιφερειών που έχουν μικρότερη χρηματοδότηση σε σχέση με την αηφορία και τις αστικές μεταφορές. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάποιο τέτοιο, να καταλήξουμε σε κάποιο τέτοιο γενικό ε, συμπέρασμα. Αναπερίπτωση πρέπει να βλέπουμε τα πράγματα. Για παράδειγμα, στο Ταλίν της Εστονίας που πήρε μεγάλα κονδύλια, η τα πράγματα δεν είναι τόσο αρνητικά. Υπάρχουν δύο στρατηγικά σχέδια ε, που έχουν παρουσιαστεί, δεν έχουν εγκριθεί από το ε, Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης. Δεν μπορούμε να καταλήξουμε όμως σε ένα τέτοιο ισοπεδωτικό συμπέρασμα ε, όπως διαφαίνεται από το ερώτημά σας. Το δεύτερο θέμα για τη συνεργασία πράγματι έχει κέρια σημασία η επικοινωνία ή σε θεσμικό ή ατομικό επίπεδο σε σχέση με τα σχέδια αυτά για τα αστικά κέντρα. Δηλαδή να έχουν ε, συζητηθεί όλα αυτά και να έχουν εξεταστεί σε βάθος ε, ε, αναλώνεται πολύ μεγάλη προσπάθεια και για το αν από πλευρά σοπή μπορούν αυτά να λειτουργήσουν ή όχι. Στο τέλος τέλος θα εξοικονομήσουμε κονδύλια και θα είναι πιο αποτελεσματική διαδικασία αν έχει, υπάρχει μια, έχει υπάρξει μια τέτοια εξέταση πιο πριν. Ναι, αλλά και ε, συνεπής ε, συνεκτική στρατηγική πρέπει να υιοθετείτε. Αν δεν υπάρχει αυτή, τότε κινεί το ένας προς τη μία κατεύθυνση, ο άλλος προς μία άλλη κατεύθυνση χωρίς συντονισμό. το ολοκληρωμένο πλαίσιο, η ένταξη σε ένα ενιαίο πλαίσιο όλων αυτών είναι πολύ σημαντικό από πλευρά συντονισμού. Ευχαριστώ. Δεν υπάρχουν άλλα σχόλια και δεν βλέπω κάποιος από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να θέλει να τοποθετηθεί εκ νέου. Θα έλεγα ολοκληρώσαμε αυτό το σημείο στην ημερησία διάταξη και πάλι πιστεύω ότι έχουμε πραγματικά πολύ χρήσιμα, μια πολύ χρήσιμη μελέτη πρόκληση για μας είναι να την χρησιμοποιήσουμε αυτήν στη διαπραγμάτευση, στη διαβουλεύση όχι μόνο του κανονισμού αλλά και της ε, των στρατηγικών προσανατολισμών και στόχων σε σχέση με ένα κοινό στρατηγικό πλαίσιο για αυτές τις πολιτικές από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βασιζόμαστε επίσης και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι έγκαιρα θα μπορέσουν να γίνουν όλα αυτά σε σχέση με τις απαιτήσει ε, για τους όρους και προϋποθέσεις. Η νομική βεβαιότητα και ασφάλεια θα πρέπει να είναι πραγματικότητα για τα κράτη-μέλη για να μπορέσουν τα πράγματα να λειτουργήσουν σωστά. Και έτσι θα ήθελα να ευχαριστήσω και πάλι για τους, τους ίδιους τους συντάκτες αυτής της μελέτης, Μελέτης ολοκληρώθηκε αυτό το σημείο, το επόμενο αναβάλλεται. Μπορούμε να περάσουμε στο επόμενο, αλλά ο, κύριος, ο υπεύθυνος, ο κύριος ε, Γιένς Γκάιρ δεν είναι εδώ, δεν παρίσταται. Μπορούμε να περιμένουμε μέχρι να προσέλθει αν υπάρχει κάποιος από τους συμβούλους ή βοηθούς που θα μπορούσαν να έρθουν σε επαφή με αυτόν για να διευκολυνθεί η νωρίτερη το δυνατόν άφηξη του κυρίου Γκάιερ εδώ θα ήταν χρήσιμο. Αν όχι, ε, τότε λυπούμε. Θα πρέπει να διακόψουμε τις συνεδρίες, αλλά δεν ξέρω για ποιο διάστημα θα πρέπει να την διακόψουμε, μέχρι να προσέλθει. Αν δεν προσέλθει, τότε θα δούμε πώς θα ανασχεδιάσουμε τις εργασίες μας. Τι είναι αυτά; είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι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 Αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα να περάσουμε στο επόμενο σημείο της ημερησίας διάταξης, στο σημείο 5 στην ημερησία διάταξη, που είναι ανταλλαγή απόψεων στο πλαίσιο της έκθεσης Jens Geier για τις περιφερειακές στρατηγικές για βιομηχανικές περιοχές στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ήθελα να ξεκινήσω δίνοντας τον λόγο στον κύριο Jens Geier και μετά θα έχουμε την παρουσίαση από τον κύριο Κλάους Σούλτς που είναι ο πολιτικός αναλυτής ε, από πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, στην Γενική Διεύθυνση Ρέγγιο Περιφερειών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ώστε να συζητηθεί το θέμα της ε, βιομηχανικής ανανέωσης. Ελπίζω ότι οι άλλοι θα προσέλθουν υστερότερα. Θα ήθελα να δώσω τον λόγο στην αρχή στον κύριο Γιάννη Γκάιερ. Παρακαλώ. Έχετε τον λόγο. Σας ευχαριστώ κυρία Χιμπνερ. Χαίρομαι για το γεγονός ότι σήμερα το πρωί λίγο πιο σε μεγαλύτερο βάθος μπορούμε να συζητήσουμε για αυτό το πολύ ενδιαφέρον θέμα. Για την σπουδαιότητα αυτού του θέματος ε, σύντομα μπορεί να αποδείξει κανείς τα δεδομένα ή βιομηχανική ε, βάση της Ευρώπης είναι εκείνη που ως θεμέλιο βοήθησε να ξεπεράσουμε τις καταστροφές του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Όμως είχαμε πρώτα τα κέντρα της χαλιβουργίας στην Δυτική Ευρώπη, στην Λίλ, Πάντε Καλέ, Μάντσεστερ, ε, η περιοχή γύρω από το Μάντσεστερ, γύρω από την Λιέγη ή την περιοχή του Ρούρ, που είναι η δική μου γενέθλια ευρύτερη περιοχή που είχαν προβλήματα που έπρεπε να αντιμετωπιστούν βιομηχανικής αναδιάρθρωσης ή εκεί όπου η διαδικασία αυτή ξεκίνησε με τον πιο σαφή τρόπο ανάλογα με την περιφερειακή στρατηγική που ακολουθήθηκε αυτές οι διαδικασίες προσαρμογής στέφθηκαν με διαφορετική επιτυχία εκάστοτε αλλά το κοινό του στοιχείο είναι μπορώ να πω ότι τα μέσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη βιομηχανική πολιτική διαδραμάτισαν σημαντικό ρόλο για το πώς τα χρησιμοποίησαν αυτά τα μέσα οι περιοχές, οι περιφέρειες αυτές και πώς ξεπέρασαν τα προβλήματά τους. Αντιμετωπίζουμε διτή πρόκληση σήμερα. Αφενός να διασφαλίσει τη βιομηχανική της βάση και να, να την επεκτείνει η Ευρώπη. Δεν θέλουμε να οπισθοχωρήσουμε στην παγκόσμια σκηνή. Αυτό είναι ένα από τα μαθήματα που συναγάγαμε από την κρίση στις περιοχές εκείνες όπου υπάρχουν βιομηχανικοί πυρήνες ή όπου υπάρχει βιομηχανική παράδοση και είναι δεδομένη, αυτές οι περιοχές και περιφέρειες μπορούν να διαδραματίσουν ένα ιδιαίτερο ρόλο. Όμως αυτές οι περιφέρειες χρειάζονται η δεδομένη υποστήριξη και ενίσχυση από την πλευρά της στρατηγικής που θα ακολουθηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να εμπεριέχονται στοιχεία όπως ε, ανάπτυξη νέων οικονομικών προοπτικών ε, ε, που θα βασίζεται στην ανάλυση των κεκτημένων και των επιτευγμάτων της κάθε περιφέρειας, η διασφάλιση αηφορίας επίσης που υπό το πρίσμα της ιδιαίτερης περιβαλλοντικής κατάστασης που αντιμετωπίζουν αυτές οι περιφέρειες το παλαιό τους βιομηχανικό παρελθόν δεν το έχουμε ξεπεράσει απόλυτα περιβαλλοντικά. Στη δική μου περιοχή δεν μπορεί κανείς να ξεκινήσει κανένα μεγάλο τέτοιο σχέδιο χωρίς πιο πριν να υπάρξει ένας συνδυασμός ε, αντιμετώπισης ερειπίων και βομβών που δεν έχουν εκραγεί από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο κατά το παρελθόν, το βιομηχανικό παρελθόν ε, της, ε, των ανθρακοριχείων και των χαλιβουργείων ε, κανείς δεν μπορεί να πληρώσει ή να ξεπεράσει τέτοιου είδους προβλήματα εύκολα. Αυτό είναι ένα παράδειγμα της ξεχωριστής κατάστασης που πρέπει να αντιμετωπίσουν αυτές οι περιοχές μας. Το τελευταίο στοιχείο που πρέπει να αναφέρουμε είναι τα προσόντα και οι ικανότητες και οι δεξιότητες. Πρέπει συγκεκριμένοι άνθρωποι να επιλεγούν που θα έχουν αυτά τα προσόντα αλλά και να διασφαλίσουν με το αναγκαίο εργατικό δυναμικό που θα έχει αυτά τα προσόντα και δεξιότητες για την οικονομική ανάπτυξη ως προοπτική αυτών των περιοχών και περιφερειών. Αυτά είναι προαπαιτούμενα που θέλω να ε, παρουσιάσω. Είχα συναντήσεις και συζητήσεις με επαΐοντες και ειδικού από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για παράδειγμα πιο πριν. Η σημερινή ακρόαση είναι αποκοίημα των προβληματισμών που από κοινού ε, διεξαγάγαμε όλοι μας. Εγώ έχω, έχω καταλήξει σε κάποια συμπεράσματα Ελπίζω ότι θα συνειφανθούν με τα συμπεράσματα των άλλων και έτσι θα έχουμε χρόνο για μια εμβαθυμένη συζήτηση επ' αυτών των στοιχείων. Ευχαριστώ. Uh, Σας ευχαριστώ πολύ. Δεν ξέρω αν θα θέλατε εσείς να παρέμβετε παρακαλώ στη συνέχεια. Euh, Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Έχετε απόλυτο δίκιο. Η έκθεση αυτή είναι πάρα πολύ σημαντική ιδίως στην παρούσα συγκυρία. Επί του παρόντος, και το επιθυμήσετε κι εσείς, η βιομηχανία σε ευρωπαϊκό επίπεδο παρουσιάζει μια πολύ σημαντική μείωση. Επομένως πρέπει να αλλάξουμε τρόπο λειτουργίας, πρέπει να αλλάξουμε κατεύθυνση. Χρειάζονται κάποιες αποτελεσματικές απαντήσεις που να ανταποκρίνονται σε όλες τις κρίσεις που γνωρίζουμε, την οικονομική, την κοινωνική, την οικολογική, αλλά επίσης και στην κρίση πολιτικής βούλησης. Πρέπει δηλαδή τα κράτη-μέλη να ακολουθήσουν ένα νέο προσανατολισμό όσον αφορά την ευρωπαϊκή βιομηχανική πολιτική. Ένα μέτρο ορόσημο, το οποίο πιστεύω θα πρέπει να μας κατευθύνει, είναι αυτός ο βιομηχανικός έπα, ο οποίος θα πρέπει να ακολουθεί πλέον μια οικολογική γραμμή, θα πρέπει να ευνέεται από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Πραγματικά πρέπει να ανταποκριθούμε σε μια πάρα πολύ σημαντική πρόκληση αυτή τη στιγμή. Η πρόκληση έχει να κάνει με τις ε, νέες ε, οικολογικές ε, βιομηχανικές πολιτικές οι οποίες θα πρέπει να αναπτύσσονται τοπικά. Ξέρετε ότι δεν υπάρχει απαραίτητη επαγγελματική κατάρτιση, δεν υπάρχουν τα απαραίτητα μέσα προκειμένου να καταφέρουμε να κατευθύνουμε τον τομέα της ενέργειας. Η έκθεση λοιπόν αυτή θα πρέπει να αποτελέσει ορόσημο, ένα ορόσημο σαφές, ξεκάθαρο. Θα μου πείτε όμως τι θα γίνει με τη χρηματοδότηση. Μα σαφώ και το ζήτημα της χρηματοδότησης είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πιστεύω λοιπόν ότι στα πλαίσια της έκθεσης αυτής θα πρέπει να εξετάσουμε τρόπους για να έχουμε τελικά και μια οικολογική φορολογία και να καταφέρουμε πραγματικά να χρηματοδοτήσουμε Μία πολιτική η οποία θα πλαισιώσει την ευρωπαϊκή βιομηχανία η οποία αυτή τη στιγμή πεθαίνει. Θα πρέπει να βοηθήσουμε τη βιομηχανική, την ευρωπαϊκή βιομηχανία να μετασχηματιστεί από οικολογική, κοινωνική και οικονομική πλευρά. Σα ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ε, thank you Σας ευχαριστούμε πολύ. Θα δώσουμε τώρα το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα ακολουθήσει και περαιτέρω συζήτηση. Θα ζητήσω τώρα από τον κύριο Κλάου Σούλτ να πάρει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Αγαπητά μέλη, ευρωβουλευτές. Δεν έχουμε διαφάνειες με τα κυριότερα σημεία από ό,τι βλέπω. Και έτσι λοιπόν, αυτό που θα κάνω είναι θα σας δώσω τα μηνύματα που έχουμε να σας διαβιβάσουμε χωρίς διαφάνειες. Δεν θα είναι μεγαλύτερη δυσκολία αυτή για την παρουσίασή μου. Θα έπρεπε να είχαμε τις διαφάνειες. Υπάρχει πρόβλημα. Κάποιος το αντιμετωπίζει από τεχνικής πλευράς για να το ξεπεράσουμε εντάξει. Μα ε, ε, βαίνει καλός εντάξει. Είναι σημαντικό οι διαφάνειες να είναι έτοιμες για την παρουσίαση του συναδέλφου που θα είναι συμπληρωματική στη δική μου παρουσίαση. Προφανώς ε, καλωσορίζουμε αυτή την πρωτοβουλία από τον Ευρωβουλευτή κύριο Γιάννη Γκάιερ και ενδιαφερόμαστε να δούμε ποια θα είναι η τελική η θετική έκβαση αυτής της πρωτοβουλίας. Υπό το πρίσμα μας ε, τονίζει την ανάγκη να υπάρχει μια πιο ολοκληρωμένη προσέγγιση για την βιομηχανική ανανέωση και καινοτομία και ανάπτυξη και την ανάγκη να έχουμε αυξημένη συνεκτικότητα και συνοχή μεταξύ διαφορετικών πολιτικών, όχι μόνο στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και στα κράτη-μέλη και στο περιφερειακό επίπεδο. Είναι σημαντικό να δούμε τι είναι εκείνο το οποίο προχωρεί και προάγει την βιομηχανική ανανέωση και ε, καινοτομία μέσα σε ένα ενρευστό παγκοσμιοποιημένο πλαίσιο και να δούμε οι παλέ συνταγέ λειτουργούν ή όχι. Τι χρειάζεται σε αυτή την περίοδο κρίση ε, να λειτουργήσει καλύτερα, τι πρέπει να πάει καλύτερα. Αυτό κάνουμε από πλευρά Ευρωπαϊκή Επιτροπή και προετοιμάζουμε για την επόμενη πολιετή περίοδο για τα διαθωτικά ταμεία. Η απάντηση μάλλον προδιατυπώνεται στην στρατηγική για το 2020 τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Το κλειδί είναι η καινοτομία φυσικά. Πώ μπορούν να καινοτομήσουν, πώ θα βρουν την σωστή δυνατότητα ω πρώην βιομηχανικέ περιοχέ ή περιφερειακέ περιοχέ περιοχές ε, οι περιοχές υπαίθρου να καινοτομήσουν. Εδώ είναι λοιπόν ο πυρήνας. Για τα επόμενα δέκα λεπτά θα ήθελα να επικεντρωθώ σύντομα και να εισαγάγω όχι σε λεπτομέρειες βέβαια, αλλά την έννοια της εφιούς εξειδίκευσης Τη εφάνταση εφιούς καινοτομία στην εξειδίκευση. Τι κάνουμε και τι πρέπει να κάνουμε για την ανάπτυξη περιφερειακών στρατηγικών, στρατηγικών για την καινοτομία που θα μπορέσουν να λειτουργήσουν καλά. Για να μπορέσουμε να προωθήσουμε την οικονομική μεταρρύθμιση και αναδιαμόρφωση και την βιομηχανική καινοτομία και να σας υπενθυμίσω σύντομα τις θετικές ε, τους θετικούς προσανατολισμούς που είχαμε προετοιμάσει και δημοσιεύσει τα προηγούμενα έτη. Είχατε ήδη ευκαιρία στις τελευταίες συνεδριάσεις σας να ακούσετε έναν δικό μου συνάδελφο που σας επεξήγησε πώς το FES και το ΑΙΦΟΡΟ μπορούν να συνδυαστούν από πλευράς προσέγγισης και ε, προσπάθειας στη στρατηγική μας. Στις κατευθυντήρες γραμμές για τις στρατηγικές για τα κράτη-μέλη, στην προσέγγιση εκ των κάτω προς τα άνω για την προετοιμασία αυτών των δράσεων. Πρώτη διαφάνεια λοιπόν. Ορίστε ευφυής εξειδίκευση. Ένας από τους κύριους πυλώνες ε, για τις νέες ναυαρχίδες ε, στρατηγικής από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι προϋποθέτει αυτό. Προϋποθέτει εντοπισμό, ταυτοποίηση συγκεκριμένου αριθμού προτεραιοτήτων από πλευράς των υπεύθυνων. Να δούμε ποια είναι τα ισχυρά σημεία τους και τα πλεονεκτήματά τους, συγκριτικά πλεονεκτήματα που έχουν. Εδώ επ' αυτόν πρέπει να ε, θεμελιώσουμε και να οικοδομήσουμε. Να υπάρξει ένα ευρύτερο πλαίσιο σε σχέση με την ε, βέλτιστη ε, επίδοση, πώς μπορεί αυτή η καινοτομία να δράσει σε αυτά τα πλαίσια. Προφανώς αυτό θα απαιτεί σαφείς προτεραιότητες που θα πρέπει να έχουν θεσπιστεί και σε βάθος διαβούλευση με τους εμπλεκόμενους. Αυτό είναι αυτό το οποίο εντάσσουμε, συνηφαίνουμε σε αυτή την προσέγγιση από πλευράς μας. Όπως γνωρίζετε, εισαγάγαμε κάποιους όρους και προϋποθέσεις που πρέπει να ισχύουν και να υφίστανται για τις, ε, τα κονδύλια των διαθροτικών ταμείων, ιδιαίτερα για την καινοτομία και την ανάπτυξη. Ωστόσο όμως ε, θα πρέπει 100 δις ευρώ να μπορέσουν να διατεθούν σε σχέση με ε, προσπάθειες δημοσιονομικές από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω αυτών των περιφερειακών ή εξειδικεύσεων θα πρέπει να μπορέσουμε να ενεργοποιήσουμε, να επανενεργοποιήσουμε το ε, οικονομικό δυναμικό των περιφερειών μας ε, και να γεφυρώσουμε το χάσμα μεταξύ έρευνας, ε, καινοτομίας και ανάπτυξης και έτσι να δράσουμε θετικά στη στρατηγική μας. Κάτι το οποίο ουσιαστικά αναπτύσσεται στην ίδια την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και είναι σημαντικό να το τονίσουμε αυτό και πρέπει να ε, επεκταθεί περισσότερο. Σε αυτού του είδους τους προβληματισμούς, τι είναι εκείνο το οποίο προάγει την ανάπτυξη στη σημερινή συγκυρία, βλέποντας τις βέλτιστες πρακτικές, τι έκαναν οι περιφέρειες κατά τελευταία, τις τελευταίες δεκαετίες, πώς μπόρεσαν να αναδιαμορφώσουν και να αναπροσαρμόσουν τις βιομηχανίες τους. Και έχουμε τέτοιες κατηγοριοποιήσεις και συνέργεια επιτόπου που είναι θετικά στοιχεία. Βασιζόμενοι λοιπόν σε σχέση με αυτά τα στοιχεία για την ε, ανάπτυξη ε, θέλω να τονίσω ότι αυτά ε, παληθεύονται και από τον ΩΣΑ από πλευράς του όσα έχουμε πραγματικά εμπλοκή σε αυτή την ευρύτερη ε, συζήτηση για τη νέα βιομηχανική ανάπτυξη, νέα αντιμετώπιση προκλήσεων και καινοτομία και πριν από τα Χριστούγεννα είχαμε αυτή την έκθεση που δημοσιεύθηκε και είχαμε και μια εκδήλωση εδώ στις Βρυξέλλες με τρεις επιτρόπους που συμμετείχαν και παρουσιάστηκε αυτή η έκθεση, η καινοτομία και η καινοτομία για την ανάπτυξη στις περιφέρειες. Ο ρόλος της εφιούς εξειδίκευσης. Αυτός είναι ο σύνδεσμος εδώ προς το θέμα του Γιέντς Γκάια με τις πληροφορίες και τα στοιχεία αυτά που πρέπει να διηθηθούν και να περάσουν στην πρακτική εφαρμογή. Και σε διαφάνεια θα μπορέσουμε να τα εξειδικεύσουμε αυτά σε σχέση με την ευφυή εξειδίκευση. Αυτό το οποίο όμως είναι σημαντικό να τονίσουμε είναι ότι εμείς χρησιμοποιούμε μια ευρύτερη βάση ορισμών για την καινοτομία. Δεν είναι μόνο η υψηλή τεχνολογίας ε, δράση, η, ε, οι νέες επιστήμες και η τεχνολογία για την καινοτομία, αλλά και οργανωτικά η καινοτομία και οι ε, νέες υπηρεσίες, καινοτόμες υπηρεσίες. Πολλά πρέπει να αντιληφθούμε πώς πρέπει να λειτουργήσουν σωστά σε σχέση και με τις δημόσιες προμήθειες και αγορές. Αν έχουμε καλύτερες δημόσιες δημόσιες υπηρεσίες, ε, καινοτομία. Όλα αυτά είναι προσεγγίσεις και στοιχεία που διαρκώς μπορούμε να τονίζουμε και να υπογραμμίζουμε και σε σχέση με τις ε, καινοτομίες στις υπηρεσίες, στον τουρισμό, στις ε, διαφορετικές εξειδικευμένες βιομηχανικές δράσεις. Η ευφυής εξειδίκευση δεν σημαίνει ότι μόνο με υψηλή τεχνολογία high-tech θα εργαστούμε. Πρέπει να δούμε πού είναι το βέλτιστο, μέγιστο δυναμικό μας και εκεί να επιλέξουμε και να αποφασίσουμε πού θα επικεντρώσουμε τους πόρους μας για τα επόμενα επόμενα 5 ή 10 έτη με μια σαφή προοπτική για την ανάπτυξη που θα έχει συμφωνηθεί συνενετικά με τους εμπλεκόμενους επιτόπου. Είναι μια, ας το πω έτσι, αναδιαμόρφωση, μια επαλήθευση αυτών που έχουν προηγηθεί και ενισχύονται αυτά με μια πιο ενδυναμωμένη και πιο αυστηροποιημένη, επικαιροποιημένη ε, διαδικασία. Με αυτή την ευφυή εξειδίκευση, αυτό το ενέταξα στην παρουσίασή μου, γιατί ζητήθηκε να γίνει παρέμβαση για τις ε, ε, τεχνολογίες ε, που έχουν σημαντικό ρόλο και που θα πρέπει να πούμε ότι βλέπετε εδώ στη διαφάνεια ποια είναι αυτά τα θέματα ξεχωριστά. Και το ITT είναι ένα από τα πιο σημαντικά στοιχεία των νέων τεχνολογιών που όμως δεν έχουμε εδώ περισσότερα στοιχεία εξειδίκευσης. Αυτά μπορούν να είναι στοιχεία για μια ανάπτυξη των ε, ε, βιομηχανιών μας. Είτε θα υπάρξει καινοτομία, είτε θα ε, αναγκαστικά θα αποκλειστούν πολλοί από το πεδίο δράσης και βλέπουμε και το θέμα της περιφερειακής ανάπτυξης ε, που την χάνει ιδιαίτερου ενδιαφέροντος. Αν η υποστήριξη δεν θα είναι μόνο στα θέματα υποδομής και θεμελιώδους έρευνας ε, για την επόμενη περίοδο ε, είπαμε ότι είναι επιλέξιμο το να μπορεί κανείς να ε, έχει από πλευρά μικρομεσαίων επιχειρήσεων υποστήριξη ώστε να προσεγγίσει καλύτερα τι ανάγκε των αγορών, να υπάρξει ε, εξειδίκευση όσον αφορά τι υπηρεσίε και ε, τα προϊόντα αυτών των υπηρεσιών. Εργαζόμαστε πολύ στενά με όλους τους αρμόδιου για να υπάρξει η δραστηριοποίηση για την για τον εξυγχρονισμό που είναι πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο. Δεν έχουμε ε, ούτε προσκόμματα που να δημιουργούνται, που να δημιουργούμε, είτε όρους και προϋποθέσεις που να δυσχεραίνουν ε, τις ε, δράσεις μας σε σχέση με την εφαρμογή αυτών των νέων τεχνολογιών και καινοτόμων δράσεων που πρέπει να υποστηρίξουν την Ευρώπη. Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο είναι η εξωτερική συνεργασία με αυτές τις περιφέρειες. Εδώ, ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία περιφερική συνεργασία. Οι ευφυείς ε, στρατηγικές δεν είναι στρατηγικές μόνο μέσα στις ίδιες τις περιφέρειες για να μπορέσει να ε, επιταχυνθεί η διεργασία και να λειτουργήσουν οι εντός εισαγωγικών έλικες ε, προώθησης και συνεργασίας. Όλα αφορούν βέβαια τη συνεργασία σε ένα ευρύτερο πλαίσιο. Ωστόσο από την άλλη πλευρά πρέπει να επικεντρωθούμε στην δημιουργία μιας κριτικής κρίσιμης γνώσης ε, που μπορεί να μας δώσει ε, την εξειδίκευση αυτών των περιφερειών. Πάντα θα υπάρχει ανταγωνισμός μεταξύ περιφερειών, αλλά θα πρέπει πιο διαρθρωμένα και συστημικά να προσεγγίζουμε αυτή τη συνεργασία. Όχι μόνο εκ των κάτω προς τα άνω υποστήριξη αυτών των ε, ε, πρωτοβουλειών όπου αναφύονται, αλλά να δούμε πώς μπορούμε να εξειδικευτούμε με τέτοιο τρόπο ώστε παγκόσμια να είμαστε ανταγωνιστικοί και με τη βέλτιστη επίδοση από πλευράς μας. Έτσι η ευρωπαϊκή εδαφική, η περιφερειακή συνεργασία μέσα σε αυτό το νέο πλαίσιο ανακτά, α το πω έτσι, νέα σημασία και σπουδαιότητα για την δημιουργία αυτών των ε, ε, βάσεων, αυτών των ε, κατηγοριοποιημένων δράσεων μέσω των καινοτόμων ευρωπαϊκών συνεργασιών και μπορούμε έτσι να πούμε ότι σε σχέση με την κατανόηση αυτού του πλαισίου θα μας δώσει τη δυνατότητα να δραστηριοποιηθούμε αποτελεσματικά θα ενισχύσουμε την υποστήριξη της κατηγοριοποίησης και ομαδοποίησης περιφερειακά επιχειρήσεων και ε, καινοτόμων δράσεων θα μπορέσουν οι εμπλεκόμενοι να ενδυναμώσουν περισσότερο τις επιδόσεις τους μέσα από αυτές τις δράσεις και σε σχέση με την ε, ε, ε, Επιτροπή Ιντερεγ για παράδειγμα και άλλες παρόμοιες δράσεις θα τύχουμε εξειδίκευσης αποτελεσματικής. Θέλω επίσης να τονίσω και κάτι άλλο η εκ των κάτω προς τα άνω προσέγγιση στην ταυτοποίηση μελλοντικών ενδυνάμει πεδίων για αυτή τη δραστηριοποίηση και αυτό είναι ένα στοιχείο που έχει ιδιαίτερη σπουδαιότητα. Η προτεραιοποίηση ε, θεμάτων δεν θα πρέπει να είναι μόνο αποκλειστικός ρόλος ε, των κρατικών αρχών, μια επιλογή εκ των άνω προς τα κάτω, επιλογή και απόφαση από τις κρατικές αρχές που βρίσκεται το δυναμικό και τι πρέπει να γίνει. Πρέπει να υπάρχει αμφίδρομη, διαδραστική προσέγγιση από τους εμπλεκόμενους. Τα πανεπιστήμια για παράδειγμα, τα ερευνητικά κέντρα όλοι αυτοί να εμπλέκονται. Να εμπλέκονται μέσα στο στόχο, ευρύτερο στόχο του να ευθυγραμμίζονται οι δικές τους, ε, οι δικές τους θεματολογικά ε, εργασίες ε, προς αυτούς τους στόχους. Διαφορετικά δεν θα υπάρχει η μάζα εκείνη που είναι αναγκαία από πλευράς τεχνογνωσίας και χρηματοδότησης και κονδυλίων για να μπορέσουν να λειτουργήσουν αποτελεσματικά οι δράσεις. Είναι περιορισμένα τα κονδύλια και πρέπει με το βέλτιστο τρόπο να χρησιμοποιηθούν με την βέλτιστη η ευφυή λοιπόν εξειδίκευση μπορεί να είναι ένα τέτοιου είδου ισχυρό χαρτί που θα εστιάζεται στην βιομηχανική καινοτομία και ανανέωση και πολυμορφοποίηση, πολυσχηδή δραστηριοποίηση ώστε να υπάρξει το βέλτιστο αποτέλεσμα. Επίσης απαιτεί ισχυρό συντονισμό ε, εγκάρσια και κάθετα για την τεχνολογία των συνέρευνα, βιομηχανική πολιτική, ε, πολιτική για την αγορά ε, για τα εργασιακά θέματα. Πρέπει να υπάρξουν συντονιστικές δράσεις μεταξύ αυτών των διαφορετικών πεδίων. Ε, οι στρατηγικές για την ανάπτυξη δεν μπορούν να ε, εκπονούνται στεγανά, σε στεγανό πλαίσιο χωρίς να συνεργάζονται άλλοι τομείς και χωρίς διαβούλευση Υπουργείων και αρμόδιων αρχών σε ευρύτερο πλαίσιο. Τώρα, αυτό που θα ήθελα να τονίσω επίσης είναι η διάσταση όσον αφορά τις πόλεις, τα αστικά κέντρα σε σχέση με όλα αυτά. Δυστυχώς οι συνάδελφοι από την Μονάδα Αστικής Ανάπτυξης των Αστικών Κέντρων δεν μπόρεσαν να προσέλθουν. Συμβαίνουν τόσα πολλά αυτή τη στιγμή και έχουν ανελημμένες υποχρεώσεις και σε άλλα, για άλλα θέματα με το Ευρωκοινοβούλιο και δεν μπορούν να παραστούν. Υπόσχομαι όμως να διαβιβάσω τα μηνύματα και τις απόψεις σας ώστε να υπάρξει αυτός ο συνδυασμός με αυτούς σε αυτή την προσέγγιση. Και θα, ολοκληρώσω. Ενώ τώρα η ευφύης εξειδίκευση πρέπει να εφαρμόζεται στις ε, περιφέρειες έχει επιπτώσεις σημαντικές και για την ανάπτυξη και των αστικών κέντρων. Δεν χρειάζεται να, το, ε, να επιμείνω περισσότερο και για τον περίγυρο αυτών των αστικών κέντρων. Για να μπορέσουν να επιτύχουν τους αναπτυξιακούς, του τους στόχους ε, τα αστικά κέντρα μέσα σε ένα σαφές πλαίσιο όσον αφορά το όραμα για την χρήση αυτών των κονδυλίων για την επίτευξη αυτών των στόχων. Ιδιαίτερα όσον αφορά βιομηχανικές από πλευρά της Ευρωπαϊκής ε, ε, Επιτροπής ε, έχει ε, προκαιρού προετοιμαστεί και ε, προλιανθεί το έδαφος και όχι, δεν επικεντρώνεται μόνο σε θέματα ευφυούς εξειδίκευσης ή ανάπτυξης αλλά και σε πολλά άλλα θέματα που είναι αναγκαία για να επανέλθουν σε μια ε, ορθή πορεία οι πόλεις και να αντιμετωπιστούν για παράδειγμα οι περιβαλλοντικές προκλήσεις και άλλες προκλήσεις. Είναι περίπλοκα τα θέματα όσον αφορά τις πόλεις και τα προβλήματα αλλά και οι ευκαιρίες που παρουσιάζονται. Θα πρέπει να μπορέσει να εξειδικευτεί στρατηγική στο δυναμικό που θα μπορέσουμε να κινητοποιήσουμε Γι' αυτό η εξειδίκευση όσον αφορά αυτά τα θέματα μπορεί να βοηθήσει πάλι μεθοδολογικά ως ένα μέσο, ως ένα εργαλείο για να επαυξήσουμε το σχεδιαστικό δυναμικό μας και το δυναμικό μας για τον προγραμματισμό για να προχωρήσει ε, η οικονομική, ο οικονομικός μετασχηματισμός και να αναδιαμορφωθούν οι πόλεις και 5% από το ε, Ευρωπαϊκό Περιφερειακό Ταμείο ε, για παράδειγμα σε σχέση με αυτές τις δράσεις αυτή την ολοκληρωμένη προσέγγιση για, τα, για τις πόλεις δεν προβλέπουμε ε, τίποτα. Ενθαρρύνουμε τις πόλεις να χρησιμοποιήσουν την, τον ευφυή e στρατηγικό σχεδιασμό ο, η, ο, e, η e εξειδίκευση δίνει δυνατότητες. Αν τώρα μεγάλα αστικά κέντρα θέλουν και επιθυμούν να επιλέξουν αυτό το εργαλείο και να το χρησιμοποιήσουν, ευπρόσδεκτο θα είναι. Βλέπουμε ότι υπάρχει και συνοχή και συνεκτικότητα και συγγένειες και συνέργειες που μπορούν να απορρέψουν για αυτά τα οποία μπορούν να γίνουν για τις πόλεις. Αυτό που προσπαθούμε δηλαδή να επιτύχουμε για καλύτερες στρατηγικές καινοτομίες στο στρατηγικό επίπεδο και να τα συναθρήσουμε όλα αυτά και να ολοκληρώσουμε. Ο ευφυής αυτός ε, ε, σχεδιασμός για την εξειδίκευση μπορεί να έχει θετικά αποτελέσματα και για τις πόλεις και για τις πρώην βιομηχανικές πόλεις αλλά και για τις ε, περιοχές της υπαίθρου. Αυτό που κάνουμε σε αυτή τη φάση, αυτή τη στιγμή είναι και θέλω να το καταδείξω αυτό στην επόμενη διαφάνεια είναι εργαζόμαστε με πολλές περιφέρειες και μάλιστα σε βάθος και με ιδιαίτερα εντατικό τρόπο. Σε, αυτό, σε αυτή την πλατφόρμα F ευφυούς εξειδίκευσης. Μπορείτε να δείτε στη διαφάνεια τις περιφέρειες εκείνες. Συγγνώμη, μου έχουν ανάψει εδώ το κόκκινο λαμπάκι οι διερμηνείς που σημαίνει πρέπει να επιβραδύνετε λίγο γιατί τρέχετε υπερβολικά, βιάζεστε κατά την ε, εκφορά του λόγου σας. Ζητώ συγγνώμη για αυτό, λέει ο μιλητής και επιβραδύνει υπερβολικά. Δεν θέλω να σας επιβραδύνω. Λοιπόν, παραμένοντας ε, στη διαφάνεια, βλέπετε το εύρος της προσπάθειας που καταβάλουμε για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε σε σχέση με τις περιφέρειες, σε σχέση με την εξειδίκευση αυτή, ευφύη εξειδίκευση. Και από πλευράς λοιπόν των, της, της περίοδου, ε, από πλευράς ε, των διαθωτικών ταμείων, τι κάνει αυτή η πλατφόρμα. Έχουμε πάνω από 100 περιφέρειες. Κάποιες χώρες έχουν λοιπόν καταχωρήσει και ε, εγγράψει ε, αυτά τα στοιχεία τα οποία ε, θα βρίσκονται υπό την, υπό την αιγίδα του Κοινού Κέντρου Ερευνών. Θα έχουμε λοιπόν από ειδικού αναλύσεις και αξιολογήσεις συλλογή δεδομένων για την αξιολόγηση. Διατίθεται πραγματογνωμοσύνη που μπορεί να βοηθήσει αυτές τις περιφέρειες. Πολλά έχουν γίνει ήδη. 58 συμβάσεις έχουμε συνάψει όπου οι πραγματογνώμονες μεταβαίνουν σε αποστολές επιτόπου σε αυτές τις περιφέρειες και αξιολογούν αυτές τις στρατηγικές για την καινοτομία και μπορούν να βοηθήσουν και βοηθούν τις περιφέρειες και τις κρατικές αρχές των κρατών μελών για αυτές τις διεργασίες που μπορούν να οδηγήσουν τελικά σε μια ευφυή εξειδίκευση για αυτές τις ε, πρωτοβουλίες καινοτομία για τις περιφέρειες. Τώρα, βλέπετε εδώ στην επόμενη ε, διαφάνεια ε, στοιχεία για αυτή την εξειδίκευση. Θεματολογικά καλύπτονται διαφορετικά πεδία. Αν δούμε όλα αυτά με τη διασύνδεση των πανεπιστημίων για την καινοτομία και τις ε, ευθύς ε, εξειδικεύσεις βλέπουμε εδώ πώς μπορεί να υπάρξει συνδυασμός της εξειδίκευσης και της καινοτομίας και των επιστημών και όλα αυτά τα στοιχεία θα είναι διαθέσιμα όσον αφορά προσανατολισμούς και βέλτιστες πρακτικές που θα είναι στη διάθεση των ενδιαφερομένων. Είμαστε πάρα πολύ καλά, έχουμε πολύ καλά προετοιμαστεί για την επόμενη περίοδο, για το μέλλον στη διάθεση αυτών των στοιχείων. Θεωρούμε ότι η ιδέα της ε, ευφυούς εξειδίκευσης θα μπορέσει να βρει τρόπο να ε, παρισφρήσει σε αυτά τα πλαίσια, πώς μπορεί αυτό να βοηθήσει δηλαδή την βιομηχανική καινοτομία και βιομηχανική ανάπτυξη, συνάγοντας τα συμπεράσματα από όσα κάναμε καλά αλλά και από όσα δεν πήγαν τόσο καλά. Κάνοντας δηλαδή σωστά τη δουλειά μας και υποστηρίζοντας αυτή την πορεία στο μέλλον. Επακούμε σε αυτά και θα ήθελα να δώσω τον λόγο στον επόμενο αγορητή. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Θα Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσίαση. Θέλω να δώσω το λόγο τώρα σε κάποιον από τον Κριστιαν Σομπλένς, Γκάμπριελ Κρίν, Κάτια Ρέπελ. 10 με 12 λεπτά παρακαλώ όμως. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, διακεκριμένοι βουλευτέ, σας ευχαριστώ πολύ που με καλέσατε σήμερα στην Επιτροπή σας. Θα ήθελα να σας δώσω λαβή προς ε, σκέψη, τροφή προς σκέψη μάλλον, και θα να δούμε βασικά τα εξή. Πρώτα απ' όλα ποιο είναι το νέο πλαίσιο για τις βιομηχανικέ περιοχές και την περιφερειακή στρατηγική, τι καινούργιο υπάρχει για την περιφέρεια, για τις ε, βιομηχανίες και αν χρειάζεται κάποια νέα υπηρεσία ή νέες υπηρεσίες υποστήριξης. Έχει σχέση και με την προηγούμενη παρουσίαση αυτό. Λοιπόν, Σήμερα σε όλους τους τομείς βλέπουμε κατακαιρματισμό ε, στην, ε, αξία, στην αλυσίδα αξίας ε, στις εταιρείες. Επίσης βλέπουμε να υπάρχει δυνατότητα μετεγκατάστασης οπουδήποτε. Το θέμα όμως είναι η παραγωγή καλών στοιχείων για μια εταιρεία ώστε να είναι assets όπως τα λέμε για να είναι ελκυστική. Θα πρέπει λοιπόν να Υπάρχουν διάφορα εργαλεία, όχι μόνο καινοτομία, αλλά και η επίδειξη, η ανάπτυξη, η τυποποίηση. Και επίσης θα πρέπει να επεξεργαστούμε και τα προσόντα ε, μιας περιοχής και το ανθρώπινο δυναμικό αλλά και τα είδη βιομηχανικών υπηρεσιών και το κοινωνικό κεφάλαιο που υπάρχει στην συγκεκριμένη περιφέρεια και θα πρέπει αυτό να κινητοποιηθεί για τους στόχους που έχουν τεθεί. Πρέπει λοιπόν να πω ότι η ιδέα τη ειδίκευση είναι κάτι θετικό γιατί βασίζεται στο τι μπορούμε να αποκομίσουμε, τι καλύτερο μπορούμε να αποκομίσουμε το καθένα. Το δεύτερο είναι η λεγόμενη θεωρία σάντουιτς για την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων. Έχουμε ε, κάποιες επιχειρήσεις που έχουν πολύ ε, καλές μάρκες, πολύ καλή ποιότητα και έχουμε όμως και του χαμηλού κόστους. Και υπάρχει στο μεσοδιάστημα πολλές άλλες επιχειρήσεις. Αυτό ε, τώρα το slide το έφτιαξα πριν από δύο χρόνια και η πεζό μάλλον δεν θα μπαινε στη μέση και το BMW θα πήγαιναν στην πάνω-πάνω, στην κορυφή της πυραμίδας. Τέλος πάντων, στην κορυφή μπορούμε να βάλουμε το Cambridge, τη Βαβαρία, κάτω μπορούμε να βάλουμε τις περιοχές του Νότου ενδεχομένως. Αλλά ποιο είναι το μέλλον για μια ε, περιοχή που ήταν παλιά βιομηχανική, Λορένη για παράδειγμα κτλ τι προσέγγιση πρέπει να ακολουθήσουν για το μέλλον, πώς θα εξασφαλίσουν την ανταγωνιστικότητά τους με το χαμηλό κόστος. Μπορούν να μπουν σε μια ε, σε ένα εξαιρετικό προσοδοφόρο μικροτομέα της αγοράς ή όχι. Τι μπορούμε να κάνουμε πρώτα απ' όλα. Θα πρέπει να δώσουμε σίγουρα χρήματα για την έρευνα ε, και την ε, ανάπτυξη. Αλλά έχουμε και νέους τομείς νάνο, βιοτεχνολογίε, ηλιακή ενέργεια. Ε, τι κάνουμε εκεί. Έχουμε διπλώματα ευρεσιτεχνία, ε, έχουμε επενδύσει στην έρευνα. Πού είναι όμω οι ευρωπαϊκέ εταιρείε. Άρα μπορούμε να κάνουμε ε, κάτι για να βρούμε μια γέφυρα σε περιφερειακό ε, επίπεδο για να έχουμε αποτελέσματα και στον τομέα τη χρηματοδότηση, στο χρηματοπιστωτικό, αλλά και στην εμπορία, αν θέλετε. Τη διάθεση του ερευνητικού αποτελέσματο στο εμπόριο. Για να το πετύχουμε αυτό, θα πρέπει να δούμε το περιφερειακό επίπεδο διαφορετικά πώς η γνώση περνάει στην αγορά. Όπως σας είπα, έχουμε καλή έρευνα, παράγουμε ε, και διαχέουμε τη γνώμη, ακόμη και σε εξειδικευμένα περιοδικά επιθεωρήσεις και λίγο πολύ προστατεύουμε τη γνώση μας. Ποιος όμως αξιολογεί το δυναμικό, τις δυνατότητες της γνώσης ε, που παράγεται από τους ερευνητές μας και προς όφελος της αγοράς αλλά και υπέρ των μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε τοπικό επίπεδο που έχουν τη δυνατότητα να διχειριστούν την καινοτομία ή να την απορροφήσουν. Και έπειτα το θέμα είναι εάν έχουμε ανοιχτή πηγή IPR ή αν δίνουμε την άδεια σε μια υφιστάμενη επιχείρηση. Το έχουμε συζητήσει σε, ε, με πολλές επιχειρήσεις και αναγνωρίζουν ότι δεν αξιοποιούνται παρκώς περιφέρεια και πρέπει εκεί να επιτευχθεί περισσότερη πρόοδος. Ένα άλλο ζήτημα είναι πώς αναγνωρίζουμε την λεγόμενη επιχειρηματική διαδικασία ανακάλυψης, entrepreneurial disclosure Ποιο Ποιος μπορεί να δώσει 10 επιχειρήσεις που πρόσβατα επένδυσαν σε νέα τεχνολογικά προγράμματα ή τεχνολογίες, νάνο, βίο, τεχνολογίες, ρομποτική, είτε για τη χρησιμοποίηση τεχνολογίας, είτε γιατί τις πολλούν. Ή ποιος μπορεί να μου δώσει 10 μικρομεσαίες επιχειρήσεις που εργάζονται στον παραδοσιακό, το, στους παραδοσιακούς κλάδους και χρησιμοποιούν αυτές τις ε, βασικές τεχνολογίες γενικής ε, εφαρμογής, τα key enabling technologies δηλαδή ή σε μη, με μη εμπορεύσιμε υπηρεσίε και προϊόντα. Πείτε μου εταιρείε που έχουν αυξήσει την παραγωγικότητά του. Ή στον κατάλογο βλέπετε κάποιες επιχειρήσεις που παρέχουν εξειδικευμένες υπηρεσίες που έχουν με του κεφαλαίου ή των πραγματικών δικαιωμάτων ή ανταμείβουν καινοτόμο προσωπικό οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις Όλα αυτά σας τα να σας δείξω ότι σήμερα, αν έχουμε μια πολιτική κλάστερ ομαδοποίησης, καλό είναι καλής να επενδύει στην μεταξύ τους συνεργασία. Μπορούν βέβαια να ομαδοποιηθούν όλες οι εταιρείε που δραστηριοποιούν στον τομέα των ε, πληροφοριών και επικοινωνιών. Αλλά το θέμα είναι πώς μπορούν να συνεργαστούν. Και έρχομαι σε αυτό που είπε ο Κλάους, ότι αυτό που χρειάζεται είναι διαπεριφερειακή συνεργασία. Δεν μπορεί κανείς να πει ότι έχει σε μία περιφέρεια 20 εταιρείε κορυφαίες ή κλάστερ κορυφαία. Πώς θα προωθήσουμε και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, έχουμε πάρα πολλά στοιχεία, δεν θα σε άλλες λεπτομέρειες. Θέλουμε όμως και ένα μύθο να τον θέσουμε από αμφισβήτηση. Έχουμε ακούσει πολλέ φορέ ότι οι μικρομεσαίε επιχειρήσει δημιουργούν πλούτο, δημιουργούν θέσει εργασία. Ξέρετε, δεν είναι αλήθεια αυτό. Λίγε μόνο το πετυχαίνουν. Πάνω από 75% των μικρομεσαίων δεν έχουν διάρκεια ζωή πάνω από 5 χρόνια, άρα δεν τα προσφέρουν όλα αυτά οι μικρομεσαίε επιχειρήσει. Θα πρέπει να επικεντρώσουμε σε έναν αριθμό συγκεκριμένων, όχι σε όλε τι μικρομεσαίε επιχειρήσει. Αυτέ οι λίγε που το πετυχαίνουν και όχι οι πολλέ και σε ό,τι αφορά οι δημόσιε αρχέ. Η καινοτομία είναι καρπό τη γνώση ή τη υψηλή τεχνολογία. Άλλο μύθο αυτό. Δεν είναι αλήθεια, το είπε και ο Κλάου. Έχουμε ε, καινοτόμε επιχειρήσει, καινοτόμο σχεδιασμό, έχουμε κάποια επιχειρησιακά μοντέλα ή και καινοτομία σε ό,τι αφορά και τον τρόπο ζωή, το lifestyle ή νέα διαδικτυ... νέα δίκτυα πρακτικών πόσες μορφές καινοτομία βλέπουμε σε αυτό το δρόμο εδώ στην Κοπενχάγη. Αν μιλήσει κανείς με αυτόν τον τύπο εκεί πέρα, θα σας πει δεν ενδιαφέρεται να διαθέσει τα προϊόντα στο εμπόριο. Και αυτό είναι και ένα ζήτημα με την επιχειρηματικότητα. Πουλάω τύπος εκεί τα προϊόντα του πώς θα μπορεί να υπάρξει ανταγωνισμό με το Starbucks τι είδους υπηρεσίες πρέπει επίσης να μπορούμε να παρέχουμε ε, σε επίπεδο εμείς, μικροπιστήριων, δηλαδή επιχειρήσεων ή μεγαλύτερων επιχειρήσεων σε μια περιφέρεια. Εάν θέλουμε να είμαστε πρώτοι, να είμαστε πρωταγωνιστές, πρέπει πρώτα απ' όλα να έχουμε το απαραίτητο προσωπικό και υπηρεσία χρηματοοικονομικής υποστήριξης, ταμιακά διαθέσιμα ή ταμιακά ισοδύναμα, τι ε, παρέχουμε, τι προσφέρουμε, διαχείριση, απόκτηση γνώσεων και μετά βλέπουμε αν θα κάνουμε coaching, καθοδήγηση, αν θα κάνουμε ευαισθητοποίηση, παρέχουμε πληροφορίες για την αγορά τεχνολογία ή επικεντρωνόμαστε πιο πολύ στο ανθρώπινο δυναμικό μιας εταιρεία και βέβαια μετά υπάρχουν και τα χρηματοοικονομικά εργαλεία, μετοχές κτλ. Και επίσης πολλές φορές Ακούω ότι το κεφάλαιο επιχειρηματικού κινδύνου του σχετική αγορά είναι μια δομική αστοχία ε, της αγοράς. Δεν είναι αλήθεια αυτό. Το θέμα είναι αν έχει καλή απόδοση, αν είναι υπερβολικά παρακινδυνευμένα τα πράγματα, δεν επενδύει κανεί σε αυτά. Αν αρχίσει κανεί να λέει όμω ότι ίσω αυτό είναι ο λόγο για τον οποίο κτλ., τότε μπορεί να παράσχει κανεί άλλε υποστηρικτικέ υπηρεσίε. Καλύτερη συμβουλή στον τομέα IPR ή πρωτότυπο επίδειξη κτλ. Οπότε ο τελικό επιχειρηματίας όταν έλθει απέναντι στους επενδυτές του θα είναι έτοιμος. Και τέλος που θέλω να τονίσω, ίσως να υπάρχουν 30 ή 40 βιβλία που μπορεί κανείς να ε, διαβάσει για το πώς θα φτιάξει μια Silicon Valley στην ανοτεχνολογία, δεν ξέρω εγώ τι. Ποιος όμως ε, αγοράζει, αν υπάρχει βιβλίο που να λέει, πώς μπορεί η αριστεία να φτιάξει την αριστεία, αλλά να την αξιοποιήσει και να την μεταφέρει κάπου αλλού να κάνει ένα μοντέλο δηλαδή για μεταφορά της ροής ε, πληροφοριών από τη μια περιφέρεια στην άλλη για δραστηριότητες ε, ε, που βασίζονται στον άνθρωπο, για παράδειγμα. Έχουμε διάφορα προγράμματα, έχουμε το Εράσμος για παράδειγμα, αλλά εσείς πόσοι από εσάς έχετε πάει σε μια συνεδρίαση που την μάλλον σε μια διάλειμμα που την κάνει κάποιος που έχει πάρει με υποτροφία Εράσμους ή Μαρή Κιουρί για παράδειγμα. Άλλες δραστηριότητες, ε, δραστηριότητες που βασίζονται στην ε, κοινότητα, κάποιες εκθέσεις, κάποια ε, εμπορικά σαλόνια. εργαστήρια και συνέδρια κτλ. Και τέλος μπορεί κανείς να εστιάσει σε ε, κάποιες εταιρίες που δεν θα περιορίζονται στις εξαγωγές, γιατί δεν είναι οι αγορές το μόνο. Τι πρέπει να αποφύγουμε τώρα. Πρώτα απ' όλα, πρέπει να μειωθεί το χάσμα μεταξύ προσφοράς και ζήτησης. Δεύτερον, πρέπει να δούμε τον μετασχηματισμό και όχι τις συναλλαγές. Transformation και όχι transaction. Μπορεί να έχει δαπανηθεί ένα εκατομμύριο ή ένα δισεκατομμύριο και όλοι είναι ικανοποιημένοι. Πού οδήγησε αυτό όμω, υπήρξε μετασχηματισμό, υπήρξε αλλαγή. Επίση, κεφάλαιο. Επενδύουμε κάποια από εσά σε μια περιφέρεια. Πού πάνε όμω, τι σημαίνει αυτό. Επίση, είμαστε οργανοκεντρικοί. Υπερβολικά ε, οθούμενοι από την πολιτική ενδεχομένω. Τώρα έχουμε τον ορίζοντα 2020, πριν ήταν στην ε, ατζέντα τη Λισαβόνα. Τι γίνεται όμω σε βιομηχανικό επίπεδο, τι γίνεται σε περιφερειακό επίπεδο. Ή κάποιε φορέ είμαστε κοντόθεροι, εστιάζουμε στο πολύ βραχυχρόνιο διάστημα και τελικά είμαστε άκαμπτοι ε, στον προγραμματισμό μας. επιση βασιζόμαστε προβολικά στι επιδοτησει και πολλε φορε δεν είναι καλή η γνώση μα ε, η διαχείριση μάλλον των γνώσεων. Νομίζω ότι σας έδωσα αρκετή τροφή για συζήτηση. Να κάνω μια σύνοψη. Πρώτα απ' όλα πρέπει να επιλέξουμε το αναγκαίο, να εκμεταλλευτούμε το δυναμικό των περιφερειών και επίσης κατάτμιση. Κατάτμιση τύπων και κατάτμιση ΜΜΕ για να έχουμε τις κατάλληλες υπηρεσίε, τις χρηματοδοτικές και μη χρηματοδοτικές. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ας ξεκινήσει λοιπόν η συζήτηση. Λάμπερτ η πρώτος. Ευχαριστώ, θα σύντομος. Είμαστε στην αρχή του τεράστιου αυτού ζητήματος και κατά τη διάρκεια της συζήτησης θα πρέπει να δούμε σε ποια θέματα πρέπει να εστιαστούμε ουσιαστικά στην έκθεσή μας που αναφέρεται στις περιφερειακές στρατηγικές για τις βιομηχανικές περιοχές στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε σχέση πάντα λοιπόν με την περιφερειακή πολιτική θα πρέπει να εστιαστούμε στο ζήτημα αυτό. Και λάβαμε κάποιες πολύ σημαντικές πληροφορίες για τα μέσα εκείνα τα οποία ενδεχομένω να μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε. Η Επιτροπή Περιφερειακής ε, Ανάπτυξης και συγκεκριμένα DG Region αν δεν κάνω λάθος, και ο κύριος Σταγιάννη παρουσίασαν μία πολιτική για τη βιομηχανία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Από την άλλη έχουμε και την Επιτροπή Ήτρε που αναφέρθηκε σε κάποιες πολιτικές καινοτομίας για την Ευρωπαϊκή Ένωση και το πώς θα καταφέρουμε να πετύχουμε μια Ευρωπαϊκή Ένωση καινοτομίας. Θεωρώ λοιπόν ότι η προσέγγιση είναι αρκετά σφαιρική και ολοκληρωμένη. Σε δύο εβδομάδες η πρώτη αντιπροσωπεία της ε, Επιτροπής ε, Ήτρε θα πάει στη Σεβίλη προκειμένου να μελετήσει πραγματικά αυτά τα οποία ακούσαμε πριν από λίγα λεπτά. Από την οπτική γωνία βέβαια της Επιτροπής Γεωμηχανίας θα γίνουν αυτά. Βρισκόμαστε πλέον λοιπόν σε μια χρονική φάση που μπορούμε να αρχίσουμε να συνδυάζουμε διαφορετικές πολιτικές, διαφορετικές οπτικές γωνίες προκειμένου να καταφέρουμε να έχουμε μια καλύτερη πολιτική για τη χρονική περίοδο 2014-2020 και θεωρώ ότι είναι σαφές ότι η έννοια αυτή της ευφυούς εξειδίκευσης, ιδίως για τις βιομηχανικές περιοχές, αποτελεί μία προϋπόθεση στα πλαίσια του συστήματος αιρεσιμότητας, δηλαδή ότι θα πρέπει στις συμφωνίες εταιρικής σχέσης οι πόλεις, οι περιφέρειες να υποβάλουν τέτοια προγράμματα επιχειρησιακά τα οποία εμπνέονται από την ευφυή εξειδίκευση. Δεν ξέρω αν όμως όλες αυτές οι χώρες θα καταφέρουν ε, σε αυτό το σύντομο χρονικό διάστημα να έχουν ε, απτά αποτελέσματα. Ενδεχομένως να πρέπει να κατευθύνουμε κάπως περισσότερο τις χώρες αυτές βάσει των βασικών αυτών προϋποθέσεων που περιλαμβάνονται στα πλαίσια του συστήματος αιρεσιμότητας και να τους δώσουμε λίγο ακόμα χρόνο, ενδεχομένω να τους επιτρέψουμε τα επόμενα βήματα να τα κάνουν μέσα στα επόμενα χρόνια και όχι σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Βλέπω εδώ πέρα τα έγγραφα τα οποία μας δόθηκαν και θεωρώ ότι ε, το Κοινοβούλιο και οι συνάδελφοι έχουν απόλυτο δίκιο όταν λένε ότι, για παράδειγμα, αναφερθώ σε ένα σημείο της παρουσίασής σας, ότι ο τομέας της πληροφορικής θα πρέπει προφανώς να βρίσκεται, να είναι παρόν σε όλες τις περιφέρειες, γιατί καταλαβαίνετε ότι εδώ πέρα υπάρχουν πολύ μεγάλες ευκαιρίες χρηματοδότησης. Επίσης, η δημιουργική βιομηχανία είναι πάρα πολύ σημαντική. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να επιτρέψει επενδύσεις στον τομέα αυτό. Θεωρώ λοιπόν πραγματικά ότι ο τομέας αυτός, καθώ επίσης και κάποιοι άλλοι τομείς, είναι πάρα πολύ σημαντικοί προκειμένου να προωθήσουν περισσότερο την ανάπτυξη. Δεν ξέρω αν εμείς στη δική μας την έκθεση θα καταφέρουμε να καλύψουμε όλες αυτές τις διαφορετικές πτυχές ή αν θα πρέπει να προβλέψουμε και μία ακόμα μελέτη η οποία επικεντρωθεί πολύ περισσότερο στην ευφύ εξειδίκευση. Νομίζω ότι στον φετινό μας προγραμματισμό θα πρέπει να προβλεφθεί και μια δημόσια ακρόαση για την ευφύ εξειδίκευση και θα πρέπει ενδεχομένως και στο μέλλον να έχουμε και μία άλλη μελέτη για την ευφύ εξειδίκευση. Γιατί όπως είπαμε η έκθεσή μας η σημερινή εστιάζεται στις βιομηχανικές περιοχές στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κάρι Μαντέλη. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ για την παρουσίαση αυτή. Εγώ δεν θα ήθελα οι δικές μας οι ευρωπαϊκές υπεριφέρειες να γίνουν Silicon Valley, σας το ξεκαθαρίζω αυτό από την αρχή. Νομίζω ότι οι περιφέρειές μας έχουν πραγματικά μια τοπική νοοτροπία, ένα τοπικό πολιτισμό, τοπικές ιδιαιτερότητες, οι οποίες σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να ενταχθούν σε ένα πλαίσιο σκληρού ανταγωνισμού και εμέσως τελικά να καταστραφούν όλα τα θετικά των περιφερειών μας, δηλαδή το τοπικό επίπεδο και η τοπική παραγωγή. Ξεκάθαρα λοιπόν το λέω από την αρχή ότι δεν θέλω οι περιφέρειές μας να γίνουν Silicon Valley. Αυτό το οποίο όμως θα ήθελα είναι η δική μας η περιφερειακή πολιτική να επα... επαναπροσανατολίσει την πολιτική μας απέντη στις προκλήσεις τις οποίες πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Η πρώτη αυτή πρόκληση είναι το ότι ε, η Ευρώπη δεν έχει αρκετά ορυκτά καύσιμα και ουσιαστικά έχουμε ξεπεράσει πάρα πολλές φορές ακόμα και τα 100 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως κάθε φορά που πρέπει να κάνουμε εισαγωγές τέτοιων πόρων. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι ε, πλήττονται πάρα πολύ και ο τομέας των ανανεώσιμων πηγών ενέργεια, ιδίω ε, απέναντι στον έντονο αγωνισμό που υπάρχει με άλλε χώρε. Θα πρέπει, πιστεύω, να επενδύσουμε πολύ περισσότερο στη δική μα την περιφερειακή πολιτική, προκειμένου να γίνουν κάποιε επενδύσει για τι τεχνολογίε του μέλλοντο. Δεν αναφέρουμε αυτή τη στιγμή σε βιομηχανίε και επιχειρήσει οι οποίε ήταν αποδοτικέ σε δύο-τρία χρόνια, αλλά σε επιχειρήσει εκείνε οι οποίε θα πρέπει να είναι αποδοτικέ μέσα σε 10-20 χρόνια. Νομίζω ότι πραγματικά οι περιφέρειέ μας θα πρέπει να στραφούν προ τέτοιε μακροπρόθεσμε επενδύσει για να αντιμετωπίσουν προκλήσει όπω κλιματικέ αλλαγέ ή ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια. Πριν από λίγο αναφερθήκατε στον τομέα τη αυτοκινητοβιομηχανίας και είπατε ότι θα πρέπει να περάσουμε από τον κλασικό τομέα τη αυτοκινητοβιομηχανίας, ο οποίο μολύνει πολύ, προς ένα τομέα ο οποίος να έχει μειωμένε εκπομπέ διοξιδίου του άνθρακα ή να επενδύσουμε περισσότερο στα μέσα μαζική μεταφορά. Τι σημαίνουν όλα αυτά. Η περίφημη ευφύης εξειδίκευση θα πρέπει να θέσει σημαινουν ολα αυτα η περιφημη ευφυηση εξειδικευση θα πρεπει να θεσει καποιε προτεραιοτητε ω προ του καινοτόμου τομεί, Έχετε απόλυτο δίκιο προ αυτό. Πιστεύω ότι θα πρέπει να επενδύσουμε όμω προ τι οικολογικέ τεχνολογίε, οι οποίε αυτή τη στιγμή δεν βρίσκονται στα πλαίσια μια κοινή βιομηχανική πολιτική στην Ευρώπη, μόλον ότι θεωρώ ότι ακριβώ εκεί πέρα θα πρέπει να εστιαστούμε ω Ευρώπη. Θεωρώ λοιπόν ότι δεν θα δούμε ποτέ μια βιομηχανική επανάσταση αν δεν εστιαστούμε πραγματικά στους τομείς αυτούς. Η βιομηχανική επανάσταση μπορεί να συμβεί μόνο αν καταφέρουμε να θεσπίσουμε σε περιφερειακό επίπεδο μία εδαφική περιφερειακή διάγνωση βάσει των τοπικών αναγκών, των ε, αναγκών των τοπικών κοινωνιών, βάσει των θέσεων απασχόλησης που υφίστανται σε κάθε περιφέρεια. Νομίζω ότι βάσει των παραμέτρων αυτών θα πρέπει να θέσουμε μελλοντικού στόχους. Αν πρέπει σήμερα να κάνουμε μία εδαφική διάγνωση για να δούμε ακριβώς τι συμβαίνει σε κάθε περιφέρεια, ποιοι είναι οι δείκτες που θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν. Ξέρετε ότι οι αστικές περιοχές, οι υπαίθρες περιοχές και το καθεξής δεν έχουν τις ίδιες ανάγκες. Είναι πάρα πολύ σημαντικό κάθε κράτος να κάνει μία εδαφική διάγνωση, να το αποκαλέσω έτσι, προκειμένου να δει πραγματικά ποιοι είναι οι τομείς στους οποίους θα πρέπει να κάνει επενδύσεις, ποιοι είναι οι τομείς αυτοί οι οποίοι μπορούν να δημιουργήσουν θέσεις απασχόλησης. Ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Χρυσόγελος έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Είναι βέβαια μεγάλη συζήτηση για τη βιομηχανική πολιτική και εγώ θα προσπαθήσω να την εστιάσω στο θέμα της, ε, το αντικειμένου της Επιτροπής μας, δηλαδή της Περιφερειακής Ανάπτυξης Καταρχήν έχουμε δύο μοντέλα βιομηχανίας. Είναι οι παραδοσιακές βιομηχανίες που αντιμετωπίζουν μια σειρά από προβλήματα και βέβαια υπάρχει και το μοντέλο της καινοτόμου βιομηχανίας που έχει άλλες ανάγκες και απαιτήσει. Ε, και από την άλλη μεριά είναι σωστό ότι κάθε περιφέρεια πρέπει να έχει λόγο για το βιομηχανικό μοντέλο το οποίο θα ακολουθεί στην περιοχή της και να συμμετάσχει στη διαδικασία διαβούλευσης και εν ώψη του συμβολέου ή της συμφωνίας εταιρικής σχέσης θα πρέπει και στο θέμα της βιομηχανικής πολιτικής οι περιφέρειες να έχουν λόγο και να συμμετάσχουν. Γιατί και τα αποτελέσματα μέσα από μια τέτοια διαβούλευση και συμμετοχική διαδικασία θα είναι πιο καλά και για τη βιομηχανική πολιτική αλλά και για την περιφερειακή ανάπτυξη. Τώρα για το θέμα της, της παραδοσιακής βιομηχανίας. Ξέρουμε ότι υπάρχει μια μεγάλη κρίση η οποία έχει δύο ρίζες. Η μία ότι πολλές φορές αυτές οι βιομηχανίες δεν μπορούν να ανταγωνιστούν στο σύγχρονο οικονομικό περιβάλλον, δεν είναι ανταγωνιστικές από οικονομική άποψη, αλλά και πολλές φορές δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις αξίες και στις απαιτήσει περιβαλλοντικές και κοινωνικές των ε, πολιτών και πολλές από αυτές τις βιομηχανίες κλείνουν γιατί δεν μπορούν να ανταποκριθούν σε περιβαλλοντικά στάνταρτς, σε ενεργειακά στάνταρτς κλπ. Άρα θα πρέπει να υπάρχει μια μεσοπρόθεσμη στρατηγική που σε κάθε περιφέρεια θα βοηθήσει αυτές τις βιομηχανίες να μεταστραφούν, να γίνουν πιο αποδοτικές και πιο υπεύθυνε κοινωνικά και περιβαλλοντικά. Είναι κάτι διαφορετικό από την καινοτομία η οποία πρέπει να υπάρχει σε κάτι που γεννιέται καινούριο. Οι καινούριε βιομηχανίες, οι καινοτόμε βιομηχανίες πρέπει να γεφυρώσουν τον σχεδιασμό της τον οικονομικό με τις απαιτήσεις αν θέλετε και με την νομοθεσία την οποία προωθούμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και θα φέρω δύο-τρία παραδείγματα για να γίνει πιο κατανοητό. Για παράδειγμα, μιλάμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την αποτελεσματική χρήση των πρώτων υλών. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να δώσουμε μεγάλη έμφαση στην βέλτιστη χρήση πρώτων υλών στην ανακύκλωση στην επανάχρηση των πρώτων υλών και όχι τόσο στην εξορυκτική δραστηριότητα γιατί μπορούμε να έχουμε έναν άλλο μοντέλο εξορίξεων το οποίο δεν είναι πια αυτό το γνωστό που ξέρουμε που σκάβουμε τη γη, ανοίγουμε τούνελ, ανοίγουμε ορυχεία αλλά είναι μια πολιτική που ανακυκλώνει. Δηλαδή είναι προτιμότερο μια βιομηχανία που επενδύει στην ανακύκλωση των πρώτων υλών που υπάρχουν σε πολλά προϊόντα σήμερα παρά το να σκάβουμε και να καταστρέφουμε το περιβάλλον και, τους, τις πρώτες ύλες που έτσι καλλιώς δεν ανανεώσουμε στην πλειοψηφία τους. Ένας δεύτερος τομέας είναι τα πλοία θέλουμε και έχουμε αποφασίσει και ψηφίζουμε στο ευρωπαϊκό κοινοβούλιο και είναι ευρωπαϊκή πολιτική να βελτιώσουμε την περιβαλλοντική απόδοση των πλοίων να μειώσουμε τις εκπομπές να μειώσουμε την ενεργειακή κατανάλωση άρα αυτό σημαίνει ότι πρέπει να ενισχυθεί αντίστοιχα και η ναυπηγική βιομηχανία ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί στις προδιαγραφές που θέτουμε. δηλαδή καινοτόμα σε αυτή την περίπτωση θα είναι ναυπηγία και η ναυπηγική δραστηριότητα που θα μπορούσε να φτιάξει πλοία μηδενικών εκπομπών αφού θέλουμε να μειωθούν οι εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα και των άλλων ρήπων από τα πλοία σημαίνει ότι πρέπει να ενισχυθεί μια τέτοια καινοτόμα έρευνα αλλά και εφαρμογή βιομηχανική έτσι ώστε σε μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο επίπεδο να έχουμε πλοία τα οποία δεν θα έχουν εκπομπές, θα βασίζονται σε ανώσιμε πηγέ ενέργεια, θα έχουν ευέλτιστο σχεδιασμό, θα χρησιμοποιήσουν πιθανά καινοτομία και έρευνα που υπάρχει στα πανεπιστήμια σήμερα αλλά που δεν γεφυρώνεται πολύ συχνά γιατί εδώ πρέπει να, παίξει ρόλο, παίξουν ρόλο και οι περιφέρειες. Αν θέλουμε παράδειγμα πολιτική τέτοια για την αυτιλία πρέπει όσον τουλάχιστον αφορά τις συνδέσεις μεταξύ περιφερειών μεταξύ νησιών ή παράκτιες συνδέσεις οι περιφέρειες σε αυτές τις περιοχές να παίξουν ένα προθετικό ρόλο σε τέτοιες πολιτικές και να αποτελέσουν τη γέφυρα για τέτοιες δραστηριότητες. Και βέβαια σε κάθε περιοχή συμφωνώ ότι πρέπει να υπάρχει αξιοποίηση του κοινωνικού κεφαλαίου και των πλεονεκτημάτων μιας περιοχής, αλλά όχι μια εξειδίκευση η οποία μπορεί να είναι ενάντια στην συνολική ταυτότητα μιας περιφέρειας. Και σε αυτό πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Ευχαριστώ πολύ. Thank uh, Uh, <clears throat> Σας ευχαριστώ. Σύντομα, πρώτα απ' όλα ένα, μια παράκληση. Θα μπορούσαμε τα έγγραφα αυτά να τα έχουμε και σε ψηφιακή μορφή της διαφάνειας τέλο πάντων των ομιλητών. Και δεύτερον, μήπως θα έπρεπε να έχουμε και ένα ε, λεξιλόγιο με όλα αυτά τα ακρονίμια, τα αρκτικόλεξα. Δεν, δεν καταλαβαίνουμε. Θα ήταν καλό να έχει η Επιτροπή μας ε, ένα κατάλογο. Εγώ άντε να γνωρίζω δύο στα πόσα, δύο, τρία. Δεν τα καταλαβαίνω τα άλλα. Και πώς να καταλάβω και τι λέτε λοιπόν άμα δεν τα γνωρίζω. Όταν συζητάμε λοιπόν ιδίω για ευφυή e, εξειδίκευση, είναι πολύ ενδιαφέρον το διάγραμμα γιατί είναι όλα αρχικά και δεν καταλαβαίνουμε τίποτα. Τέλος πάντων, το τρίτο στοιχείο. Υπάρχει κίνδυνος. Η ευφυής εξειδίκευση όπως και η ευφυής πόλης από τη μια πλευρά ναι μεν να έχουμε ενδιαφέρουσες αναλύσεις, εξελίξεις, εκθέσεις, οσά λοιπά... που δείχνουν ε, την ιδιαιτερότητα της νέας προσέγγισης. Από την άλλη όμω πλευρά, να λέμε ότι καλό είναι απλά καλά διαχειριζόμενο. Δηλαδή ευφυα σημαίνει καλή διαχείριση. Φυσικά πρέπει να προσαρμοστούμε στο νέο περιβάλλον, στην αλλαγή των νέων τεχνολογιών, αλλά το ερώτημα είναι αν υπάρχει καλή ή κακή διαχείριση. Και πολύ συχνά στην, στη δημόσια συζήτηση βλέπουμε ότι FES σημαίνει καλό, πολύ απλά. Αυτό που χρειάζεται λοιπόν να δείξουμε είναι την πραγματική διαφορά που υπάρχει στον τρόπο σκέψης και στην ε, κατάρτιση αυτών των σχεδίων εφίους εξειδικευσή. Υπάρχει αυτή η πλατφόρμα από την κατάλαβα εφίους εξειδικευσή. Τι χρειάζεται όμω, πρέπει να δοθεί μια σαφή εξήγηση. Γιατί εμεί είμαστε νομοθέτε. Μπορεί οι, οι επιχειρήσει συγγνώμη, να το καταλαβαίνουν, αλλά πρέπει να το καταλαβαίνουν και οι περιφέρειε, αλλά και εμεί. Πώ εμεί μπορούμε λοιπόν να το μεταφράσουμε σε ένα νομικό κείμενο. Είμαι εισηγητή ε, για το Ταμείο, το ΕΤΠΑ. Ε, και επειδή πολλές φορές έχω ακούσει ένα λόγος για θέλω να σας ρωτήσω, πού υπάρχει στην νομοθεσία, πού θα μπει, σε κάποια εκτελεστική πράξη, δεν το έχω δει πουθενά μέχρι τώρα. Είναι απλά, όπως είπα και το πρωί νωρίτερα, μία πρόταση, μία πλατφόρμα, μία κατευθυντήρια γραμμή, ο πρώτος πυλώνας, ε, smart, εφής. Θέλουμε να έχουμε συγκεκριμένα πράγματα, απτά. Καταλαβαίνω την ιδέα αλλά υπάρχει κάποια προσπάθεια αυτό να μεταφραστεί σε ένα συγκεκριμένο νομικό κείμενο χειροπιαστό και θα έχει κάποια στοιχεία υποχρεωτικά, υποχρεώσει κτλ. κτλ. Γιατί εντάξει καλέ είναι οι πλατφόρμες και οι ανταλλαγέ εμπειριών, αλλά έχουμε αρκετέ Και σε ό,τι αφορά αυτή την ε, διοργανική, διπηρεσιακή ε, διαδικασία για τις ευφύς πόλεις και αυτή η διαβούλευση που θα γίνει, τι αποτέλεσμα θα έχει για τη νέα περίοδο προγραμματισμού. Δεν ξέρω, μπορεί να λέω τετριμένα πράγματα, αλλά θα μπορούσα να ξέρω πού υπάρχουν όλα αυτά στα νομικά κείμενα. Ναι, παρακαλώ. Κύριος Μάνκα. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αρχικά δεν ήθελα να ζητήσω τον λόγο να παρέμβω, Πρόεδρε, αλλά η παρουσίαση με οδήγησε, με όθησε να παρέμβω. Το 1999, όταν ήμουν δήμαρχος στη χώρα μου, προσπάθησα τότε τα πανεπιστήμια σε όλες τους τις δραστηριότητες της ζωής της πόλης μας να τα εντάξω σε αυτές τις δραστηριότητες και στο σχεδιασμό και προγραμματισμό. Τα επιμέρους πανεπιστήμια δεν ήθελαν να το κάνουν αυτό. Είχαν όμως πάρα πολλές γνώσεις ε, και πραγματογνωμοσύνη. Δεν ήθελαν όμως να κάνουν αυτό, να τολμήσουν αυτό το πρώτο βήμα, αυτή την προώθηση. Χρειαζόντουσαν κάποιον που θα τους έλεγε χρειαζόμαστε ένα βαθμό διαχείρισης και θέλουμε να σας εντάξουμε στην περιφέρειά μας ένα συγκεκριμένο βαθμό στο έργο μας. Οι στρατηγικές που παρουσιάζονται σήμερα δεν είναι μόνο κάτι εποφελές για την οικονομία αλλά και για την περιφερειακή πολιτική και περιφερειακή ανάπτυξη. Τίθεται το ερώτημα τώρα. Πώς μπορούμε αυτές τις αναλύσεις να τις χρησιμοποιήσουμε θετικά στην πρακτική τους εφαρμογή. Διότι αν οι στρατηγικές και οι αναλύσεις μόνο από ένα στενό κύκλο προνομιούχων μπορούν να ε, οδηγήσουν σε κάποιο αποτέλεσμα δεν έχουν όφελο. Πρέπει να δούμε πώ αυτέ οι αναλύσει μπορούν να βοηθήσουν την περιφέρεια περαιτέρω και να καταδείξουν πώ μπορούν τα πράγματα να εξελιχθούν θετικότερα. Έχω αμφιβολίε αν οι περιφέρειε μπορούν και με ποιο τρόπο μπορούν να συμμετάσχουν. Ερωτώ, ερωτώ λοιπόν τι μπορούν να κάνουν οι περιφέρειε. Η απάντηση είναι αυτό το οποίο χρειάζονται είναι η απάντηση. Ευχαριστώ. Grazie Presidente. Io ho apprezzato Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εκτιμώ ιδιαίτερα τη μελέτη η οποία μας παρουσιάστηκε και θεωρώ ότι πραγματικά εντάσσεται πάρα πολύ καλά στο πλαίσιο του φακέλου που εξετάζουμε. Ωστόσο, υπάρχουν κάποια όρια και αυτά τα βλέπουμε στις υπερβολικές θεωρητικές προσεγγίσεις που γίνονται στις μελέτες αυτές. Δεν ακούσαμε πάρα πολλά πράγματα συγκεκριμένα. Θα πρέπει όλα να τα θέσουμε στο σωστό τους πλαίσιο και ιδίω στην τρέχουσα συγκυρία. Αυτή τη στιγμή επεξεργαζόμαστε κάποιους κανονισμούς οι οποίοι θα πρέπει ουσιαστικά να συνδέονται με τις μελέτες αυτές οι οποίες μας παρουσιάστηκαν. Διαφορετικά, δεν νομίζω ότι θα καταφέρουμε να κάνουμε κάτι ουσιαστικό. Όταν θα ολοκληρώσουμε εμεί τη δική μα μελέτη, ήδη τα αποτελέσματά μα θα είναι πεπερασμένα και τελικά θα παραμείνουν θεωρητικά. Πρώτον αυτόν. Δεύτερον, όπω είπε και ο κύριο Βανίστερόι, θεωρώ ότι θα πρέπει να αρχίσουμε σιγά σιγά να εξετάσουμε πολύ περισσότερο την πραγματικότητα κάποιων μεμονωμένων περιφερειών στην Ευρώπη, γιατί τι αντιμετωπίζουμε πολύ γενικά και σφαιρικά αυτή τη στιγμή. Να δούμε πώς αυτή η ευφυή εξειδίκευση μπορεί να εφαρμοστεί στην πράξη σε ξεχωριστέ περιφέρειες. Με άλλα λόγια, πιστεύω ότι θα πρέπει πραγματικά να ασχοληθούμε περισσότερο με το ζήτημα αυτό και θα πρέπει όλα αυτά τα σημαντικά πορίσματα της μελέτης να χρησιμοποιηθούν ουσιαστικά για τη μελλοντική μας νομοθετική εργασία. Σας ευχαριστώ. Ε, thank you. Πρόεδρος, σας ευχαριστούμε. Πρωτού δώσω το λόγο στους εμπειρογνώμονες, θα ήθελα και εγώ να πω ότι ένα πρώτο συμπέρασμα της σημερινής συζήτησης είναι ότι τελικά χρειαζόμαστε μία ακόμα συνάντηση προκειμένου να συζητήσουμε περισσότερο τα ζητήματα της ευφύης εξειδίκευσης, πράγμα το οποίο πρότεινε και εκπρόσωπος Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Να δούμε πώς θα καταφέρουμε να βοηθήσουμε τις περιφέρειες ε, να χρησιμοποιήσουν τη νέα αυτή διαδικασία που προβλέπεται στην προτινόμενη βιομηχανική πολιτική, ιδίως όσον αφορά τον στόχο της ευφύους ε, εξειδίκευσης. Επίσης θα ήθελα να γνωρίζω ποια είναι η άποψη της DG Regio ή μάλλον τι κάνει η DG Regio προκειμένου να προετοιμαστούν οι περιφέρειες για τη νέα αυτή πολιτική και για να τονιστεί στις περιφέρειες ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό το ζήτημα της ευφύους εξειδίκευσης και της καινοτομίας. Τα όσα κάνετε πιστεύω ότι αντιστοιχούν τελικά στη δημιουργία ενός συστήματος ή ουσιαστικά θέλετε να δημιουργήσετε μία υψηλότερη, καλύτερη δυνατότητα, ικανότητα των περιφερειών για να ανταποκριθούν στην παγκόσμια οικονομική συγκυρία. Πιέστε δηλαδή κατά κάποιο τρόπο τις περιφέρειες να ανταποκριθούν στις νέες προκλήσεις καινοτομία και τεχνολογίας προκειμένου να καταφέρουν να είναι λίγο πιο ανταγωνιστικές σε διεθνές, σε παγκόσμιο επίπεδο. Μήπως θα πρέπει δηλαδή να αναθεωρήσει η Ευρώπη τη δυνατότητά της στην καινοτομική προκειμένου να καταφέρει να γίνει λίγο πιο ανταγωνιστική σε παγκόσμιο επίπεδο. Θέλετε ουσιαστικά μέσω της περιφερειακής πολιτικής να δημιουργήσετε μεγαλύτερη ανταγωνιστικότητα στις περιφέρειες, προκειμένου αυτές να απτυχθούν περισσότερο και να δημιουργήσουν περαιτέρω θέσεις εργασίας και να αντιμετωπίσουν κατ' επέκταση τα κοινωνικά τους προβλήματα. Θεωρώ ότι αυτό αποτελεί μια τεράστια πρόκληση για την Ευρώπη. Και συνειδητοποιώ ότι έχει ξεκινήσει μια νέα συζήτηση για τη βιομηχανική πολιτική, στα πλαίσια της οποίας η περιφερειακή πολιτική θα πρέπει να δει πώς μπορεί να συμβάλλει στην εκπόνηση αυτής της νέας βιομηχανικής πολιτικής, προκειμένου πραγματικά να ακολουθήσει η βιομηχανική πολιτική ένα σωστό δρόμο και να καταφέρουν τελικά και οι περιφέρειες να συμβάλλουν σε αυτή τη νέα βιομηχανική πολιτική. Είμαι ιδιαίτερα ευγνώμων λοιπόν προς τον κύριο Γκάιλ, ο οποίος αναφέρθηκε σε αυτή την διάσταση πολύ συχνά δεν συζητάμε την συνεισφορά των περιφερειών στη βιομηχανική πολιτική. Χαίρομαι λοιπόν πάρα πολύ που εξετάστε εσείς το ζήτημα από την οπτική αυτή γωνία. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να δούμε πραγματικά ποιες είναι οι κοινωνικές, πολιτισμικές, τεχνολογικές ή γνωστικές δυνατότητες των περιφερειών και πώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν αυτές προκειμένου να συμβάλλουν οι περιφέρειες στη βιομηχανική πολιτική. Όπως είπαν όμως και οι συνάδελφοι, βρισκόμαστε στην αρχή μόνο της συζήτησης. Θα πρέπει να συνεχίσουμε τη μελέτη του ζητήματος αυτού. Και θα ήθελα να σας ζητήσω να απαντήσετε κυρίως στο ερώτημα του κυρίου Όλμπριχτ. Δηλαδή, σε ποιο βαθμό χρειαζόμαστε ένα νομικό πλαίσιο ή σε ποιο βαθμό τελικά αναφερόμαστε σε κάποιες διαδικασίε οι οποίες δεν απαιτούν νομικές διατάξεις στα πλαίσια της πολιτικής. Βρισκόμαστε μέσω των διαπραγματεύσεων και αν πραγματικά πιστεύετε εσείς ότι ε, θα πρέπει να δημιουργηθεί ένα νομικό πλαίσιο και ότι θα πρέπει να συμβάλλει σε αυτό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τότε ενδεχομένω να υπάρχει ακόμα χρόνο για να γίνει κάτι τέτοιο. Αλλά από ό,τι κατάλαβε η προσέγγιση Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι διαφορετική, ότι δεν χρειάζεται ένα νομικό πλαίσιο. Ότι μπορούν δηλαδή οι περιφέρειε να αναλάβουν δράση και πρωτοβουλίε στα πλαίσια τη εφιστάμενη βιομηχανική πολιτική. Ενδεχομένω ο ίδιο επίτροπο θα μπορούσε να μα απαντήσει στο ζήτημα αυτό και όχι οι σημερινοί συμμετέχοντε. Κλάου, έχει το λόγο και συνέχεια και ο Κρίστιαν μπορεί να συμπληρώσει εφόσον το επιθυμεί. Uh, Ευχαριστώ πολύ. Φυσικά και ο Κριστιαν θα απαντήσει και αυτό. Σε αυτό το αμικό πλαίσιο δεν είμαι βέβαια, όπω καταλαβαίνετε, σε θέση να απαντήσω εξ ονόματο ε, ολόκληρη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά εκτιμώ τι προσπάθειε που κάνετε για να διευκρινιστούν όλα αυτά τα ζητήματα. Και επειδή εγώ προσωπικά ασχολούμαι με την πρόθεση και την ανάπτυξη τη ε, φιού εξειδίκευση, ε, μπορώ να πω ότι υπάρχουν δύο στοιχεία τα οποία θέξατε κι εσεί. Πρώτον, και κάτι που είναι καινούριο, το να καταστεί υποχρεωτικό να ακολουθεί κανείς μια αυστηρή μεθοδολογία και όχι απλά να λέει ότι ναι, ξέρετε, κάναμε ανάλυση SWOT, και ορίστε τα πορίσματα. Και αυτό θα πρέπει να χρηματοδοτήσετε. Επομένως υπογράψτε τα επιχειρησιακά προγράμματα και ορίστε και οι δαπάνε για τα επόμενα 7 χρόνια. Υπάρχει και κάτι που λέγεται capacity building, δημιουργία υποδομών. Επειδή πλέον έχουμε αυτή την αιρεσιμότητα, το conditionality και οι περιφέρειες θέλουν να είναι καλοί μαθητές και να πληρώνουν τους όρους και τις προϋποθέσεις για να μπορέσουν να έχουν τις, ε, τη χρηματοδότηση και να δαπανούν πόρους. στο CSF, τον Γενικό Κανονισμό, στο Στρατηγικό Πλαίσιο, στο παράρτημα, έχουμε συγκεκριμένες ε, ε, συγκεκριμένα κριτήρια, τα οποία δεν χρειάζεται να σας τα αναγνώσω. Περιορισμένες είναι αυτές οι κατευθυντήριες γραμμές, αλλά πέραν αυτών που ορίζονται σε αυτό το παράρτημα, έχουμε αρχίσει να εκδίδουμε κατευθυντήριες γραμμές πολιτικής, policy guidelines και εργαζόμαστε με πάρα πολλές περιφέρειες ε, που φτιάχνουν μαζί με άλλες περιφέρειες τις λεγόμενες peer reviews, ε, τις αναθεωρήσεις, ε, εκτιμήσεις από ομοτήμους. Για να δουν, τα κάναμε καλά, μπορούσαμε να κάνουμε κάτι καλύτερο κτλ. Και έτσι μπορούν να αξιοποιήσουν καλύτερα και τα κονδύλια. Άρα υπερβαίνουν τις νομικές υποχρεώσεις πολλές φορές, τις στενές αυτές. Υπάρχουν πολλές περιφέρειες, μπορώ να σας πω, που ούτε καν είναι ακόμη καταχωρισμένες στην πλατφόρμα, αλλά τελικά εξετάζουν το παρελθόν, τι έχουν γίνει, τι έχει γίνει κατά το παρελθόν στον τομέα των στρατικών καινοτομία. Και όλα αυτά τα συγκρίνουν με τι κατευθυντήριε γραμμέ. Και επαναλαμβάνω, του βοηθούν κορυφαίοι εμπειρογνώμονε. Και έτσι ευθυγραμμίζονται για να, με τι βέλτιστε πρακτικέ. Γιατί αλλιώ, και θα σα δώσω ένα υποθετικό εντελώ σενάριο. Ξέρετε, κάποιε περιφέρειε μπορεί να μην είναι σε θέση να δαπανίσουν τα κονδύλια τα οποία λαμβάνουν ε, για την καινοτομία με σόφρονα τρόπο. Μπορεί δηλαδή να κάθονται σε μια επιτροπή προγραμματισμού και να τι κάνουμε τώρα με αυτά τα κονδύλια που πήραμε για την καινοτομία και μετά έρχονται τα πανεπιστήμια και του λένε Ξέρετε, εμεί χρειαζόμαστε μια μηχανή για να βρούμε την ε, ακολουθία του DNA και δεν ξέρω εγώ πόσε χιλιάδε ευρώ τελικά ε, μπορεί κάποιος να παίρνει χρήματα ε, είναι σαν να έχουμε τη Φεράρι μέσα στον Καράζ. και μοιράζονται τα χρήματα και δεν γίνεται τίποτα. Υποθετικό παράδειγμα αυτό με την Ελλάδα. Τέλο πάντων, το θέμα είναι να υπάρχει μια στρατηγική. Να υπάρξει συμφωνία με του εμπλεκομένου φορεί. Ο Κρίστιαν, φαντάζομαι, θα θίξει την ουσία όλων αυτών των ζητημάτων τη κολλική καινοτομία, τη διακυβέρνηση. Όλα αυτά τα βλέπουμε, είναι καινούρια. Βλέπουμε να κινείται κάτι πάντω. Και θα σα ήμασταν ευγνώμονε αν συνεχίσετε να συζητάτε μαζί μα, ε, να μα ε, θέτετε τι απορίε και τι αμφιβολίε σα, γιατί αξίζει να τα συζητήσουμε όλα αυτά. Ο Κρίστιαν. Κάποια άλλα επιπλέον σχόλια. Αυτή η διαδικασία άλλαξε πολλές νοοτροπίες και απόψεις στις περιφέρειες. Έχω ταξιδέψει παντού και πολλοί και γνωρίζουν οι εμπλεκόμενοι αυτές τις διεργασίες. Είναι μια πολυσχηδή διεργασία για να απαντήσω. Ναι, υπάρχει μια τοπική διάγνωση της περιφέρειας και σε σχέση με τις δυνατότητες καινοτομία που μπορούν να αναλυθούν κτλ. Υπάρχει μια διαδικασία διακυβέρνησης, διαχείρισης που περιγράφεται με ε, περιεκτικό τρόπο για να εντοπιστούν για τους ενδιαφερόμενους οι μοναδικές ευκαιρίες που προσφέρονται ανάλογα με κάθε περιφέρεια. Παρ' όλα αυτά έχουν και ένα περιθώριο ελευθερίας οι περιφέρειες να δράσουν και έχουμε κάποια τέτοια παραδείγματα. Δεν θα κατονομάσω περιφέρειες αλλά μπορεί να σας ε, κάνει να στοχαστείτε αυτό σχετικά. Ζήτησαν λοιπόν από καθηγητές ε, πανεπιστημίου να κάνουν μια τέτοια ανάλυση και να ληφθεί απόφαση για το τι είναι σημαντικό από πλευράς τους. Μια άλλη δυνατότητα, πραγματογνώμονες, να συντάξουν μέχρι 10 προτεραιότητες και να εγκριθούν κάποιες από αυτές ώστε να ευθυγραμμίζονται και να συμμορφώνονται με τις διατάξεις του κανονισμού. Μετά έχουμε περιφέρειες που πραγματικά διαδραματίζουν τον ρόλο της δημιουργίας συναντήσεων, συνειδητοποίησης και ευαισθητοποίησης στις ιστοσελίδες, στο διαδίκτυο και εδώ και σε σχέση και με τις ίδιες ε, τις ε, αρχές και τους συμβούλους Όλα αυτά μπορούν να συνεισφέρουν να διατυπωθούν ε, οι προτάσεις για περί του πρακτέου. Και ένα τέταρτο πρότυπο μία εκ παραλίλου άτυπη ε, διαδικασία διαχείρισης και ένα σε πιο τυπικό επίσημο επίπεδο που εμπλέκει και τους πολίτες που είναι οι ε, εκφραστές σε αυτό το επίπεδο και οι προ... Ε, εκείνοι που πρέπει να ε, επιλέγουν. Τώρα, το θέμα είναι το πώς θα μπορέσουν όλα αυτά να καταλήξουν στα έγγραφα και στις προτάσεις. Ποιος όμως θα ελέγχει την υλοποίηση όλων αυτών. Ποιος θα είναι ο επόπτης. Αυτό είναι το κέρια σημασία ε, θέμα. Το επόμενο βήμα είναι η ανάλυση και αξιολόγηση. Ποιος θα ελέγχει λοιπόν όλα αυτά. Ποιος θα είναι ο ελεγκτής. Το ελεγκτικό συνέδριο μήπως. η Γενική Διεύθυνση Περιφερειών ε, Regio, DG ε, Regio στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή η Γενική Διεύθυνση ε, Έρευνας DG Research ή ποιος. Και όταν λέω υλοποίηση, εφαρμογή είναι αυτό το οποίο αναφέρεται με μείγμα πολιτικής, policy mix θα πρέπει να δούμε την κατηγοριοποίηση, ομαδοποίηση, clusters. Αυτό είναι ένα κύριο θέμα σήμερα. Αν δεν επιλέξουμε αυτό, αν δεν επιλέξουμε επενδύσεις σε όλα αυτά, τότε δεν μπορούμε να κατηγορήσουμε κανέναν ότι είναι υπεύθυνο για μια τέτοια κατάσταση. Εμείς θα είμαστε υπεύθυνοι. Περί αυτού πρόκειται. Και παραπάνω απ' όλα χρειάζεται να πείσουμε τις περιφέρειες να επενδύσουν σε αυτό που αποκαλούμε περιφερειακή ευφυΐα, regional intelligence, γιατί τι γίνεται. Γίνονται αναλύσεις, ε, έχουμε ένα διάστημα εξαετές. Ε, πρέπει να μπορέσουμε μέσα σε αυτά τα έξι χρόνια να κάνουμε κάτι. Κανείς όμως ε, δεν βλέπει τι γίνεται, τι έχει αλλάξει, ποια είναι η νέα κατάσταση για τις περιφέρειες. Αυτά πρέπει να αναλυθούν και να αξιολογηθούν και για τη διαφοροποίηση μεταξύ παραδοσιακής και καινοτόμου βιομηχανίας ακόμα και για τις ε, παραδοσιακές βιομηχανίες ε, πρέπει να καινοτομήσουν. Ή θα καινοτομήσουν ή θα αποβιώσουν, θα πεθάνουν. Δεν είναι τώρα ε, το θέμα επιλογής ενός επαΐοντος για κάποια περιφέρεια. Για παράδειγμα, για το, τα θέματα τουρισμού π.χ. Αν δεν καινοτομήσουν και αυτές οι περιφέρειες θα αποτύχουν. Και για να επανέλθω σε κάποιον που ανέφερε το θέμα, που ανέφερε το θέμα της διαχείρισης, ενεργειακής διαχείρισης έχει ξεκινήσει για παράδειγμα ένα πιλωτικό σχέδιο με κάποιο ξενοδοχείο μπόρεσαν να περικόψουν το κόστος κατά 12% μόνο με τη διαχείριση των πόρων ε, όσον αφορά το νερό και, την, ε, ε, και την ηλεκτρική, το ηλεκτρικό ρεύμα. Βλέπετε λοιπόν πολλά μπορούν να γίνουν. Και ένα άλλο σημαντικό θέμα να υπάρξει ένα κλάστερ, μια ομαδοποίηση ώστε να μπορεί ο τοπικός παραγωγός να μπορεί να, παρέχει, να παράσχει τα προϊόντα του αυτά σε κάποιον που βρίσκεται κοντά π.χ. σε ένα ε, ξενοδοχείο ή κάτι συναφές. Υπάρχει λοιπόν και η πτυχή της καινοτομίας. Δεν είναι η, τεχνολογία της, ε, η καινοτομία στην τεχνολογία, είναι καινοτομία στις υπηρεσίες για παράδειγμα, στην παροχή υπηρεσιών. Εκεί πρέπει να θέσουμε κέντρο βάρους περισσότερο από στο παρελθόν για παράδειγμα. Σας ευχαριστώ κύριος Γκάιερ θα ήθελε να σχολιάσει. Καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Σούλτσε και τους άλλους που συμμετείχαν ως ε, πραγματογνώμονες στις εκθέσεις που μας εξέθεσαν, στις παρουσιάσεις. Ε, συμμετείχαν και με ρίμνησαν για μια ενδιαφέρουσα συζήτηση και ευχαριστώ και τους συναδέφους για τις ε, παρατηρήσεις τους. Έχουμε το πρόβλημα, δεν μπορούμε πραγματικά να φανταστούμε πώς αυτές οι στρατηγικές στις περιφέρειές μας, στις χώρες μας θα μπορέσουν να λειτουργήσουν χειρόπιαστα. Εμείς όμως ε, οι δυστυχείς ε, αρμόδιοι για την πολιτική και την ανάπτυξη αυτών των περιφερειών τώρα σε σχέση με τον κύριο Όλμπριχ σε δύο κατηγορίες για παράδειγμα. Πρώτον, τι μπορούμε να κάνουμε. Αυτό πρέπει να δούμε. Και είτε λοιπόν θα εφαρμοστεί η νομοθεσία, είτε θα έχουμε κάποια προγράμματα τα οποία ε, θα πρέπει, αν δεν ευθυγραμμίζονται, να ε, απαλληφθούν. Αρχίζω και προβληματίζομαι. Πού τώρα είναι η δική μας δουλειά ως Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης. Να ενταχθούμε σε τι, σε αυτά που μας περιγράψατε, σε συγκεκριμένες πολιτικές που πρέπει να διαμορφωθούν και να εφαρμοστούν. Πρέπει κάπως να στοχαστούμε και να προβληματιστούμε όμως πρώτα για όλα αυτά. Να δούμε τι μπορεί να γίνει και να ενασχοληθούμε περισσότερο με αυτό το θέμα. Είναι αναγκαίο να γίνει αυτό. Η κυρία Πρόεδρος Χούμπνερ με τα όσα ανέφερε προς αυτή την κατεύθυνση στοχεύει. Θα έλεγα λοιπόν καταρχήν ή θα πρότεινα, θα πρότεινα στα μέλη της κοινοβουλευτική μας επιτροπής αυτό το θεματολογικό πλέγμα, αυτό το, τη στρατηγική μιας ευφυούς εξειδίκευσης smart specialization για τις περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να δούμε πώς μπορεί να διαμορφωθεί εξειδικευμένα για κάθε περιφέρεια ξεχωριστά. Γιατί το λέω αυτό. Διότι το σημείο κίνησής μου ήταν να σκεφτούμε τις ιδιομορφίες, ε, τα ξεχωριστά χαρακτηριστικά βιομηχανιών, βιομηχανικών, βιομηχανικών περιφερειών, για παράδειγμα των κοινοτήτων και ε, περιφερειών άνθρακα και σιδηρουργίας και χαλιβουργίας και να δούμε τις περιφερειακές εξειδικεύσεις εξειδικευμένες στρατηγικές που θα μπορούσαν να ακολουθηθούν. Δεν πρόκειται για κάποιο ε, ας το πω έτσι παρεκκλίνον πρότυπο αυτό. Αν δούμε τις περιφέρειες Ευρώπης που αρχικά ε, προανέφερα δεν βρισκόντουσαν σε ένα τέτοιο δίκτυο. Όλα αυτά μπορούν να αλλάξουν βέβαια στο μέλλον. Αλλά από τη συζήτηση συνάγω το συμπέρασμα ότι θα πρέπει να προσπαθήσουμε στην έκθεση ιδίας πρωτοβουλίας που έχω εγώ ε, με την ευθύνη μου να προβληματιστώ να δω πώς αυτή η στρατηγική ευφυούς εξειδίκευσης smart specialization μπορεί να διαμορφωθεί και να πάρει σάρκα και οστά σε αυτές τις περιφέρειες και να δούμε τι αυτό συνεπάγεται για την περιφερειακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τα μέσα και τα εργαλεία τους. Κατανομή δηλαδή επιμερισμό κονδυλίων ή νομοθετικό έργο τι σημαίνει για όλα αυτά συγκεκριμένα. Όχι σήμερα να τα κάνουμε όλα αυτά γιατί βρισκόμαστε υπό πίεση χρόνου. Αλλά θα έλεγα αυτή είναι η επισήμανση προ του συναδέφους και θα ήμουν ευγνώμων για τι παρατηρήσει των συναδέφων και προτάσει και των πραγματογνωμόνων τι μπορούμε να κάνουμε στο μέλλον διότι δεν το έχω κατανοήσει απόλυτα, δεν το έχω αφομοιώσει και χωνέψει απόλυτα. Να δούμε με αυτή τη στρατηγική, με τι περιφέρειες, τι μπορούμε ακριβώ να κάνουμε με τι συγκεκριμένε ανάγκε και ιδιομορφίε αυτών των περιφερειών. Τι μπορούμε να κάνουμε. Προτείνει μεθοδολογικά μια μέθοδο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Καλό αυτό. Θεωρητικά μια τέτοια μέθοδος μπορεί να προέρχεται και από think tanks, από δεξαμενές προβληματισμού ή από πανεπιστήμια και πάλι για τη διαμόρφωση τώρα μιας τελικής πολιτικής. Πώς μπορούν όλα αυτά να διαμορφώσουν μια τέτοια πολιτική τελικά. Δεν το έχω κατανοήσει απόλυτα. Πρέπει να προβληματιστούμε και να δούμε και αποκινούμε άλλους πραγματογνώμονες σε σχέση με το Ευρωκοινοβούλιο να δούμε τι μπορεί να γίνει. Ευχαριστώ. Θα περιμένουμε από τον εισηγητή να μας στείλει ένα έγγραφο εργασίας, ελπίζουμε για την επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής μας και έτσι ολοκληρώνω αυτό το σημείο και δίνω και την Προεδρία στον Μάρκους Βίμπερ. Thank you very much. Okay, dann haben wir then... Εντάξει, λοιπόν πρώτα απ' όλα Έχουμε μια παρέμβαση για την ημερήσια διάταξη επί του κανονισμού. Παρακαλώ, έχετε τον λόγο εσείς. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, για την ημερήσια διάταξη. Θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή ξεπεράσαμε λίγο το χρόνο που προβλεπόταν σε σχέση με το αρχικό χρονοδιάγραμμα. Εγώ ουσιαστικά θα ήθελα να αντικαταστήσω τον κύριο Τόρεγερ για όσον αφορά την έκθεση για τις φιλευθέρους που έχει να κάνει με την απαλλαγή 2011, γενικό προπολογισμό. Δεν ξέρω αν θα μπορούσαμε να αντιστρέψουμε την ημερήσια διάταξη, γιατί εγώ πρέπει να αποχωρήσω, έχω και κάποιε άλλε υποχρεώσει. Αν γίνεται να αντιμετωπίσουμε πρώτα λοιπόν το σημείο 7. Νομίζω ότι και ο εισηγητή άλλωστε πρέπει να είναι παρόν, επομένω δεν υπάρχει πρόβλημα. Ich verstehe Ihr Anliegen. Κατανοώ το ετοιμά σα βέβαια. Το κατανοώ και ο κύριο Όλμπριχτ θα ε, μπορούσε να είναι παρόν. Αλλά για την επόμενη έκθεση ο εισηγητή και οι άλλοι σκιώδει εισηγητέ είναι παρόντε και έχουν προετοιμαστεί και έτσι μπορούμε να προχωρήσουμε. Πρέπει δυστυχώ να ακολουθήσουμε τη σειρά, να τα πάρουμε με τη σειρά. Ένα προ ένα, όπω τα προβλέπει η ημερήσια διάταξη. Δυστυχώ δεν έχουμε κάποια άλλη δυνατότητα. Και εγώ θα το ευχόμουν αυτό. Και εγώ για, αυτό, για τον κύριο Όλμπριχτ θα είχα αρκετά πράγματα να πω για αυτή την έκθεση. Όμως και οι άλλοι νομιμοποιούνται, μια και η ημερήσια διάταξη προβλέπει τη συνέχιση με τα άλλα σημεία. Θα προχωρήσουμε με τα επόμενα σημεία. Η έκθεση Όλμπριχτ είναι η, η πρώτη. Μετά την Ιρλανδική Προεδρία θα έχουμε τον Γιάνν Όλμπριχτ που θα παρέμβει. Εντάξει, ωραία. Πολύ ωραία. Περνάω τώρα λοιπόν στο σημείο 6 της ημερησίας διάταξης. Εσείς παρακαλώ, δεν το κατανόησα τι είπατε. Πριν από τη δική μου έκθεση ή το απόγευμα μετά την Ιρλανδική Προεδρία. Δεν το κατάλαβα αυτό πιο πριν. Αμέσως μετά την Ιρλανδική Προεδρία, το απόγευμα λοιπόν, η δική σας σειρά, Όλμπριχτ. Εντάξει, πολύ καλά. Λοιπόν, περνάμε καταρχήν πρώτα στο σημείο 6 της ημερήσιας διάταξης, Ταμείο Ενίσχυσης Απόρων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο κύριος Ομάτζη έχει τον λόγο, παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ. Καθυστερήσαμε λίγο με την ημερήσια διάταξη. Ωστόσο, θα ήθελα με τη δική σας την άδεια να αφιερώσουμε τον απαραίτητο χρόνο προκειμένου να μιλήσουμε για τον κανονισμό αυτό, ο οποίος είναι πολύ σημαντικός για τη δική μας την Επιτροπή. Η Επιτροπή μας θα πρέπει να εκφράσει μια γνωμοδότηση για τον κανονισμό αυτό για τη θέσπιση Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους. Πρόκειται για έναν καονισμό ο οποίος θα αντικαταστήσει τελικά το πρόγραμμα επισητιστικής βοήθειας για τους απόρους. Συζητήσαμε πάρα πολύ το ζήτημα αυτό στο τέλος του 2012, μετά από την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου της 13ης Απριλίου του 2011, που ουσιαστικά απειλούσε με εξαφάνιση το πρόγραμμα αυτό. Ενδεχομένω να θυμούνται οι συνάδελφοι ότι έγινε μία συζήτηση στην Ολομέλεια και η πλειοψηφία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ήταν σαφής. Οι περισσότεροι ευρωβουλευτές είπαν ότι το πρόγραμμα αυτό θα έπρεπε να συνεχιστεί, καταρχάς πέρα από το 2013, και κυρίως θα έπρεπε να συνεχιστεί χωρίς χρονικό όριο. Οι συζητήσεις στην Ολομέλεια επίσης αναφέρθηκαν στην αγανάκτηση που αισθανόντουσαν οι περισσότεροι ευρωβουλευτές, οι οποίοι συνειδητοποίησαν ότι δεν ήταν δυνατό στο πλαίσιο της υφιστάμενης οικονομικής κρίσης, η οποία, ας μην το ξεχνάμε, αφήνει πλέον όλο και περισσότερους ε, Ευρωπαίους σε κατάσταση ένδυας, ότι δεν θα ήταν δυνατό λοιπόν σε μια τέτοια οικονομική συγκυρία να προταθεί ποτέ μια κατάργηση του προγράμματος αυτού. Και εγώ ίδιος είχα πει ότι ήταν πραγματικά επέσχυντο να απειλούμε το πρόγραμμα αυτό με εξαφάνιση, ενώ υπάρχουν ε, χιλιάδες ευρώ τα οποία δίνονται στις τράπεζες. Δισεκατομμύρια, με συγχωρείτε, ευρώ τα οποία δίνονται στις τράπεζες. Νομίζω λοιπόν ότι ε, είναι πάρα πολύ σημαντικό να τονίσουμε το πρόγραμμα αυτό, τη σημασία του προγράμματος αυτού, καθώς επίσης και το ότι ε, υπάρχουν πάρα πολλά κράτη-μέλη που ζήτησαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εκπονήσει ένα νέο πρόγραμμα το οποίο να λαμβάνει υπόψη του και την απόφαση του Απριλίου του 2011 του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Για να καταλάβουμε όμως την απόφαση αυτή θα πρέπει να σας υπενθυμίσω ότι το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα προς τους Απόρους δημιουργήθηκε το 1987 στα πλαίσια της κοινή γεωργικής πολιτικής. Το διευκρινίζω αυτό γιατί ακριβώς επειδή πρόκειται για την κοινή γεωργική πολιτική η οποία πλαισίωνε το πρόγραμμα αυτό, γι' αυτό το λόγο δημιουργόντουσαν κάποια προβλήματα για ορισμένα κράτη-μέλη, ιδίως για τη Γερμανία, η οποία έκανε την προσφυγή αυτή ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Για ποιο λόγο το πρόγραμμα αυτό εντασσόταν στην κοινή γεωργική πολιτική. Εξ αρχής ήταν ένα πρόγραμμα το οποίο επέτρεπε να δοθούν από θέματα τα οποία δεν είχαν πουληθεί προς κάποιους οργανισμούς οι οποίοι κάναν διανομή τροφίμων ή οργάνωναν συσίτια ή δίνανε κάποια πακέτα, δέματα με γεωργικά προϊόντα τα οποία δεν είχαν πουληθεί. Σιγά σιγά τα προγράμματα αυτά εξαφανίστηκαν εξαιτία των νέων λογικών τη αγορά στα πλαίσια του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου και σιγά σιγά είδαμε ότι και στην Ευρωπαϊκή Ένωση αρχίσαμε όλο και περισσότερο να έχουμε κάποιες χρηματοδοτικές ενισχύσεις από τα κράτη-μέλη. Επομένως, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο ακριβώς αυτό καταδίκασε, την αλλαγή της φύσης της επιστηστικής αυτής βοήθειας και ουσιαστικά τη στρέβλωση η οποία είχε προκύψει σε σχέση με τον κανονισμό αυτό. Και για αυτό το λόγο ορισμένα κράτη όπως η Γερμανία κάνανε προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Τώρα, βάσει της απόφασης του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, το πρόγραμμα αυτό το οποίο θα έπρεπε να ολοκληρωθεί από το 2012 μετά από την κινητοποίηση των πολιτών καθώς επίσης και μετά την τοποθέτηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θεωρήθηκε ότι θα έπρεπε να τροποποιηθεί από πολιτικής πλευράς. Η πρώτη πολιτική λύση που προτάθηκε ήταν να παραταθεί το πρόγραμμα αυτό μέχρι το 2013 και η δεύτερη λύση ήταν η ε, γενικότερη αναθεώρηση του κανονισμού λαμβάνοντας υπόψη την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Και τελικά αυτό προτείνεται σήμερα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή των συναδέλφων σε ένα σημείο το οποίο είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τη δική μας την Επιτροπή. Η νομική βάση. Νομική βάση στην οποία βασίζεται το νέο αυτό ταμείο. Πρόκειται για το άρθρο 175 της συνθήκης. Το άρθρο αυτό ανήκει στον τίτλο 18 της συνθήκης, η οποία αναφέρεται στην οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και θα ήθελα επίση να αφαιρθώ στη μελέτη αντικτύπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία διευκρινίζει ότι το βασικό μέσο τη Ευρωπαϊκή Ένωση προκειμένου να προωθηθεί η απασχολησιμότητα, να καταπολεμηθεί η ένδυα είναι ακριβώς το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Η νομική ανάλυση κατέδειξε ότι χρειάζεται ένα ξεχωριστό μέσο, δεδομένου ότι η νομική βάση 162 του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου προβλέπει μια κοινή δράση στα πλαίσια των κρατών μελών. Επομένως, δικαιολογείται βάση του άρθρο 174 η πρόταση αυτή εφόσον προβλέπεται μια εναρμονισμένη πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και επίσης δικαιολογείται και βάση του άρθρου 175 του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου με τη χρησιμοποίηση των διαρθρωτικών ταμείων. Αναφέρομαι στα άρθρα αυτά για να σας πω ότι τελικά η έκθεση αυτή είναι πάρα πολύ σημαντική για τη δική μας την Επιτροπή, γιατί ουσιαστικά εντάσσεται στην περίμετρο της πολιτικής συνοχής. Και γι' αυτό το λόγο θεωρώ ότι η δική μας η Επιτροπή θα μπορούσε πραγματικά να είναι η αρμόδια επί της ουσίας Επιτροπή. Λαμβάνω υπόψη μου τα όσα μου είπε η Γραμματεία, στα πλαίσια της, και αναφέρομαι επίσης και στην ενισχυμένη συνεργασία, την οποία θα έχουμε με την Επιτροπή Απασχόλησης. Θεωρώ πάντως ότι εμείς θα μπορούσαμε να προωθήσουμε πάρα πολύ μέσα από την έκθεση αυτή, μέσα από την γνωμοδότηση αυτή, την περιφερειακή πολιτική. Όσον αφορά τώρα τον συγκεκριμένο κανονισμό, τον προτινόμενο κανονισμό, νομίζω ότι θα πρέπει καταρχάς να θέσουμε το ζήτημα το χρηματοδοτικό. Το συνολικό ποσό το οποίο θα δοθεί για το ταμείο αυτό θα είναι 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ για την περίοδο 2014-2020 και η συμμετοχή των κρατών μελών θα καλύψει το 15% των δαπανών των εθνικών προγραμμάτων. Το υπόλοιπο 85% θα καλυφθεί από τα κοινοτικά ταμεία. Το δεύτερο σημείο του κανονισμού αναφέρεται στο πεδίο εφαρμογής του ταμείου αυτού, το οποίο θα ισχύει προφανώς σε όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά προβλέπει επίσης και την διανομή των τροφίμων. Αναφέρεται ουσιαστικά σε έναν εξοπλισμό ο οποίος δεν προβλεπόταν στο προηγούμενο πρόγραμμα. Δηλαδή γίνεται συγκεκριμένη αναφορά στη διανομή ρούχων, υποδημάτων και το καθεξής. Γίνεται μια λεπτομερής αναφορά σε όλα αυτά τα είδη τα οποία χρειάζονται οι πιο άποροι πολίτες. Θεωρώ ότι εδώ πέρα υπάρχουν όμως και κάποια προβλήματα. Καταρχάς, από ό,τι φαίνεται, διευρύνουμε το πεδίο εφαρμογής του προγράμματος, αλλά από την άλλη μειώνουμε, μειώνουμε τα κονδύλια τα οποία δίνουμε σε αυτό το πρόγραμμα. 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ μας λένε οι οργανώσεις ότι δεν φτάνουν. Θα πρέπει να διπλασιαστεί το ποσό αυτό. Δηλαδή να διατεθούν περίπου 4 δισεκατομμύρια προκειμένου πραγματικά να αποκριθούμε στις επισητιστικές και μόνο ανάγκες των απόρων. Θεωρώ λοιπόν ότι εδώ πέρα υπάρχει ένα σημαντικό πρόβλημα και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να κάνει κάτι, θα πρέπει να τοποθετηθεί πολύ ισχυρά Ιδίω πριν από την επόμενη Ευρωπαϊκή Σύνοδο, προκειμένου να καταφέρουμε να πούμε προς αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων ότι πρέπει να σταθούμε στο ύψο των περιστάσεων, στο ύψο των αναγκών των περισσότερων οργανώσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης που λειτουργούν υπέρ των απόρων. Υπάρχει και ένα ακόμα πρόβλημα το οποίο σχετίζεται περισσότερο με τι περιφέρειες φοβόμαστε ότι τα κράτη-μέλη τελικά δεν θα έχουν τα απαραίτητα οικονομικά χρηματοδοτικά μέσα για να χρηματοδοτήσουν το πρόγραμμα αυτό και ότι θα βασιστούν πολύ περισσότερο στην τοπική αυτοδιοίκηση. Θα ζητήσουν τελικά από την τοπική αυτοδιοίκηση να πληρώσει το λογαριασμό. Και ξέρετε ότι στι περισσότερε χώρε, σε πολλέ αν μη τι άλλο χώρε, τα χρήματα αυτά δεν υπάρχουν σε τοπικό επίπεδο. Επίσης είναι πάρα πολύ σημαντικό να συνειδητοποιήσουμε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει και για το ζήτημα αυτό να τοποθετηθεί ιδιαίτερα στεναρά, να έχουμε ένα ενιαίο μέτωπο. Ξέρετε ότι ε, εναπόκειται σε εμά να λάβουμε δράση. 116 περίπου εκατομμύρια άνθρωποι απειλούνται από την ένδια. Περίπου ε, 18 εκατομμύρια δέματα τροφίμων και άλλων ειδών έχουν διανεμηθεί, αυξάνονται όμως όλο και περισσότερο οι απαιτήσει και οι ανάγκες. Πρέπει εμεί να ανταποκριθούμε στις νέες αυτές ανάγκες και θα πρέπει να ζητήσουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κάνει σε κάποια σημεία και για κάποια ζητήματα διορθώσεις και βελτιώσεις. Αναφέρθηκα στο ζήτημα της ένδυσης των ρούχων. Πέρα από αυτό όμως, νομίζω ότι θα πρέπει να υπάρχουν και τα απαραίτητα κονδύλια για να ανταποκριθούν τα κράτη-μέλη στο πρόγραμμα αυτό και στι απαιτήσει του. Σας ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο που μου διαθέσατε. Πιστεύω ότι θα γίνει μια ανταλλαγή απόψεων και προσβλέπω και σε μελλοντικές συζητήσεις για να καταφέρουμε να βελτιώσουμε την έκθεση αυτή. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κύριε η σκιώθηση συγγήτρια του ΕΛΚ θα λάβει πρώτη τον λόγο. Η κυρία Σάντσες Σμιτ. Παρακαλώ, έχετε τον λόγο κυρία Σάντσες Σμιτ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ και τον συγητή για την πληρέστατη παρουσίαση. Θα ήθελα καταρχάς να σας επενθυμίσω ότι το θέμα αυτό αποτελεί ένα καταπληκτικό παράδειγμα ενός θέματος όπου όλοι οι βουλευτές, ανεξαρτήτως ε, οικογένειας πολιτικής, ε, δίνουν τον κοινό αγώνα για να σωθεί αυτό το ταμείο. Έχουμε ψηφίσει πολλά ψηφίσματα, έχουμε υποβάλει και γραπτές ερωτήσεις ε, προς την Κομισιόν. Πολύ καλή δουλειά κοινή λοιπόν. Θα ήθελα πραγματικά να χαιρετήσω και τη μάχη των φιλανθρωπικών οργανώσεων που κατάφεραν να ευαισθητοποιήσουν την κοινωνία των πολιτών και είδαμε μια πραγματική κινητοποίηση σε όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, που τα αφορά πιο πολύ αυτό το ταμείο. Και επίσης θα πρέπει να βρεθούν οι τεχνικοί, νομικοί και οικονομικοί πόροι για τον νέο κανονισμό. Υπάρχουν κάποιες ε, ε, γκρίζε ζώνες ακόμη, υπάρχουν κάποιες σκιέ και ξέρουμε ότι υπάρχει μια διαδικαστική ακαμψία σε κάποιες χώρες που απέτρεψε τις επικοδομητικέ συζητήσεις. 116 εκατομμύρια άτομα, όπως είπε και ο εισηγητή, απειλούνται με ένδια ή κοινωνικό αποκλεισμό. 40 εκατομμύρια δεν έχουν ε, τα προστοζήν και θα ήθελα να σας δώσω ένα παράδειγμα στη χώρα μου. Έχουμε την πολύ γνωστή οργάνωση τα εστιατόρια της καρδιάς, Γαϊστόντικερ. Πάνω από 115 εκατομμύρια γεύματα έχουμε διανύμει. Και το 23% ε, ε, βοηθά χρηματοδοτείται και από την Ευρωπαϊκή Ένωση διανομή τους. Θέλω να σας πω ότι έχουμε ένα ποσό 2,5 δις, είπε ο κύριος Μαρζή, για την επόμενη περίοδο. Εγώ είχα, νόμιζα ότι είναι λιγότερα τα κονδύλια. Δεν θέλουμε όμως να διαταραχθεί το πρόγραμμα αυτό το επισητιστικό. Δεν έχει οριστεί ακόμη το ποσό για τον προπολογισμό. Ο εισηγητή είπε πολύ καλά για πού προορίζονται αυτά τα κονδύλια. Επίση πρέπει να πούμε ότι οι νέε διαδικασίε μπορεί να είναι πολύπλοκε και θα ήταν καλό να επανέλθουμε στο παλαιό σύστημα, απλέ διαδικασίε, αγορά τροφίμων, επιστημική βοήθεια ή ίσω ε, αντιπροσωπεία σε φιλανθρωπικά ιδρύματα με εθνική συγχρηματοδότηση. Πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι είναι συμπληρωματικά τα διεθνωτικά ταμεία και δει το ΕΚΤΑ Πρέπει να παρασχεθεί βοήθεια στους ε, άπορους, γιατί αυτό είναι και ένα στόχος της πολιτικής συνοχής. Πρέπει λοιπόν να δοθεί κατεπίγουσα βοήθεια. Έχει δοθεί χάρη σε αυτό το ταμείο. Έχει παρασχεθεί και εκπαίδευση στο πλαίσιο της έκτα και έχουν δημιουργηθεί και θέσεις εργασίας χάρη στις επενδύσεις από το Ταμείο Επενδύσεων, το ΦΕΝΤΕ. Σας ευχαριστώ κυρία Σάντσια Σμιτ. Ο κύριος είπε επόμενος, παρακαλώ. Κύριε Τυρολή, παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, αν μου επιτρέπετε, και κατόπιν ετοίματος της κυρίας Ντάντσιλα, θα την εκπροσωπήσω και θα διαβάσω ουσιαστικά την παρέμβασή της. Καταρχάς, λοιπόν, ε, χαιρετίζω το έργο της ηγητή και ελπίζω να μπορέσουμε να δώσουμε απάντηση στις προσδοκίες των πλέον ενδεών, ιδίως ε, το 2013 που είναι το Ευρωπαϊκό Έτος των Πολιτών όλοι όσοι έχουν ανάγκη θα πρέπει για μια ακόμη φορά να γνωρίζουν ότι είναι αλληλέγγυη η Ευρώπη απέναντί τους, ότι έχει τη βούληση να τους βοηθήσει, να αντιμετωπίσουν ε, την ψηφαλή κατάσταση στην οποία βιώνουν και να μπορέσουν να ενταχθούν στην κοινωνία. Η οικονομική κρίση ευθύνεται για την αύξηση των ατόμων που απειλούνται από τη φτώχεια και τα οποία ε, χρειάζονται ε, βοήθεια, ευρωπαϊκή βοήθεια. Ο προπολογισμό του προγράμματο έχει μειωθεί κατά 40% περίπου. Βλέπουμε ε, σήμερα και αυτό υπογραμμίζεται και στις εκθέσεις ε, των αρμόδιων ε, οργανισμών, αρμόδιων για την εφαρμογή του προγράμματος, ότι είναι μακρύς ο κατάλογος των ενδεών, των αστέγων, μονογονεϊκών οικογενειών, ανέργων ή ατόμων που δεν λαμβάνουν πλέον επίδομα ανεργίας ή και ατόμων που ζουν στο σπίτι τους, ακόμη την οικογένειά τους, γιατί δεν έχουν δική τους κατοικία. Επίσης, επισφαλής στην των φοιτητών, των συνταξιούχων, ατόμων που δεν έχουν οικογένεια, ατόμων που μπορεί να έχουν ή να μην έχουν οικογένεια, αλλά αντιμετωπίζουν κάποια νοητική ή σωματική αναπηρία και δυσκολεύονται να πληρώσουν το ενίκιο του ε, και ακόμη και να εξασφαλίσουν ε, τροφή. Θα πρέπει λοιπόν να, ε, πρώτα απ' όλα να εντοπίσουμε όλα αυτά τα άτομα και να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τα άτομα αυτά μέσω του ταμείου ή να δούμε τι γίνεται με τις ε, εγγύους ή με τις νέες ε, μητέρες με παιδί μικρό που ζουν ε, στην επαρχία. Ποιες από αυτές χρειάζονται βοήθεια. Σίγουρα θα πρέπει επίσης να φροντίσουμε και την ε, επιστηστική εκπαίδευση, τον εμβολιασμό, την παροχή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. Θέλουμε με το Ταμείο αυτό και με αυτό το πρόγραμμα να προσφέρουμε ποιοτική βοήθεια στα άτομα τα οποία τη χρειάζονται σε περιπτώσεις ανάγκης και θέλουμε στα ενδέη αυτά άτομα να εξασφαλίσουμε τη μέρημνα, τη φροντίδα και να μπορέσουμε να επανενταχθούν τα άτομα αυτά στην κοινωνία. Θα πρέπει επίσης ε, να βοηθήσει και την κοινωνική και την οικονομική ένταξη αυτών των ατόμων. Γιατί αυτά τα άτομα πρέπει να μπορούν να βγουν από το σπίτι τους για να έχουν κοινωνικές σχέσεις και να μπορούν να ξανενταχνούν στην κοινωνία. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι σήμερα το πρόγραμμα αυτό εφαρμόζεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο με τη βοήθεια 31.000 ενώσεων. 800 είναι στο τύπο απασχολούνται, αλλά 10.000 και πάνω είναι εθελοντές οι οποίοι βοηθούν. Και μεταξύ των μισθωτών βλέπουμε άτομα τα οποία ε, παίρνουν αυτή την βοήθεια από την Ένωση στο τέλος του μήνα. Θα πρέπει η Ένωση να προβλέψει ένα ταμείο εκτακτής ανάγκης ε, για τέτοιες καταστάσεις και θα μπορεί να παρεμβαίνει σε περίπτωση που επιδεινώνει την κατάσταση. Επίσης τα κρατημέλη θα πρέπει να μπορούν να δίνουν κάποιες διευκολύνσεις ε, στο γεωργοδιατροφικό κλάδο, στην αλυσίδα διανομής τροφίμων όταν, παραδείγματο χάρη, τα τρόφιμα φτάνουν σχεδόν στην ημερομηνία λήξη και δεν πολλούνται, θα πρέπει να φτάνουν εύκολε στι αποθήκε των ε, τραπεζών τροφίμων, ώστε να αποφευθεί η κατασπατάληση των τροφίμων που δεν μπορέσαν να πουλήσουν ε, τα σούπερ μάρκετ, για παράδειγμα. Και όταν βέβαια είναι ακόμα βρόσιμα καταναλώσουμε αυτά τα προϊόντα. Θα πρέπει επίση να είναι μεγαλύτερη ποικιλία των διανεμόμενων προϊόντων. Να μην είναι περιορισμένη η ποικιλία επειδή λέγεται ότι ουσιαστικά ε, μόνο τα, επιλέξιμα προϊόντα προς δημόσια αποθήκευση είναι αυτά τα οποία μπορούν να λάβουν μέρος σε αυτό το πρόγραμμα. Θα πρέπει λοιπόν να ε, έχουμε υπόψη μας όλα αυτά τα ζητήματα, αλλά και την πολιτική, την κοινωνική. Θέλουμε να βελτιώσουμε την συνολική μας προσέγγιση. Και τώρα Προσωπικά, να επιτρέπετε κύριε Πρόεδρε, να προσθέσω και εγώ κάποια πράγματα. Να πω ότι σήμερα μελετούμε μια πρόταση με μεγάλη, τεράστια συμβολική σημασία ε, που δεν συνάδει με τους πόρους που βλέπουμε να χορηγούνται και γι' αυτό βλέπουμε να διακινδυνεύεται αυτή η βοήθεια Και πραγματικά υπάρχουν κάποια επιχειρήματα που ίσως να ήταν σκόπιμα για τη μείωση αυτών των πόρων, αλλά πραγματικά πρέπει να έχουμε υπόψη μας τι θα συνιστούσε μια μείωση της πρικοδότης αυτού του προγράμματος. Τι στηρίζουμε τελικά περισσότερο, τις τράπεζες και όχι τους πολίτες. Όχι, πρέπει να προσπαθ... προασπίσουμε το πρόγραμμα αυτό γιατί δίνει ένα διαφορετικό πρόσωπο της Ευρώπης προς τα έξω. Όταν συζητήσαμε την πολιτική συνοχή, εγώ είχα πει ότι θα πρέπει το πρόγραμμα αυτό να επαναξιολογηθεί ως προς την πρικοδότησή ε, του, γιατί είναι ε, επίκαιρο όσο ποτέ άλλοτε. Θα πρέπει να στείλουμε λοιπόν με την έκθεση αυτή σαφές μήνυμα και εγώ θα καταθέσω και τις τροπολογίες που θα κρίνω σκόπιμα. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Σας ευχαριστώ πολύ. Στον κατάλογο έχουμε Έξι που έχουν ζητήσει τον λόγο, έξι ευρωβουλευτές. Θα τα καταφέρουμε, πρέπει να βιαστούμε και να είμαστε σύντομοι, να το λάβετε υπόψη. Η, η κυρία Ντέλη, επόμενη που θα λάβει τον λόγο, παρακαλώ. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι ε, οι Ευρωπαίοι υπεύθυνοι έχουν γίνει τόσο ανέστητοι αυτή τη στιγμή που δεν δείχνουν μια ενεργή αλληλεγγύη απέναντι πιο ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού. Έχουμε μια στρατηγική Ευρώπη 2020, σύμφωνα με την οποία πρέπει να μειωθούν κατά 20 εκατομμύρια τα άτομα αυτά τα οποία βρίσκονται κάτω από το κατόφλι της φτώχειας. Τα, πίσω από τα στατιστικά όμως αυτά δεδομένα έχουμε άνδρες, γυναίκες και παιδιά τα οποία πραγματικά υποφέρουν. Κάνω λοιπόν μία έκκληση προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το οποίο θα πρέπει να αναλάβει ουσιαστική δράση, όπως μπορεί να το κάνει. Η δική μας η Επιτροπή θα πρέπει πραγματικά να αναλάβει δράση. Ακούσαμε κάποια αριθμητικά δεδομένα πάνω από 115 εκατομμύρια Ευρωπαίοι σήμερα απειλούνται από τη φτώχεια. Ανάμεσα στους ανθρώπους αυτούς, 40 εκατομμύρια δεν έχουν πρόσβαση σε υγιή διατροφή και 18 εκατομμύρια Ευρωπαίοι εξαρτώνται από το επιστημιστικό ταμείο. Η πρώτη ε, αποδοκιμασία που θα μπορούσα να κάνω, η πρώτη επίκριση για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους έχει να κάνει με την μείωση, με το περιορισμένο ποσό από 3,5 δισεκατομμύρια, περνάμε σε 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Περιορισμός λοιπόν της χρηματοδότησης. Επομένως η πρώτη μάχη που πρέπει να δώσουμε είναι να πούμε ότι θα πρέπει να καταφέρουμε να διατηρήσουμε τον πρώτερο προπολογισμό, τον υψηλό προπολογισμό. Επίσης ξέρετε ότι δίνουμε μία μάχη για τον κοινοτικό προπολογισμό, στα πλαίσια του οποίου βλέπουμε ότι ο προπολογισμό προβλέπεται για την πολιτική συνοχή θα μειωθεί. Πρέπει λοιπόν να στείλουμε ένα ξεκάθαρο μήνυμα. Το ποσό θα πρέπει να διατηρηθεί. Δεύτερον, στο παρελθόν οι οργανώσεις εταίροι λάμβαναν άμεσα τις ενισχύσεις αυτές. Ενώ τώρα με τον, νέο, με τον νέο χρηματοδοτικό μηχανισμό βλέπουμε ότι προβλέπεται συγχρηματοδότηση. Για παράδειγμα στη Γαλλία προβλέπεται συγχρηματοδότηση της του 15%. Σε χώρες όμως όπου η κοινωνική και η οικονομική κατάσταση είναι καταστροφική, πώς θα είναι ποτέ σε θέση να θεσπιστούν προγράμματα συγχρηματοδότησης. Επομένως, δεν θα καταφέρουν οι χώρες αυτές να χρησιμοποιήσουν αυτό το πρόγραμμα ακριβώς επειδή θα πρέπει να χρηματοδοτήσουν άλλα προγράμματα, θα δώσουν προτεραιότητα σε άλλα προγράμματα. Θα πρέπει λοιπόν να ασχοληθούμε και με την διάταξη αυτή της χρηματοδότησης. Τρίτη κριτική που θα ήθελα να κάνω. Ξέρετε ότι υπολείπεται πάρα πολύ πρόταση αυτή από αυτό το οποίο εμεί θα θέλαμε. Νομίζω όμως ότι θα πρέπει πραγματικά να τα αποκριθούμε ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στα διαρθρωτικά αίτια της φτώχειας πότε πραγματικά θα ασχοληθούμε με τα διαρθρωτικά αίτια της φτώχειας. Κάθε φορά που μιλάμε για την πολιτική για την καταπολέμηση της φτώχειας, μιλάμε για το ότι θα πρέπει να δημιουργηθεί μία πλατφόρμα σφαιρικής αντιμετώπισης του προβλήματος. Τι περιμένουμε όμως για να λάβουμε δράση. Μιλάμε σήμερα για την επιστηστική βοήθεια, αλλά από την άλλη υπάρχουν και άστεγοι, παιδιά τα οποία δεν έχουν κάποιες βασικές υποδομές, ενώ υποτίθεται ότι έχουμε μια ευρωπαϊκή στρατηγική για να αντιμετωπίσουμε όλα αυτά τα, τα προβλήματα. Τι περιμένουμε. Πρέπει να σας πω ότι 20 από τις 27 χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης θα χρησιμοποιήσουν αυτά τα προγράμματα επιστηστικής βοήθειας. Βλέπουμε ότι υπάρχει μια αντίδραση από κάποια κράτη-μέλη στο Συμβούλιο. Πρέπει να κινητοποιηθεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, γιατί πραγματικά υπάρχουν πάρα πολλοί πολίτες που για να επιβιώσουν εξαρτώνται από τα προγράμματα αυτά. Η έκθεση βέβαια αυτή θα πρέπει να διαρθρωθεί με την περιφερειακή πολιτική. Κατά ποιο τρόπο. Πρώτον, εμείς θα πρέπει να προωθήσουμε κάποιες ε, καινοτομίες στην διαχείριση της επισητιστικής βοήθειας. Και αυτό γιατί στόχος μας είναι ακόμα και οι πιο φτωχοί να έχουν πρόσβαση σε μια υγιεινή βιώσιμη διατροφή. Πρέπει λοιπόν να στηρίξουμε περιφερειακά καινοτόμα οικολογικά προγράμματα σαν αυτά τα οποία υπάρχουν στη δική μου την περιοχή, στην περιοχή του Ατού Σαρόντ, προγράμματα τα οποία υλοποιούνται μέσω της οργάνωσης UNITE. Υπάρχει μια συνεργασία μέσω κάποιων καταστημάτων τροφίμων που προσπαθούν να βοηθήσουν τους ανθρώπους δίνοντας συστηματικά τρόφιμα και λαχανικά. Φρούτα και λαχανικά, με συγχωρείτε. Επίσης, θα πρέπει να προωθήσουμε όλες αυτές τις δράσεις οι οποίες δημιουργούν μια καλύτερη ελεγγύη ανάμεσα στον παραγωγό και τον καταναλωτή. Γιατί ξέρετε ότι ε, οι επισητιστικές τράπεζες μπορούν πραγματικά να αποτελέσουν ένα χώρο κοινωνικής αλληλεγγύης, όπου πραγματικά ακούμε τους άπορους και δεν τους φέρνουμε σε δύσκολη θέση και μπορούν, για παράδειγμα, να γίνουν παράλληλα και κάποια άλλα προγράμματα, όπως προγράμματα καταπολέμησης των αναλφαβητισμού κτλ. Πιστεύω λοιπόν ότι θα πρέπει να προωθήσουμε και αυτά τα προγράμματα. Και τρίτον, νομίζω ότι θα πρέπει να έχουμε και μία τοπική πλέον γεωργική παραγωγή. Το είπαν αυτό και άλλοι. Διανύουμε μια οικονομική κρίση σήμερα. Κανεί όμως δεν μιλάει για το ρόλο που θα μπορούσε να διαδραματίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση προκειμένου να ρυθμιστούν σωστά οι τιμές των τροφίμων. Ολοκληρώνω την παρέμβασή μου αυτή λέγοντας το ακόλουθο. δεν νομίζω ότι θα πρέπει να προσεγγίσουμε το μηχανισμό αυτό ως απλό φιλανθρωπικό οργανισμό, ως ένα, ως ένα απλό φιλανθρωπικό πρόγραμμα. Εμείς αυτή τη στιγμή θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι προασπίζουμε ένα θεμελιώδες δικαίωμα των Ευρωπαίων πολιτών να έχουν πρόσβαση σε τρόφιμα καταγράφεται αυτό στη συνθήκη μα ω θεμελιώδη δικαίωμα των Ευρωπαίων πολιτών. Αυτή είναι η πρώτη μα προτεραιότητα. Δεύτερον, θα πρέπει να διατηρήσουμε προφανώ το Ταμείο αυτό. Δεν χρειαζόμαστε όμω απαραίτητα ένα εξειδικευμένο πρόγραμμα. Και τρίτον, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η γενικότερα Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να δείξουν ότι υποστηρίζουν ένα πραγματικό φιλολαϊκό πρόγραμμα το οποίο θα στείλει και ένα μήνυμα συμφιλίωσης ανάμεσα στην Ευρώπη και τους πολίτες Σας ευχαριστώ. Σα ευχαριστούμε. Πέντε λεπτά για τέσσερις που απομένουν τώρα. Πώς θα τα καταφέρουμε. Παρακαλώ να το λάβετε υπόψη να είστε σύντομοι. Η κυρία δεν ξέρω το όνομά σας, δεν το πρόφερα σωστά, Μένοβα. Ευχαριστώ πολύ, δεν έχουμε και πολύ χρόνο. Να συγχαρώ τον εισηγητή. Τι να πω. Να πω ότι πρέπει αυτά τα στατιστικά στοιχεία που μας αναφέρατε, κύριε Σιγητά, τα τελευταία αυτά δεδομένα της Eurostat από το 2011, αυτά, αυτά αναφέρομαι, αλλά θα πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη ότι αυξάνει ο αριθμός των αστέγων στην Ευρώπη. Τα τελευταία πέντε χρόνια στα 15 κράτη μέλη της Ένωσης αυξήθηκε και επίσης όλο και περισσότερες ΜΚΟ ζητούν να γίνει δεκτή μια ευρωπαϊκή στρατηγική για την καταπολέμηση του φαινομένου αυτού των αστέγων. Επίσης, η οικονομική κρίση συνεχίζεται, φτωχαίνει ο πληθυσμός στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα, κατά την άποψή μου, οι κυβερνήσεις που θα χρειαστεί να διαχειριστούν αυτά τα κονδύλια θα πρέπει να εφαρμόσουν πιο ελαστικούς κανόνες για να βοηθήσουν ευρύτερα κοινωνικά στρώματα η διαδικασία που προβλέπει το πρόγραμμα ε, ίσως ε, βοηθήσουν να φτάσουν ε, το συντομότερο με τόσους δικαιούχους ε, τα κονδύλια σε συνεργασία και συνάντηση και με τα άλλα κοινωνικά προγράμματα. Επίσης πρέπει να υπάρχει και οικονομικός έλεγχος, αυστηρός οικονομικός έλεγχος, αλλά με τρόπο που δεν θα προσβάλλει την αξιοπρέπεια των ενδεών ατόμων θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε με αποτελεσματικό και αποδετικό τρόπο αυτή τη διαδικασία και αυτό το μέσο. Ευχαριστώ. Είσαστε, πραγμα... πραγματικά πολύ σύντομοι και περιεκτικότατοι. Παρακαλώ εσείς κύριε Χρυσόγελε, έχετε τον λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είναι σίγουρο ότι η κρίση έχει αυξήσει τον αριθμό των απόρων και φτωχών και η Ευρώπη πρέπει να δείξει ότι είναι μια Ευρώπη της αλληλεγγύης το ταμείο, αυτό που συζητάμε εδώ πέρα, το Ευρωπαϊκό Ταμείο για τους Απόρους στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα έχει πόρους που δεν ξεπερνούν το 1% του κόστου των προγραμμάτων διάσωσης των χωρών του, του Νότου. Επομένως μιλάμε για ένα πολύ μικρό, αλλά βέβαια παραμένει σημαντικό ταμείο για την ενίσχυση των ανθρώπων που είναι στα όρια της επιβίωσης προφανώς πρέπει να συνεχιστεί για την περίοδο 2014-2020 και οι δράσεις αυτού του Ταμείου θα πρέπει να συνδυάζονται και να συνδέονται με τις άλλες πολιτικές που έχουν σαν στόχο να εξαλείψουν τη φτώχεια. Θυμίζω ότι έχουμε αφασίσει ότι η στρατηγική Ευρώπη 2020 στοχεύει στο να μειώσει τον αριθμό των φτωχών σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ενώ αυτό που συμβαίνει σήμερα είναι η αύξηση του αριθμού των φτωχών και από την άλλη μεριά έχουμε και νέες μορφές φτώχεια που δεν είχαμε σε τόσο μεγάλη ένταση στην Ευρώπη, όπως είναι η ενεργειακή φτώχεια, δηλαδή οι άνθρωποι που δεν έχουν πρόσβαση σήμερα στη θέρμανση, στον κλιματισμό του σπιτιού του. Ε, σίγουρα θα πρέπει να απλοποιηθούν οι διαδικασίες αλλά κυρίως αυτό που θα πρέπει να γίνει είναι να δώσουμε έμφαση στο αποτέλεσμα δηλαδή πράγματι αυτοί που θα υποφελούνται από το Ταμείο να υποφελούνται πραγματικά, να καταναλώνουν προϊόντα τα οποία είναι ποιοτικά, δεν θα είναι προϊόντα τα οποία απλώς έχουν περισσέψει μια διαδικασία, επειδή Νάποροι δεν σημαίνει θα πρέπει να έχουν και υποβαθμισμένη πρόσβαση, να έχουν πρόσβαση σε υποβαθμισμένα προϊόντα. Άρα αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να συνδυάσουμε και το Ταμείο με την ενίσχυση μιας παραγωγής που είναι ποιοτική, οικολογική και υγιεινή. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Να μην απλώς χρησιμοποιήσουμε την ένδια των ανθρώπων ως ευκαιρία για να ξεφορτωθούμε πράγματα τα οποία δεν είναι ποιοτικά. Και βέβαια μέσα στους όρους του Ταμείου νομίζω θα πρέπει να είναι και η συνέργεια με διαδικασίε οι οποίε προβλέπουν την κοινωνική επανένταξη των ανθρώπων που σήμερα έχουν χάσει το επάγγελμά του, δεν έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίε. Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι σήμερα που, δεν έχουν, που είναι και άνεροι και δεν έχουν πρόσβαση στο σύστημα υγεία στην Ελλάδα. Πάνω από το 20-30% σήμερα δεν έχει πρόσβαση σε ένα αξιοπρεπέ σύστημα υπηρεσιών υγεία. Άρα θα πρέπει να δούμε και τέτοιε διαδικασίε συμπληρωματικά μέσα από άλλε πολιτικέ που θα συνδυάσουν αυτά τα δύο. Και εγώ σας ευχαριστώ. Κορώνα παρακαλώ. Κορώνα έχετε τον λόγο. Ε, Κοιτάξτε δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο. Δύο λοιπόν παρατηρήσεις θα κάνω και μία ερώτηση στη συνέχεια προς τον εισηγητή. Πρώτη παρατήρηση. Νομίζω ότι και η δική μας Επιτροπή θα πρέπει να ασχοληθεί ιδιαίτερα με την απόκληση που βλέπουμε πλέον ανάμεσα στην Ευρώπη και τους πολίτες της. Το χάσμα αυτό το οποίο δημιουργείται. Νομίζω ότι αυτό είναι πάρα πολύ επιζήμιο. Και ήταν ε, ιδιαίτερα επιζήμια η όλη συζήτηση που έγινε για τα χρήματα αυτά που έπρεπε να δοθούν σε κάποιες περιφέρειες για να αντιμετωπίσουν τους σεισμούς και νομίζω ότι επιζήμια ήταν και επιπτώσεις από τη χαμηλή χρηματοδότηση του προγράμματος αυτού που βασίζεται πάρα πολύ στην τοπική αυτοδιοίκηση τελικά. Και ως προς αυτό λοιπόν ω Επιτροπή περιφερειακή Ανάπτυξης εμείς θα πρέπει να στείλουμε ένα πολύ δυνατό μήνυμα. Ακόμα και όσον αφορά τη χρηματοδότηση, τη χρηματοδότηση του Ταμείου αυτού. Τώρα δεύτερη παρατήρηση που απευθύνεται περισσότερο στον εισηγητή. Νομίζω ότι θα πρέπει πραγματικά να υπάρχει εδώ πέρα μία διασύνδεση ανάμεσα στο σχέδιο αυτό, το ταμείο αυτό και το ψήφισμα εκείνο το οποίο εμεί εγκρίναμε πριν από ένα χρόνο κατά τη διατροφική πατάλη. Θα θυμάστε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με πάρα πολύ μεγάλη πλειοψηφία ενέκρινε ένα ψήφισμα το οποίο καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αρχίσει να λαμβάνει σε ευρωπαϊκό επίπεδο δράσει, δράσει οι οποίε θα περάσουν έπειτα σε εθνικό και σε τοπικό επίπεδο προκειμένου πραγματικά να καταπολεμηθεί η κατασπατάληση των τροφίμων. Το θέμα αυτό συνδέεται πάρα πολύ και με το ταμείο το οποίο συζητάμε τώρα. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό στο κείμενο της γνωμοδότησης, στην έκθεση, να γίνεται μια κάποια μνήα, μια αναφορά στο ψήφισμα αυτό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Και ως προς αυτό βέβαια θα υποβάλω και σχετική τροπολογία. Ευχαριστώ πολύ. Ο Νίλσον και μετά πολύ σύντομα ο εισηγητής. Ευχαριστώ πολύ. Θα προσπαθήσω να είμαι πολύ σύντομος, Πρόεδρε. Η φτώχεια. Η φτώχεια αυξάνει παντού, αυξάνεται παντού στην Ευρώπη. Υπάρχει όλο και μεγαλύτερη ανεργία. Ζούμε σε μια περίοδο κρίση. Σε μια τέτοια κατάσταση είναι φυσικά δύσκολο ένα τέτοιο θέμα να το διαμορφώνουμε όπως εγώ θα επιθυμούσα. Δηλαδή να ρωτώ, διαρωτηθούμε ποια είναι η ευθύνη μας στο τοπικό, περιφερειακό, εθνικό επίπεδο ώστε να βοηθήσουμε τους φτωχούς. Θέλω δύο πράγματα να επισημάνω. Πρώτον, εγώ ομιλώ από εκπείρας. 15 χρόνια ήμουν δήμαρχος στη Σουηδία. Στο τοπικό επίπεδο έχουμε διατάξεις για την ευθύνη, ευθύνη, υπευθυνότητα που έχουμε έναντι των πτωχών, για την ενδυμασία τους, τη στέγασή τους, ε, την σύντησή τους στο τοπικό επίπεδο. Σύμφωνα με την νομοθεσία μας είμαστε εμείς υπεύθυνοι. Συνεργαζόμαστε με άλλους αρμόδιους ώστε τα προβλήματα να μπορέσουν να επιληθούν τα προβλήματα των φτωχών. Αυξάνει αυξάνεται η φτώχεια στην Σουηδία. Η καλύτερη δυνατότητα για να αντιμετωπιστεί η φτώχεια είναι να δημιουργηθούν θέσει απασχόληση. Να υπάρχει δουλειά. Δουλειά ώστε οι φτωχοί να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τα προβλήματά του. Έτσι μπορούμε με τέτοιε προσπάθειε να προσπαθήσουμε να εκριζώσουμε, να καταπολεμήσουμε τη φτώχεια. Γι' αυτό ανησυχώ Ανησυχώ για αυτή την κατάσταση. Φυσικά έχει απόψει αυτή η Κοινοβουλευτική Επιτροπή για τι πιθανέ επιπτώσει των κονδυλίων του Κοινωνικού Ταμείου για την δημιουργία θέσεων απασχόληση. Υπάρχουν σημαντικά σχέδια και προγράμματα στο τοπικό επίπεδο για τα κράτη-μέλη για να δημιουργηθούν θέσει απασχόληση και να υπάρχουν δυνατότητες που θα βελτιώσουν, θα βελτιωθεί η αγορά εργασίας με αυτά τα κονδύλια. Αυτά τα κονδύλια λοιπόν προβλέπονται από το Ταμείο, αλλά δεν είμαι βέβαιος αν αυτό είναι ευθύνη των κρατών μελών και δεν θα έπρεπε εκείνοι να επομίζονται αυτή την ευθύνη. Εμείς επομιζόμαστε την ευθύνη για την περιφερειακή ανάπτυξη και για την χρήση των, κονδυλίων του Κοινωνικού Ταμείου να δούμε τι πρέπει να γίνει για να είμαστε αποτελεσματικοί. Παρακαλώ να είσαστε πολύ σύντομος γιατί έχουμε ξεπεράσει το χρόνο μας. Παρακαλώ κύριε, εσείς έχετε τον λόγο. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να κάνω κάποιες πολύ σύντομες ε, παρατηρήσεις. Ο τόνος των συζητήσεων εδώ πέρα κατέδειξε ότι ομόφωνα οι ευρωβουλευτές συμφωνούν για τη σημασία του ταμείου αυτού, μολονότι μπορεί να αποκλίνουν λίγο οι απόψεις μερικές φορές, Ωστόσο όλοι συμφωνούμε ότι θα πρέπει να διατηρηθεί καταρχάς το πρόγραμμα και ότι θα πρέπει να έχει και την απαραίτητη χρηματοδότηση προκειμένου να ανταποκριθεί στις πολύ μεγάλες ανάγκες που έχουν προκύψει. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να επιστρέψουμε λίγο στην πηγή του θέματος. Η δημοσιονομική λιτότητα και όλα τα υπόλοιπα σχετικά θέματα δεν υπάρχουν προφανώς στη συνθήκη της Ρώμης, δεν προβλέπονται από τη συνθήκη της Ρώμης. Αντίθετα όμως η συνθήκη της Ρώμης προβλέπει ότι θα πρέπει οι Ευρωπαίοι πολίτε να έχουν πρόσβαση στο εξή θεμελιώδε δικαίωμα, ισορροπημένη υγιεινή διατροφή. Γι' αυτό το λόγο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να ανταποκριθεί σε αυτή την υποχρέωση, σε αυτή την ευθύνη που έχει να παρέχει το δικαίωμα αυτό στου Ευρωπαίου πολίτε. Επίση, θα ήταν πάρα πολύ σημαντικό οι Ευρωβουλευτέ να τοποθετηθούν για το ζήτημα αυτό πριν την επόμενη Ευρωπαϊκή Σύνοδο, προκειμένου να επενθυμίσουν το ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό η πολιτική συνοχή να έχει ένα πάρα πολύ καλό προπολογισμό που να ανταποκρίνεται πραγματικά στι προκλήσει και να επενθυμίσουν επίση ότι σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θυσιαστεί αυτό το πάρα πολύ σημαντικό πρόγραμμα. Και ουσιαστικά διακυβεύεται εδώ πέρα η πραγματική αξιοπιστία τη Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί ξέρετε, όπω υπόθηκε, ότι υπάρχει ένα τεράστιο χάσμα αυτή τη στιγμή ανάμεσα στου Ευρωπαίου πολίτε και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ πολύ. Τώρα θα αναμένουμε το σχέδιο έκθεσή σα που θα υποβληθεί στι 19 Φεβρουαρίου. Προθεσμία για τι τροπολογίε είναι 21 Φεβρουαρίου. Εδώ τουλάχιστον, αυτό αναφέρεται, 21 Φεβρουαρίου. Θα περιμένουμε πρώτα το σχέδιο έκθεση στι 19 Φεβρουαρίου και θα καθορίσουμε τα επόμενα τότε. Ευχαριστώ, καλό σα απόγευμα, θα τα ξαναπούμε το μεσημέρι, μετά το απόγευμα.